Good morning everybody. Καλημέρα σε όλους και bonjour σε διάφορες γλώσσες. Καλή σας μέρα. Buongiorno. Let's now get started. Please try... Λοιπόν, ας αρχίσουμε. Παρακαλώ προσπαθήστε να βρείτε τη θέση σας το σύντομότερο γιατί έχουμε καθυστερήσει λίγο ήδη. Ώρα Βρυξελών, εντάξει, πάνω κάτω πέντε λεπτά. Θα ήθελα να σας καλωσορίσω στη σημερινή συνεδρίαση που είναι πάρα πολύ μεγάλη. Έχω και μερικές ανακοινώσεις για τις αποφάσεις των συντονιστών. Εγκρίναμε ε, την ημερησία διάταξη για τη 16η Μαΐου και θα προσθέσουμε διάφορα σημεία σε αυτή. Μια αναφορά για τις υδατοκαλλιέργειες, για την έλλειψη ε, ε, αντικειμενικότητα στην Ισπανική τηλεόραση, μια τεχνητή λίμνη στην Ελλάδα, άλλα θέματα στη Λετωνία, ε, μετεκατάσταση του ΕΟΦ, κλιματική αλλαγή και την 0586 για ε, μια μονάδα επεξεργασίας αποβλήτων στη Γαλλικία και ε, τον Ιούνιο τον Ιούνιο, όχι ακόμα, δεν είναι σίγουρο υπό την προϋπόθεση ότι θα έχουμε λάβει απάντηση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή μέχρι τότε. Αλλιώς θα αναβληθεί λίγο. Και μετά την ανακοίνωση του Αντιπρόεδρου Φραν μας ότι δεν θα μπορέσει να είναι στι 16 Μαΐου, αποφασίσαμε να διοργανώσουμε έκτακτη συνεδρίαση στι 3 Τις 3 Μαΐου με τον κύριο Τίμερμανς ε, μόνο ε, ένα σημείο, όχι άλλο θέμα. Για τις εκθέσεις και τις νομοδοτήσεις αποφασίσαμε να κάνουμε δύο νομοδοτήσεις. Ένα για την έκθεση εφαρμογή ε, της Γεωργίας για την προστασία των ζώων κατά τη μεταφορά τους ε, που ε, θα αναλάβει η ΓΚΟΕ την γνωμοδότηση αυτή. Και η δεύτερη γνωμοδότηση είναι στην έκθεση ΑΦΚΟ για την υλοποίηση των διατάξεων της συνθήκης, εφαρμογή που αφορούν την Ευρωπαϊκή Ιθαγένεια και το έχει αναλάβει το ECR. Για τι αντιρρήσει. 11.53 και 12.01 παραμένουν ανοιχτές, 11.64, 11.78 και 11.86 θα κλείσουν. 12.47 θα κηρυχθεί παραδεκτή και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα κληθεί να δώσει συμπληρωματική ενημέρωση. Οι υπόλοιπε αμφισβητούμενες ε, συστάσεις εγκρίθηκαν με τον τρόπο που πρότεινα εγώ. Στα σημεία Β κλείσαμε το 67 το 244, 1360, 463 και την αναφορά 2.45 την κρατάμε ανοιχτή μέχρι να απαντήσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. 2.77 αναφορά 2.11 4.72 θα εγγραφούν στη μερίσια διάταξη επόμενης συνεδρίασης. Πάμε στην διερευνητική αποστολή στην Κύπρο και το πρόγραμμα. Ενέκναν το ενημερωμένο πρόγραμμα οι συντονιστές. Αποφασίσαμε επίσης να ζητήσουμε να συναντηθούμε με την ευτική δύναμη των Ηνωμένων Εθνών στην Κύπρο. Αυτά αποφάσισαν οι συντονιστές για το Jugendamt, το γερμανικό, αποφασίστηκε να ε, αποσταλεί ε, πρόσκληση, επιστολή στην ε, γερμανική κυβέρνηση για να κληθούν οι αρμόδιοι, ο αρμόδιος υπουργό σε επόμενη συνεδρίαση της ομάδας, της Επιτροπής, συγγνώμη. Στη διαδικασία του καταλόγου 3 είχαμε μια πολύ σύντομη ανταλλαγή απόψεων, συνεδρίαση με την ομόλογη επιτροπή μας στη Γερμανική Βουλή, Bundestag, θα έρθουν στις 9 Οκτωβρίου. Θέλουν και εκεί να συναντηθούμε μαζί. Γιατί υπάρχει μια συγκεκριμένη αφορά η 12-12 ε, του 2016 για τα ενότια σήμανση των ε, βοηδών. Αυτά ε, ζητήθηκε και η γνώμη της Επιτροπής Γεωργίας και 0224 για τις εξετάσεις στα σχολεία σε όλες τις επίσημες γλώσσες της αποφύτησης. Θα συνεργαστούμε με την αρμόδια νομοθετική επιτροπή, ε, Επιτροπή Πολιτισμού και θα γίνει προφορική ερώτηση στην Ολομέλεια του Ιουνίου στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να συνάδει με την ε, έκθεση δία πρωτοβουλίας της Επιτροπής Πολιτισμού για τον εξχωρισμό της εκπαίδευση στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Επιπλέον, οι συντονιστέ έλαβαν γνώση στα ενημερωτικά σημεία των θεμάτων και στα διάφορα ενό αιτήματο των πρασίνων. για την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών. περιμένουμε και κάποιους Φιλανδούς ε, αργότερα από τη διεύθυνση του κόμματος των Πρασίνων της Φιλανδίας. Δεν έχουν έρθει ακόμα οι επισκέπτες. Θα τους καλωσορίσω ιδιαίτερα. Αν δείτε 20 άτομα να μπαίνουν στην αίθουσα, θα ξέρετε ποιοι είναι. Είναι οι Φιλανδοί πράσινοι. Ε, προχωρούμε λοιπόν στην ψηφοφορία. Η γνωμοδότηση για την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που τροποποιεί τον κανονισμό 83-2004 ε, για το συντονισμό των συστημάτων κοινωνικής ασφάλειας και ε, ε, τον αντίστοιχο κανονισμό του 2004. Ψηφίζουμε λοιπόν. Έχετε τις κάρτες σας. Δεν νομίζω να τις χρειαστούμε καν. Θα δούμε. Η τροπολογία 66 ψήφι υπέρ παρακαλώ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 67 ήταν ταυτόσημη όπως βλέπετε στο κατάλογο ψηφοφορίας. 68 υπέρ. Κατά. Αποχές. Έλεγχος παρακαλώ. Αρχίζει ψηφοφορία. And the vote is closed τελειώνει. Κοιτάξτε να δείτε τώρα τι έγινε. Ισοψηφία και περίφθη. 69, 70, 71 υπέρ. Κατά. Απόχες εγκρίνονται. Η τροπολογία 72, 73 και 74, όχι, όχι, μία-μία. 72 και 73 μαζί, υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 74 υπέρ κατά αποχές αυτό χρειάζεται έλεγχο και πάλι σας παρακαλώ πέρας απορρίπτεται η τροπολογία 75 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 76 και 77 υπέρ κατά, αποχές, απορρίπτεται. 78 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 14 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 79 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 80 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 81 υπέρ, τσεκ. Ωραία, ελέγχουμε την 80 παρακαλώ, αρχίζει τώρα η ψηφοφορία. Και λίγη μέσος. Απορρίπτεται. 81 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 82 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 83 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 84 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται 85 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 15 υπέρ κατά αποχές εντρύνεται. 86 υπέρ κατά Α, μάλιστα, έχετε δίκιο. 87 υπέρ. Κατά. Άποχες. Απορρίπτεται. 88 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 89 υπέρ, κατά, απόχες, απορρίπτεται. 16 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Η 90 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Τώρα έχουμε τη την 91, 92, 93, σε όλες αυτές και τις ψηφίζουμε μαζί. Υπέρ. Κατά αποχές νομίζω ότι χρειάζεται έλεγχος εδώ. Άρχισε η ψηφοφορία και τώρα μπορεί να κλείσει. Μάλιστα, ό, έχει εγκριθεί. Να σηκώνετε χέρια παρακαλώ. 94 ε, υπέρ, κατά. Αποχές απορρίπτεται. 95 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 97 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται η τροπολογία 100 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 101 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 102 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 103 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 104 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Η 18 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 105 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 19 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 20 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική 4 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Compromise 5 in favor. Συμβιβαστική 5 υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. Συμβιβαστική 7 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 24 και 116 ταυτόσημες υπέρ κατά αποχές δεκτές. 25 και 117 ταυτόσημες υπέρ κατά αποχές δεκτές. 118 και αυτές οι δύο έχουν καταπέσει 18 και 19, πηγαίνουμε στην 120 υπέρ, κατά, αποχές, απερίφθη. 121 υπέρ, κατά, αποχές, απερίφθη. 122 υπέρ, κατά, αποχές, απερίφθη. 123 υπέρ, κατά, αποχές, απερίφθη. 124 υπέρ, κατά αποχές απερίφη 125 υπέρ κατά αποχές απερίφη 26 ε, υπέρ κατά αποχές νομίζω ότι είναι δεκτή 126 υπέρ κατά αποχές δεκτή 27 και 127 υπέρ κατά αποχές δεκτές 128 καταπίπτει. Περνάμε στη συμβιβαστική 8 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 125, 135 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 136 υπέρ κατά αποχές ηλεκτρονικός έλεγχος για την 136 ψηφίζεται. Απερίφθη. Οριακά. 137 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απερίφθη. 29 υπέρ. 29 υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. 30 υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. 31 υπέρ. Κατά. Αποχές. Ηλεκτρονικός έλεγχος γιατί 31 ψηφίζεται. πέραση ψηφοφορίας. Δεκτή. Η 138 καταπληκτή και περνάμε στην 139 υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. 140 υπέρ. Κατά. Αποχές. απερίφη 141 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απερίφη. 142 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απερίφη. 143 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απερίφη. 144 καταπίπτει. 145 υπέρ. Κατά. Αποχές. Ηλεκτρονικός έλεγχος. ψηφίζεται, παρακαλώ για την 145. Δεκτή. 32 υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. 146 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απερίφη. 147 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απερίφη. 33 υπέρ, κατά, αποχές, απερίφθη. 34 υπέρ, κατά, αποχές, απερίφθη. Συμβιβαστική 1, υπέρ, κατά, αποχές, δεκτή. Δεύτερο τμήμα τις 35 που είναι συμβατή με την συμβιβαστική εναρχή είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. Συμβιβαστική 2. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. Τροπολογία 3. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. Αυτή πηγαίνει μαζί με την 37. 39 υπέρ. Κατά. Αποχές. απερίφη 4 υπέρ. Ή μάλλον ηλεκτρονικός έλεγχος για την 39. Ψηφίζετε παρακαλώ. Πέρασε ψηφοφορίες και απερίφη Και βλέπετε με ποιο τρόπο απερίφη Λοιπόν 4 υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. 5 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 41 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 7 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 8 και 43 από κοινού υπέρ κατά αποχές. Ηλεκτρονικός έλεγχος για 8 και 43 ψηφίζεται. Πέρας ψηφοφορίας. Απερίφθη με μία ψήφο διαφορά. 44 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απερίφθη. 45 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απερίφθη. 46 υπέρ. Α, ηλεκτρονικός έλεγχος για τις 45. Θα ελέγχουμε όλες τις τροπολογίες όταν έχουν το όνομα Μαριάς. Λοιπόν, ψηφίζεται Απερίφθη πράγματι με μία ψήφο πάλι διαφορά. Ίσως γιατί κάποιος προσετέθη την τελευταία στιγμή ή κάποιος ε, που ε, τώρα ξεκινάει να ψηφίζει. Λοιπόν 46 υπέρ, κατά, αποχές, απερίφθη. 47 υπέρ, κατά, αποχές. Αυτό θα πρέπει να το ελέγξουμε. Άρχεται η ψηφοφορία για τις λεπτά. Πέρας της απερίφη Με μικρή διαφορά πάντα. Συμβιβαστική 3 υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. Συμβιβαστική 6 υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. 53 υπέρ κατά αποχές απερίφθη 54 υπέρ κατά αποχές απερίφθη 55 υπέρ κατά αποχές απερίφθη Πώς και δεν ζητήσατε έλεγχο εκ νέου. Λοιπόν, 56 υπέρ, κατά, αποχές, απερίφη. 11 υπέρ, κατά, αποχές δεκτή 57 υπέρ κατά αποχές δεκτή 12 υπέρ κατά αποχές δεκτή 58 έχει καταπέσει 60 υπέρ κατά αποχές απερίφη 61 υπέρ κατά αποχές απερίφη 13 υπέρ κατά αποχές δεκτή 62 υπέρ κατά αποχές δεκτή 64 υπέρ κατά αποχές απερίφη 65 υπέρ κατά αποχές απερίφη και τώρα περνάμε στην τελική ψήφο ηλεκτρονική ψηφοφορία άρχεται η ψηφοφορία Πέρας της ψηφοφορίας και υπάρχει απόλυτη αποδοχή με μία αποχή. Αυτά. Α, όχι, έχουμε ένα θέμα ακόμα για να ψηφίσουμε. Για το Ταραντό, τον Τάραντα, εν βάση περιπτώσει, που είχαμε πάει, είχε, ήταν εξαιρετική επίσκεψη, είχαμε μια εξαιρετική ομάδα, περάσαμε πάρα πολύ καλά και αυτά που είδαμε ήταν πολύ ενδιαφέροντα είναι πάρα πολύ σημαντικό για να γνωρίζουμε το τι σημαίνει στην περιοχή αυτή. Περνάμε λοιπόν στην ψηφοφορία τώρα για τον Τάραντα. Τροπολογία 1 υπέρ, κατά, αποχές, δεκτή. 2 υπέρ, κατά, αποχές, απερίφη. 3 υπέρ, κατά, αποχές, υπέρ κατά αποχές δεκτή. Η τέσσερα έχει αποσύρθει, η πέντε υπέρ κατά αποχές. Ηλεκτρονικός έλεγχος για την τροπολογία πέντε ψηφίζεται. Πέρα της ψηφοφορίας δεκτή. έξι υπέρ κατά αποχές απερίφθη. επτά υπέρ κατά αποχές απερίφθη 11 υπέρ κατά αποχές απερίφθη 8 σε διάφορα τμήματα πρώτο τμήμα υπέρ κατά αποχές δεκτό δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές δεκτό τρίτο τμήμα υπέρ κατά αποχές δεκτό Τέταρτο τμήμα υπέρ κατά αποχές δεκτό. Περνάμε στην 9 σε δύο τμήματα. Πρώτο ψηφίζεται. Κατά αποχές απερίφθη. Ηλεκτρονικός έλεγχος λοιπόν για το πρώτο τμήμα της 9. Μεγάλη διαφορά δεκτό δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές απερίφθη. Τροπολογία Α. Ηλεκτρονικός έλεγχος λοιπόν και για το δεύτερο τμήμα. Ψηφίζουμε. Πέρα στις ψηφοφορίες. Δεκτό. Τροπολογία 10 πρώτο τμήμα. Υπέρ. Κατά αποχές δεκτό. Δεύτερο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές δεκτό. Τροπολογία 12 υπέρ, κατά, αποχές δεκτό. Ηλεκτρονικός έλεγχος και για τη 12 ψηφίζεται. Πέραση ψηφοφορίες δεκτή. 13 υπέρ κατά αποχές δεκτή 15 υπέρ Α, συγγνώμη, 14 έχει καταπέσει, οπότε ψηφίζουμε την 15 υπέρ, κατά, αποχές, δεκτή. Ηλεκτρονικός έλεγχος για τη 15. And now It has been rejected. Απερίφθη. Τροπολογία 16 υπέρ. Κατά. Ηλεκτρονικός έλεγχος για την 16. Ψηφίζεται. Απερίφθη. 17 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απερίφθη. Ηλεκτρονικός έλεγχος. Το πρώτο τμήμα της 17 ψηφίζουμε. Κάποιος δεν ψηφίζει. Πέρας της φοφορίας δεκτή. Το δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές δεκτό. 18 υπέρ κατά αποχές απερίφθη. 19 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απερίφη. 21 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απερίφη. 20 υπέρ. Κατά. Αποχές. Ηλεκτρονικός έλεγχος για την 20 ψηφίζεται. Πέρα της ψηφοφορίας δεκτή. Τελική ψήφος, ηλεκτρονική κλίση, ψηφίζεται. Πέρα της ψηφοφορίας. Πράγματι γίνεται δεκτή. Ολοκληρώνουμε, αλλά πριν φύγετε να κάνω μια σημαντική ανακοίνωση, την πιο σημαντική για σήμερα. Ο κύριος Πέτερ Γιάρ έχει γενέθλια. Δεν θα πω ποια είναι η πραγματική του ηλικία. Ο κύριος Γιάρ λοιπόν έχει γενέθλια. Ήταν η πιο σημαντική ανακοίνωση που είχα να κάνω σήμερα. Δεν αποκαλύπτω την ηλικία του. Για μένα πραγματικά θα είναι πάντα forever young ή forever young. Λοιπόν, ε, θα είναι μια μεγάλη μέρα αλλά μια καλή μέρα για όλους, ιδιαίτερα για τον Πέτερ. Καλώς σας ευχαριστώ. Όσοι θέλετε να φύγετε παρακαλώ να το κάνετε γρήγορα. Παρακαλώ όσοι επιθυμούν να εγκαταλείψουν την αίθουσα να το πράξουν τώρα. So πρέπει να προχωρήσουμε. Προφορική ερώτηση λοιπόν και ψήφισμα σχετικά με τις ε, αναφορές οι οποίες αφορούν την καταπολέμηση της επισφαλούς και προσωρινής απασχόλησης στην Ευρώπη. Είμαστε στο θέμα 15 στην ημερήσια διάταξη το κείμενο υπάρχει μόνο στα αγγλικά ε, και ε, στις 26 ε, του μηνός ή στις 3 το μεσημέρι λύγει η προθεσμία για την υποβολή τροπολογιών. Η ψηφοφορία θα γίνει στις, προβλέπεται στις 16 Πέμπτου και η τελική συζήτηση κάποια στιγμή αργότερα, αλλά δεν ξέρουμε ακόμα. Πρώτα απ' όλα θα ήθελα να καλωσορίσω την κυρία Λαγκαρίγκε, και ελπίζω να την πρόφερα σωστά το όνομά της. Ε, ε, έχει το λόγο πάντως. Δίνω το λόγο στην εκπρόσωπο της Κομισιόν. Καλή σας μέρα. Εμείς εξετάσαμε με ιδιαίτερη προσοχή την προφορική ερώτηση και το κείμενο του ψηφίσματος που υπευλήθη από την Επιτροπή σας. step after uh, the very uh, hearing. Επίσης ε, ε, ελάβαμε υπόψη μας ε, το, την πολύ ενδιαφέρουσα ακρόαση του μηνός Νοεμβρίου και την μελέτη που έχει προετοιμάσει η Επιτροπή σας και όλα αυτά αποτέλεσαν πολύ σημαντικά στοιχεία σκέψης για μας σε σχέση με τα όσα υπόθηκαν και το Νοέμβριο. Βεβαίως εμείς συνεχίζουμε τις διαδικασίες επί παραβάση οποτεδήποτε έχουν προκύψει ε, παραβιάσεις της ε, νομοθεσίας. Εν τω όμως πρέπει να πω ότι εγκρίναμε μια πρόταση οδηγίας για ε, ορθές και προβλέψιμες συνθήκες εργασίας και μάλιστα και στην γραπτή δήλωση αναφέρονται όλα αυτά τα στοιχεία και επιπροσθέτως ε, ε, αναφέρεται και ένα ευρύτερο πεδίο εφαρμογής της οδηγίας αυτής καθώς επίσης ε, και κάποια νέα συγκεκριμένα δικαιώματα για τους νέους και όλους όσοι αντιμετωπίζουν ιδιαίτερα προβλήματα σε σχέση με την επισφάλεια και τους επισφαλείς όρους εργασίας. Πραγματικά ε, πιστεύω ότι είμαστε στο σωστό δρόμο και βεβαίως ε, με, υπολογίζουμε και στην ε, δικιά σας υποστήριξη σε αυτήν την καινοτόμα προσπάθεια. Θα συζητηθεί το θέμα στην Ολομέλεια σύντομα οπότε δεν χρειάζεται να πούμε κάτι άλλο, αλλά πραγματικά περιμένουμε την υποστήριξή σας σε σχέση με την πρωτοβουλία μας, έτσι ώστε να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε ε, γενικότερα την επισφάλεια για όλους τους εργαζόμενους στην Ευρώπη. Ευχαριστώ πολύ, λέει η Πρόεδρος. Ευχαριστώ που μας δώσατε πληροφορίες, ενώ, δεν, ε, ενώ ε, είσαστε πολύ σύντομοι. Ευχαριστώ πολύ. το, η προφορική ερώτηση και το ψήφισμα στο προσχέδιό του ε, μας βρίσκουν σύμφωνους με την έννοια ότι αντιμετωπίζουν προβληματισμούς που συχνά μας έχουν απασχολήσει στην Επιτροπή μας ε, και που βεβαίως ε, κορυφώθηκε και με την ακρόαση και τη συζήτηση που είχαμε τον προηγούμενο Νοέμβριο. Η διατύπωση του κειμένου ακριβώς ενδικατοπτρίζει τους προβληματισμούς που προέκυψαν από αυτήν την συζήτηση. Βεβαίως πρέπει να πούμε ότι σε αυτό το στάδιο έχουμε όλο και μεγαλύτερη επισφάλεια ασφάλεια ε, στην ε, Ευρώπη και αυτό βεβαίως ε, δυναμητίζει τις προσπάθειες για κοινωνική ειρήνη και οικονομική σταθερότητα των εργαζομένων επανειλημμένα και μέσω διαφόρων αναφορών από διάφορες χώρες υποβλήθηκε και συζητήθηκε ο προβληματισμός αυτός. Ξέρουμε ότι τώρα υπάρχουν πάρα πολλοί καταχρηστικοί τρόποι με τα συμβόλαια μηδενικής ώρας, με ειδικά συμβόλαια υπερβολικά ευέλικτα αλλά πίσω από αυτά τα συμβόλαια υπάρχουν άνθρωποι υπάρχουν άνθρωποι που θέλουν να ζήσουν και θέλουν βεβαίως να δημιουργήσουν καλύτερη ισορροπία ανάμεσα στη ζωή τους και τη δουλειά τους αλλά βεβαίως θα πρέπει να προσπαθήσουμε έτσι ώστε και οι εργασιακές σχέσεις ανάμεσα σε εργοδότες και εργαζόμενους να είναι ε, καλύτερες. Γι' αυτό λοιπόν καλωσορίζουμε το γεγονός ιδιαίτερος ότι η Επιτροπή ε, αναφορά ε, ακριβώς βασιζόμενοι στα αιτήματα των αναφερομένων ε, φέρνουν το θέμα στην ε, Ολομέλεια. θα πρέπει οπωσδήποτε να κρατήσουμε τον ρόλο μας ε, και να μην οπισθοχωρήσουμε καθόλου και ενώπιον της Ολομελίας ε, τον ρόλο μας λέω ως εκπροσώπων των αναφερομένων. Ε, πιστεύω ότι θα πρέπει να έχουμε μια καλή συζήτηση στην Ολομέλεια όπου θα καταδείξουμε αυτά τα προβλήματα τα οποία αποτελούν καρκίνωμα για την κοινωνία και που πρέπει οπωσδήποτε να ε, τα αντιμετωπίσουμε. Ευχαριστώ. Γερέκ Βαλένσα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Συμφωνούμε με το κείμενο όσο έχει, αλλά χωράει και βελτίωση, πιστεύουμε, σχετικά με την επικεφαλίδα. Νομίζω ότι θα πρέπει να είναι πιο γενικόλογη, αφού μιλούμε για διάφορα είδη απασχόληση, διάφορες μορφές απασχόλησης. Και σε ό,τι αφορά τη συμβάση μηδενικών ορών υπάρχει καλύτερη διατύπωση, ευέλικτες μορφές απασχόλησης. Ε, για το ψήφισμα θα ήθελα να τονίσω ότι για μας η επισφελής εργασία σημαίνει ε, απασχόληση που δεν ανταποκρίνεται σε ευρωπαϊκές ή εθνικές προδιαγραφές και πρότυπα, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά την ασφάλεια ή την υγεία στην εργασία. Η μερική απασχόληση, η προσωρινή απασχόληση, η εποχιακή απασχόληση ε, είναι απαραίτητες μορφές συμβάσεων και χρήσιμες και για τους εργαζομένους και για τους εργοδότες. Για τους λόγους αυτούς ε, οι άτυπες μορφές ε, απασχόλησης όταν συνδυάζονται με το επισφαλής δεν νομίζω ότι είναι σκόπιμο ούτε ακριβές. Σε σχέση με τις προτάσεις της τελευταίας Ευρωπαϊκής Επιτροπής έχω να πω το εξής. Όπως γνωρίζετε η Κομισιόν έκανε μια ανακοίνωση για μια οδηγία για διαφανείς και προβλέψιμες συνθήκες εργασίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση το Δεκέμβριο, σε σύγκριση με άλλες οδηγίες όπως είναι αυτή για τη μερική απασχόληση ή ορισμένου χρόνου ή ε, με απόσπαση εργαζομένων προσωρινή από interim. Αυτό αφορά τις τρέχουσες μελλοντικές ε, συμβάσεις. Πριν από λίγες εβδομάδες η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε ε, προτάσεις για μια ε, Ευρωπαϊκή Αρχή Εργασίας και για την κοινωνική προστασία. Ε, τι στόχο έχουν αυτές οι προτάσεις σύντομα, να προστατεύσουν πολλούς νέους εργαζόμενους, επιπλέον καινούριου δηλαδή, ε, με άτυπες μορφές εργασίας και να βοηθήσουν τα κράτη-μέλη να υποστηρίξουν την πρόσβαση σε αυτές τις μορφές εργασίας για όλους τους εργαζομένους μισθωτούς και αυτοαπασχολούμενους. Θα πρέπει να λάβουμε υπόψη αυτές τις προτάσεις και στα πλαίσια αυτής της προφορική ερώτησης και του ψηφίσματος. Ζητώ συγγνώμη που θα φύγω, πρέπει να πάω να ψηφίσω γρήγορα σε άλλη επιτροπή. Σα ευχαριστώ πολύ για τη συνεισφορά σας και για την ακρίβεια. Καλά, δεν χωράει καμία αμφιβολία πλέον για το που βρίσκεστε σε αυτό το θέμα η ομάδα σας. Θα ήθελα να ζητήσω συγγνώμη που είμαι λίγο αφηρημένη. Είμαι κρυωμένη και ε, το Σαββατοκύριακο πραγματικά με τσάκισε. Ε, από χτες πάω λίγο καλύτερα. Ε, η Ελεονόρα, Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θεωρώ ότι η πρόταση ψηφίσματος και την οποία και η προφορική ερώτηση την οποία εγώ πρότεινα ε, βεβαίως αναφέρεται σε ένα πρόβλημα το οποίο είναι ε, σαφές και μάλιστα έχει πάρει πλέον εκρηκτικές διαστάσεις τα τελευταία χρόνια. Ε, θα πρέπει οπωσδήποτε να το δείξουμε αυτό και να το, πούμε στους διευθύνοντες ε, είναι με γεωμετρική αύξηση ε, η ε, μετριέται η αύξηση του φαινομένου της επισφάλειας και επομένως θα πρέπει και σε εθνικό και σε ευρωπαϊκό επίπεδο να ληφθούν άμεσα μέτρα έτσι ώστε να σταματήσει και να χτυπηθεί στη ρίζα της αυτή η τάση για συμβάσεις μηδενικών ορών υπερβολικά ευέλικτων κλπ. Παραδόξως βεβαίως τώρα τελευταία ε, στον δημόσιο τομέα, στη χώρα μου τουλάχιστον στην Ιταλία, ε, είδαμε πολίτες που έχουν αναγνωριστεί θύματα ε, των ε, παράνομων και καταχρηστικών συμβάσεων να έχουν ε, απολυθεί εν τέλει. Πρόκειται για μια κατάσταση η οποία δεν μπορεί να γίνει πλέον αποδεκτή. Βεβαίως κάποιες ευθύνες φέρει οπωσδήποτε και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διότι έχει ενόχως καθυστερήσει τις διαδικασίες παρά το κατεπήγον της κατάστασης και παρά τις, τα πολλά έγγραφα τα οποία έδειχναν την ανάγκη άμεσης λήψης μέτρων. Ε, μέχρι τώρα πειθαρχικά μέτρα δεν έχουμε δει από την πλευρά της Κομισιόν. Ε, βεβαίως ε, υπάρχουν κάποια στοιχεία εντός του ψηφίσματος ε, τα οποία καταδεικνύουν ακριβώς την ανάγκη αποτελεσματικής αντιμετώπισης και βεβαίως με βρίσκουν σύμφωνοι. Ε, το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο έχει δηλώσει ότι ο, ένα το, μέτρο της ε, τροποποίησης ενός ε, συμβολέου συγκεκριμένου χρόνου σε συμβόλαιο αρίστου χρόνου ε, είναι συμβατό με την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία. και ε, η οδηγία 1979 ε, ακριβώς πρέπει να ολοκληρωθεί και να τροποποιηθεί κατά την έννοια αυτή. Θα πρέπει ε, να πούμε ότι σε ορισμένους τομείς ή για συγκεκριμένες απασχολήσεις και δραστηριότητες μπορούν να υπάρχουν συμβόλαια συγκεκριμένου χρόνου λόγω της φύσης της εργασίας. Επίσης θα ήθελα να πω ότι θα πρέπει να υπάρξουν και κάποιες τροπολογίες, κάποιες τροποποιήσεις ε, κυρίως να υπογραμμίσουμε ότι σε περίπτωση κατάχρησης οποτεδήποτε ε, οι δικαστές αποφασίσουν υπέρ αποζημίωσης των θυμάτων η αποζημίωση δεν θα πρέπει να είναι συμβολικού χαρακτήρα αλλά θα πρέπει πραγματικά ε, να αποκαθιστά την ζημία την οποία έχουν υποστεί οι ενδιαφερόμενοι. Θα ήθελα να ζητήσω και να παρακαλέσω τους συναδέλφους να συμμετάσχουν ενεργά στην διαδικασία αυτής της προφορικής ερώτησης γνωμοδότησης και του ψηφίσματος γιατί είναι πολύ σοβαρό ε, θέμα και πρέπει να εμείς να ε, γίνουμε η φωνή όλων αυτών των ανθρώπων που ζουν ε, στην Ευρώπη με επισφαλείς όρους εργασίας. Ευχαριστώ πολύ. Thank you, Mr. Maria. Ευχαριστώ κύριος Μαριάς παρακαλώ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Θεωρώ σημαντική την πρωτοβουλία για την προφορική ερώτηση, τη συζήτηση και το ψήφισμα για τις ευέλικτες ε, μορφές απασχόλησης. Είναι ένα τεράστιο πρόβλημα το οποίο απασχολεί πλέον ολόκληρη την Ευρώπη. Αλλά βεβαίως ξεκινά από την αντίληψη πριν από ορισμένα χρόνια ότι θα πρέπει στο όνομα της δίθεν ανταγωνιστικότητας της ευρωπαϊκής οικονομίας να μειωθούν οι μισθοί. Διότι από εκεί ξεκινάει όλη η διαδικασία. Θεώρησαν ορισμένοι κύκλοι στην Ευρώπη ότι μπορεί να είναι ανταγωνιστική η ευρωπαϊκή οικονομία εάν οδηγήσουν σε μια κινεζοποίηση των μισθών. Ενώ απεδείχθη μετά από χρόνια ότι η ανταγωνιστικότητα στην οικονομία κατά κύριο λόγο στηρίζεται στις καινοτομίες, στις νέες τεχνολογίες, στα χαμηλά επιτόκια δανεισμού και στο χαμηλό κόστος ενέργειας. Επομένως, μετά από αρκετά χρόνια και παρότι και εγώ και πολλοί άλλοι, εγώ και σαν καθηγητή στο Πανεπιστήμιο τη Κρήτη, που ασχολούμαι με τα θέματα αυτά, αλλά και σαν δικηγόρο, είχα επισημάνει ότι δεν πρόκειται να ενισχυθεί η ανταγωνιστικότητα τη Ευρωπαϊκή Οικονομία, διαλύοντα του μισθού και το κράτο πρόνοιας. Δυστυχώ, όμω, οδηγηθήκαμε σε αυτή την κατάσταση. Πλέον αυξάνονται οι άτυπε μορφές απασχόληση, Φτάσαμε στο άλλο άκρο, δηλαδή να έχουμε συμβόλαια μηδενικών ορών, να έχουμε πλέον μια αυθαιρεσία των επιχειρήσεων, να μην υπάρχει ασφάλεια και στους ίδιους τους εργαζομένους και ταυτόχρονα με αυτές τις μορφές απασχόλησης να έχουμε και χτύπημα και της κοινωνικής ασφάλισης. Διότι όταν έχεις μειωμένο αριθμό ωρών απασχόλησης και όταν οι εργοδότες ασφαλίζουν για πολύ μικρό αριθμό ωρών εργασίας στους ίδιους εργαζομένους, αυτό σημαίνει ελαχιστοποίηση των ε, εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, άρα διάλυση του κοινωνικού ασφαλιστικού συστήματος, άρα πέρασμα σε μέτρων μείωσης των συντάξεων, διότι αυτή είναι η πραγματικότητα. Χαίρομαι λοιπόν που θα συζητήσουμε αυτό το ζήτημα, αλλά τα συμπεράσματά μας πρέπει να είναι αποφασιστικά. Ότι πρέπει να περάσουμε σε τέτοιες μορφές απασχόλησης οι οποίες να στηρίζουν την ίδια την απασχόληση και ταυτόχρονα να αντιληφθούμε ότι η υποτιθέμενη ευελιξία και μάλιστα η ασφάλεια στο πλαίσιο της ευελιξίας, αυτό που κάποιοι ονόμασαν flexicurity, δεν απέδωσε, δεν βοήθησε και διάλυσε την αγορά εργασίας. Κάποιοι πρέπει να κάνουν την αυτοκριτική τους, διότι επέμεναν πριν από 15-20 χρόνια και επέβαλαν αυτές τις μορφές απασχόλησης και στον ιδιωτικό τομέα, αλλά και στο δημόσιο τομέα. Θα έλεγα λοιπόν ότι θα πρέπει να δούμε και κοινωνικά μέτρα στήριξη της απασχόλησης, θα πρέπει να υπάρξει η σκέψη και για ένα ελάχιστο ευρωπαϊκό μισθό και ταυτόχρονα η σκέψη για ε, ένα ενιαίο ελάχιστο επίδομα ανεργίας στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επομένως νομίζω ότι κατά τη συζήτηση οι διάφορες πολιτικές ομάδες, οι συνάδελφοι θα εκφράσουν τις απόψεις τους, αλλά καλό είναι να χτυπηθεί η αντίληψη που θεωρεί ότι η δίθεν ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής οικονομίας στηρίζεται στη διάλυση των εργασιακών σχέσεων και στην ελαχιστοποίηση των μισθών παρότι ακόμη και η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα θέλει να πετύχει την αύξηση του πληθωρισμού, βλέπουμε ότι δεν επέρχεται αύξηση των μισθών. Και δεν επέρχεται αύξηση των μισθών ακριβώς διότι είναι διαλυμένες οι εργασιακές σχέσεις. Ακριβώς γι' αυτό το λόγο δεν επέρχεται η αύξηση των μισθών, άρα και η άνοδος του πληθωρισμού κοντά στο 2% το οποίο υποτίθεται θέλει και η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Νομίζω με αυτές τις σκέψεις εμείς ε, ως ECR θα παρουσιάσουμε τις απόψεις μας και κατά τη συζήτηση και βεβαίως στην πορεία ε, όλης αυτής της ε, διαδικασίας. Ευχαριστώ. Thank you very much. παρακαλώ. σας. Ε, νομίζω πως οι συνάδελφοι έχουν ήδη καλύψει τολμώ να πω το σύνολο και των δικών μας απόψεων. Έχει γίνει μια πάρα πολύ καλή δουλειά και συγχαρητήρια σε όσους εργάστηκα. Η, η ερώτηση ε, καλώς ε, ήλθε ενώπιόν μας και εξετάζεται. Νομίζω ότι έχουμε ένα πρόβλημα σε όλες τις κοινωνίες της Ευρώπης που αφορά τη δύναμη των εργοδοτών. Είτε αυτοί είναι ιδιώτες είτε είναι το κράτος είναι η δύναμη των εργοδοτών γιατί πάντα το χρήμα επηρεάζει είτε μέσα ενημέρωσης είτε και ε, περιοχές ανθρώπων που παίρνουν τις αποφάσεις. Το ζητούμενο τώρα είναι, επειδή και παλαιότερα το Ευρωκοινοβούλιο ασχολήθηκε με αυτό το ζήτημα και στην Ολομέλεια και έχουν γίνει και άλλες εκθέσεις, <clears throat> αυτό που κάνουμε τώρα έρχεται ως ενισχυτικό αυτών των προσπαθειών. Το ζήτημα που μπαίνει είναι τι αναμένουμε τι συγκεκριμένο αναμένουμε από την Κομισιόν να φέρει ενώπιον μας ως ε, τροποποιητικές νομοθεσίες. Αυτό είναι το ένα. Και το δεύτερο είναι τι πίεση ασκούμε εμείς στα κράτη-μέλη μέσα από τα μέσα επικοινωνίας που έχουμε στη διάθεσή μας αλλά και πίεση πάνω στα αρμόδια Υπουργεία έτσι ώστε να εφαρμοστούν οι οποιασδήποτε αποφάσεις σωστές παίρνει ε, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ε, γιατί δεν βλέπω ότι είναι εύκολο δυστυχώς να αλλάξει όσο το δυνατόν πιο σύντομα γιατί αυτό είναι που πρέπει αυτή η κατάσταση δεδομένης δε και της κρίσης της οικονομικής που χτύπησε αν όχι όλα τα κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης μερικά από αυτά πάρα πολύ σκληρά η εργοδοσία αξιοποιεί ή χρησιμοποιεί και την οικονομική κρίση ε, προκειμένου να επιβάλλει ε, αυτούς τους ε, όρους εργασίας πιο εσχρό τρόπο το λεγόμενο συμβόλαιο μηδενικών ωρών, Αλλά υπάρχει και από την ανάποδη πρόβλημα. Στην Κύπρο ξέρω κόσμο που εργάζεται πολύ πέραν του 8ωρου ή και του 10ωρου. Τα Σαββατοκυριακά ουσιαστικά δεν υπάρχουν, παίρνουν κάποιες μέρες μέσα στη βδομάδα. Ε, και άκουσα μια έκφραση η οποία είναι συγκλονιστική και καθορίζει την δυσκολία των εργασιών αυτών. Κάνουν συμβόλαια επιτραπέζιων χεριών, λέει. Επιτραπέζια χέρια τι σημαίνει. Είναι ένας άνθρωπος που κάθεται σε ένα ταμείο και όλη μέρα κινούνται τα χέρια του. Δεν, δεν, δεν, δεν κάνει κάτι άλλο. Επί δέκα ώρες να χτυπάει συνεχώς ε, στη μηχανή. Δεν ξέρω πώς δεν τρελαίνεται ένας τέτοιος άνθρωπος. Και ονόμασαν, τόλμησαν μάλιστα να ονομάσουν αυτή τη δουλειά συμβόλαιο επιτραπέζιων χεριών. Ε, σημαίνει ότι η, η εκτίμηση, η λέξη δεν είναι σωστή, η αντίληψη που έχουν για τους εργαζόμενους είναι ε, επίπεδου κάτω από, κάτω από το ζήρο. Εμείς και όλοι μας εδώ πιστεύω ότι στη συνέχεια στα κράτη-μέλη θα προσπαθήσουμε να περάσουμε το μήνυμα ότι υπάρχει ισχυρή βούληση του Κοινοβουλίου αυτά τα πράγματα να αλλάξουν. Ευχαριστώ. εγώ σας ευχαριστώ. Δεν έχει δει κανεί άλλο το λόγο στον κατάλογο των ομιλητών. Όπω σα είπα, η ψηφοφορία θα γίνει στις 16 Μαΐου. Στο μεταξύ θα ε, φροντίσουμε να διοργανώσουμε μια συνεδρίαση όπου θα συναντήσουμε τις διάφορες ομάδες. Στις 2 Μαΐου, στις 2 Μαΐου έχει ήδη προβλεφθεί και προγραμματιστεί η συνεδρίαση αυτή και περιμένω να γίνει. Και την άλλη φορά στην Επιτροπή μας ελπίζω να εγκρίνουμε το κείμενο και να προχωρήσουμε. Σας ευχαριστώ πολύ για τη συμμετοχή σας στη συζήτηση αυτή και για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Και θα προσπαθήσουμε να προτείνουμε και να ε, προωθήσουμε πολύ διαρθρωμένες συγκροτημένες ερωτήσεις για να βοηθήσουμε. Και εσείς και εμείς ε, εργαζόμαστε βάσει των αναφορών που λαμβάνουμε και είναι πολύ καλή αυτή η διοργανική συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Πηγαίνουμε τώρα στο επόμενο θέμα, αναπηρία 16, ε, αναφορά 535 σχετικά με τις μετακινήσεις των ατόμων με αναπηρία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ε, απουσιάζει ο αναφέρον, αλλά θα παρακολουθεί ε, πιθανότατα από το διαδίκτυο της συνεδρίασή μας. Αν μας ακούτε, σας καλωσορίζουμε στην Επιτροπή μας και ελπίζω να σας δούμε και προσωπικώς κάποια άλλη φορά. Ε, παρίσταται όμως όπως πάντα Ευρωπαϊκή Επιτροπή και με χαρά θα της δώσω το λόγο. Σας ευχαριστώ Πρόεδρε. Σοφή Μαγακομπό λέγομαι και εργάζομαι στη Γενική Διεύθυνση ΜΟΒ για τα δικαιώματα των ε, ε, επιτροπών και θα συνεχίσω στα γαλλικά που είναι και η μετρική μου γλώσσα. Λοιπόν, για να συμπληρώσω τις πληροφορίες που έχετε λάβει, ε, θα επιθυμούσα να σας δώσω λίγο το πλαίσιο ε, των κανόνων που ισχύουν για τα δικαιώματα των επιβατών ε, σε ό,τι αφορά τα άτομα με αναπηρίες ή με περιορισμένη κινητικότητα. Αυτά τα στοιχεία και διατάξεις εντάσσονται στο ευρωπαϊκό δίκαιο και στα δικαιώματα των πολιτών. Θα ήθελα λίγο να επανέλθω στον τρόπο με τον οποίο παρέχεται η βοήθεια στα άτομα με αναπηρίες ή με περιορισμένη κινητικότητα. Τι προβλέπουν οι κανονισμοί λοιπόν θα πρέπει να υπάρχει μία ε, ειδοποίηση εκ των προτέρων. Αν χρειάζεσαι βοήθεια, θα πρέπει να το δηλώνεις. Υπάρχει μια προθεσμία την οποία αμφισβητεί ο αναφέρον και θα σας εξηγήσω για ποιο λόγο ε, γίνεται λόγος για 36 ώρες ή 48 ώρες ανάλογα με το μέσο μεταφοράς. Γιατί έχει ενταχθεί η ε, πρόνοια στον κανονισμό. Για δύο βασικούς λόγους. Πρώτον, θα πρέπει να βεβαιωθούμε ότι και το προσωπικό που χρειάζεται για να βοηθήσει τους ανθρώπους με μειωμένη ε, κινητικότητα αλλά και το υλικό που χρειάζεται ο εξοπλισμός θα πρέπει να είναι στη διάθεσή του τη στιγμή της ε, ε, αναχώρησης του ακόμα και όταν είναι σε περίοδο εχμής για το συγκεκριμένο μέσο μεταφοράς. Εξού και ο κανονισμός λέει ότι θα πρέπει να είναι μια βοήθεια προσαρμοσμένη και κατάλληλη για το πρόβλημα που αντιμετωπίζει ο εκάστοτε επιβάτης. Δεν ξέρω αν το έχετε ζήσει εσείς. Να σας δώσω ένα παράδειγμα ή αν έχετε λάβει αυτή τη βοήθεια. Παράδειγμα, αν είναι κάποιος σε ε, ε, ε, μια αναπηρική καρέκλα και θέλει να ταξιδεύσει με αεροπλάνο, χρειάζεται δύο υπαλλήλου στο αεροδρόμιο, ανελκυστήρα για να φτάσει η πολυθρόνα στο αεροπλάνο. Μπορεί να χρειαστεί να αλλάξει και πολυθρόνα για να χωράει στο αεροπλάνο Όλα αυτά θα πρέπει να γίνουν χωρίς να καθυστερήσει η αναχώρηση της πτήσης. Καταλαβαίνετε ότι με το ίδιο αεροπλάνο κάποιοι επιβάτες φτάνουν και θα πρέπει να βγουν πριν μπουν οι νέοι επιβάτες για την καινούρια πτήση. Άρα... Όλα αυτά χρειάζονται μια ελάχιστη ε, οργάνωση εκ των προτέρων και ένα συντονισμό για να μπορούν τα αεροδρόμια να ε, κανονίσουν την πορεία τους. Και επίσης όλες αυτές οι διατάξεις είχαν στόχο να επιτρέψουν στους επιβάτες αυτούς να ταξιδεύουν μόνοι τους. Να μην χρειάζονται οπωσδήποτε να έχουν ένα συνοδό ή κάποιον για να τους βοηθάει και να είναι αυτόνομοι στις μετακινήσεις τους. Για αυτούς τους δύο λόγους λοιπόν ε, ορίστηκαν αυτές οι προθεσμίες. Μας φαίνονται λογικές. Και γι' αυτό εντάχθηκαν στην νομοθεσία. Ευχαριστώ και αφήνω το λόγο στη συνάδελφό μου από τη Γενική Διεύθυνση Απασχόλησης. Σας ευχαριστώ. Χάνα Βαλέτσκα λέγομαι από τη Γενική Διεύθυνση Employment, ε, απασχόληση. Εμείς ε, συνεισφέραμε με πληροφορίες ε, για το πιλωτικό μας πρόγραμμα. Τώρα εφαρμόζουμε ένα πιλωτικό πρόγραμμα που κανονικά στόχο έχει να βοηθήσει την ελεύθερη κυκλοφορία και την ε, ε, εθελούσια αναγνώριση του καθεστώτος αναπηρίας. Μέχρι στιγμής αυτό εφαρμόζεται μόνο σε 8 χώρες. Αλλά φέτος θέλουμε να κάνουμε πρώτα την αξιολόγηση και να το επεκτείνουμε. Ελπίζουμε να μπορέσουμε να το προσφέρουμε και σε άλλες χώρες αυτό το μοντέλο. Και το σχέδιο του πιλωτικού βασίζεται σε θελούσια αμοιβαία αναγνώριση. Ε, τώρα αφορά τον πολιτισμό, τον αθλητισμό, την ψυχαγωγία και τις μεταφορές φυσικά. Αυτή είναι οι τομείς που καλύπτονται, αλλά και ε, ε, οι μεταφορές είναι σημαντικός τομέας αλλά και πολύ δαπανηρός. Οπότε όλες οι χώρες δεν εμφανίζουν προθυμία να εντάξουν και το θέμα των μεταφορών σε αυτό το πιλωτικό πρόγραμμα. Ελπίζουμε στο μέλλον να συμμετέχουν και περισσότερες χώρες αλλά και ο τομέας των μεταφορών. Ένα άλλο θέμα για το οποίο ρώτησε ο αναφέρον είναι τι γίνεται με την παροχή βοήθειας ε, προσωπικής. Τα συστήματα που αναπτύσσονται και πάλι βασίζονται στην ε, εθελοντική αμοιβαία αναγνώριση. Δηλαδή κάθε χώρα θα αποφασίσει αν θα εντάξει στο σύστημα αυτό την βοήθεια προς τους επιβάτες. Πώς έχει σήμερα η κατάσταση. Τα πιλωτικά προγράμματα έχουν ολοκληρωθεί και τώρα είμαστε στο στάδιο της ε, Αξιολόγηση και ελπίζουμε του χρόνου να ε, μπορέσουμε να διαπραγματευτούμε και με άλλε χώρε για να ενταχθούν σε αυτό το πιλωτικό πρόγραμμα και στη συγκεκριμένη δράση. Σας ευχαριστώ. Thank also Σας ευχαριστώ πολύ. ήταν και σαφέστατοι. Ε, τώρα ε, είναι εθελοντικές οι συμφωνίες αυτές και ξέρουμε πολύ καλά τι σημαίνει και τι αποτέλεσμα έχουν. Είμαστε πολύ παλιές καραβάνες εδώ για να έχουμε πολύ μεγάλες ελπίδες. Λοιπόν, το λόγο έχουν οι συνάδελφοι και καλωσορίζω και τη Σολεδάδ Καπεθών ε, Ρουίτ στην Επιτροπή μας. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Ευχαριστώ και τον αναφέροντα που έφερε και πάλι αυτό το θέμα το οποίο έχει απασχολήσει επανειλημμένα την Επιτροπή μας, που είναι η πρόσβαση των ατόμων με αναπηρίες στις μεταφορές. Και το λέω ότι ε, το έχουμε ξαναδεί και επανειλημμένα το έχουμε συζητήσει και θέλω να το επαναλάβω. Ξέρω ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει ένα πιλωτικό πρόγραμμα και το καταλαβαίνω, αλλά θέλω να πω ευθύ εξ αρχή ότι ε, αμφισβητώ τη βιωσιμότητα του προγράμματος αν ε, προτείνεται αυτό να είναι σε εθελοντική βάση. Εξαρτάται από την βούληση και την προθυμία των κρατών μελών. Αν θα κάνουν συστάσεις και υποχρεώσεις σε κάποιες εταιρείε. Αφήστε που είναι και εθνικέ αρμοδιότητε και όχι ευρωπαϊκέ πολλέ φορέ αυτά τα πράγματα. Νομίζω ότι χρειάζεται μεγαλύτερη φιλοδοξία. Μεγαλύτερη φιλοδοξία. Γιατί από την Ευρωπαϊκή Ένωση χρειάζεται να υπάρχει μια πολιτική για τα άτομα με αναπηρίες. Όχι απλώ να τα λαμβάνουμε σοβαρά υπόψη και να κάνουμε συζητήσει. Συγκεκριμένα μέτρα χρειάζονται. Θα σας έλεγα λοιπόν ότι εδώ ακριβώς ήρθε αυτό το θέμα με συγκεκριμένα προβλήματα σε εταιρείε ε, χαμηλού κόστους αεροπορικές, low cost. Υπάρχουν συγκεκριμένες αναφορές και ειδικέ περιπτώσεις για το πώς συμπεριφέρονται σε αυτούς τους ανθρώπους οι εταιρείε low cost. Και δεν μπορούμε να είμαστε ούτε συγκαταβατικοί ούτε να περιμένουμε ε, τι θα κάνουν τα κράτη-μέλη. Πολλέ φορές τους υποχρεώνουν να έχουν συνοδό, δηλαδή να αγοράσουν δύο εισιτήρια. Μα τι είναι αυτά, διακρίσεις κατάφορες. Θα πρέπει να ληφθούν κάποια μέτρα έτσι ώστε εάν υποχρεούνται να έχουν συνοδό να είναι δωρεάν το δεύτερο εισιτήριο. Ξέρετε ότι εδώ έχουμε ψηφίσει μια γνωμοδότηση σήμερα μόλις για το συντονισμό των συστημάτων κοινωνικής ασφάλειας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Στην Επιτροπή μας μας ενδιαφέρει πολύ αυτό το θέμα των ατόμων με αναπηρίες. Και θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση να έχει ενιαίο ορισμό για τις αναπηρίες και εναρμονισμένα κριτήρια. Το ζητάει και ο αναφέρον αυτό. Δεν σας μιλώ για παροχές, γιατί εκεί μπορεί να υπάρχουν προβλήματα με το Συμβούλιο. Αλλά μόνο αν έχεις κάρτα αναπήρου ευρωπαϊκή θα λυθεί το πρόβλημα και δεν θα υπάρχουν ε, διακρίσεις. Αν είναι αναγνωρισμένα όλα τα άτομα με αναπηρίες, να έχουν κάρτα αναπηρίας και να ισχύει αυτή σε όλες τις χώρες, σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Υπάρχουν κάποιες χώρες που χαρακτηρίζουν μια κατάσταση αναπηρία και κάποιες άλλες όχι. Δηλαδή τι θα κάνεις, έχεις ισπανική κάρτα αναπήρου, πας στην Κροατία και σου λένε δεν είσαι ανάπηρος. Δεν έχεις δικαιώματα και δεν στα αναγνωρίζουν για κάποιες παροχές. Δηλαδή ο ίδιος άνθρωπος που έχει την ίδια αναπηρία θεωρείται στην Ισπανία άτομο με αναπηρία και στην Κροατία όχι. Και δεν μπορεί να διεκδικήσει τα δικαιώματά του. Αυτά. Πολύ απλά να υπάρχει μια ευρωπαϊκή κάρτα αναπηρίας που θα βοηθήσει πάρα πολύ. και δεν θα υπάρχουν διακρίσεις και θα εναρμονιστούν έτσι τα κριτήρια στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Όλα αυτά είναι πάρα πολύ απαραίτητα και επίγοντα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Μαριάς. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θεωρώ πάρα πολύ σημαντική την ε, αναφορά και βεβαίως παρότι ο αναφέρον δεν είναι παρόν και προφανώς θα έχει ίσως πρόβλημα μετακίνησης. Νομίζω ότι τα όσα τέθηκαν και από την Κομισιόν αλλά και από την ε, συνάδελφο ε, στην παρέμβασή της είναι ιδιαίτερα σημαντικά. Ήδη έχουμε συζητήσει πάρα πολλές φορές το θέμα της πρόσβασης των ατόμων με αναπηρία ε, και της δυνατότητάς τους να μετακινηθούν στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θυμόσαστε ε, την συζήτηση που κάναμε με αφορά το, με σε σχέση με το πρόβλημα που υπάρχει στη Ρουμανία, όπου δεν μπορούν πρακτικά τα άτομα με αναπηρία να αξιοποιήσουν τους σιδηροδρόμους όπου επί της ουσίας πρέπει να ειδοποιούν αρκετές ημέρες πιο πριν ότι πρόκειται να ταξιδέψουν για να έχουν κάποιες παροχές. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι αυτό δεν μπορεί να συνεχίζεται και θα πρέπει ιδίω σε υποδομές οι οποίες χρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και είναι πάρα πολλές αυτές οι υποδομές όπως είναι βεβαίως και η λειτουργία των σιδηροδρόμων αλλά και των αεροδρομίων θα πρέπει να υπάρχει η δυνατότητα της πλήρους πρόσβασης των ατόμων με αναπηρία. Το δεύτερο θέμα βεβαίως αφορά τους συνοδούς ότι θα πρέπει να υπάρξει μια πρόβλεψη είτε για την δυνατότητα Παροχή ενός δωρεάν εισιτηρίου για τους συνοδούς είτε ενός ε, εισιτηρίου με πάρα πολύ μεγάλη έκπτωση προκειμένου να μπορούν να συνοδεύσουν τα άτομα με αναπηρία. Ε, το τρίτο θέμα έχει σχέση με την αναγνώριση της αναπηρίας. Ε, επειδή θεωρώ πολύ σωστή την παρατήρηση ότι πρέπει να θεσμοθετηθεί η Ευρωπαϊκή Κάρτα Αναπηρίας, το ζήτημα είναι ότι μέχρι να θεσμοθετηθεί αυτή η κάρτα τι κάνουμε. Πιστεύω λοιπόν ότι σε πρώτη φάση θα μπορούσε να υπάρξει μια αμοιβαία αναγνώριση τη κάρτα αναπηρία που υπάρχει σε κάθε κράτο μέλο. Δηλαδή να υποχρεούται κάθε κράτο μέλο να αναγνωρίζει την κάρτα αναπηρία που εκδίδουν τα υπόλοιπα κράτη-μέλη. Αυτό θα διευκολύνει τους αναπήρους να κινηθούν και δεύτερον θα ασκήσει μια πίεση σε όλα τα κράτη-μέλη επιτέλους να θεσμοθετήσουν την Ευρωπαϊκή Κάρτα Αναπηρίας και έτσι να ενοποιήσουν σε μεγάλο βαθμό τα κριτήρια. Θα έλεγα λοιπόν ότι και αυτή η αναφορά για άλλη μια φορά αναδεικνύει τα προβλήματα που έχουν τα άτομα με αναπηρία σε σχέση με την πρόσβασή τους και την δυνατότητα να κυκλοφορούν ελεύθερα στην Ευρωπαϊκή Ένωση ε, είτε με αεροπλάνο είτε με άλλα μέσα μαζικής μεταφοράς. Ευχαριστώ. Ε, Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ε, η εμπειρία μου είναι τεράστια και οι πίκρες ε, επίσης τέρα, πάρα πολλές γιατί συνέχεια μετακινούμε και με αεροπλάνα και με τρένα και με διάφορα μέσα μαζικής μεταφοράς σε όλη την Ευρώπη και το ξεκινάω πρώτα με τις Βρυξέλλες γιατί είναι ίσως η πιο άσχημη κατάσταση σε όλη την Ευρώπη, σε όλες τις ε, πρωτεύουσες της Ευρώπης. Είναι απαράδεκτο που οι Βρυξέλλες στεγάζει 90% από τις ευρωπαϊκές οργανώσεις και δεν έχει προσβασιμότητα. Όχι μόνο σαν δομή η πόλη, αλλά είναι πολύ κακές εξυπηρετήσεις και στα τρένα και, στο αεροδρόμιο. Δεν είναι καλά οργανωμένοι, δεν έχουν τη λογική που χρειάζεται να έχουν αυτές οι υπηρεσίες. Στη Γαλλία, αν δεν έχεις δηλώσει 48 ώρες νωρίτερα στα τρένα, ότι θα με τρένο, δεν σου δίνουν βοήθεια ή τουλάχιστον σε δυσκολεύουν πάρα πολύ μέχρι να σου δώσουν. Δηλαδή δεν έχω δικαιώμα να αποφασίζω σήμερα ότι ταξιδεύω. Γιατί υπάρχει αυτή η διάκριση με του ανθρώπου με αναπηρία και του περιορίζουν και έχουν μεγάλε ελευθερίε οι εταιρείε και το νομικό πρόσωπο του εμπορίου και εμεί δεν έχουμε αυτή την ελευθερία σήμερα να αποφασίζω ότι ταξιδεύω και να μου δώσουν βοήθεια. Μετά, ε, η κάρτα αναπηρίας είναι αναγκαία, αναγκαία επίγον, γιατί τα άτομα με αναπηρία έχουν θα πρέπει να έχουν ίσα δικαιώματα και τις δυνατότητες να μετακινούνται στην Ευρώπη και να έχουν τις, τα, τα ωφέλη όλων των χωρών της Ευρώπης. Δεν είναι τόσο δύσκολο. Έχουμε το ε1, έχουμε τα ε2, έχουμε τόσο πολλά έγγραφα τα οποία βοηθάνε σε θεραπεία σε διάφορες περιπτώσεις ατόμων με αναπηρία και δεν έχουμε την κάρτα αναπηρίας που μπορεί να μας δώσει τα αυτονόητα, να μετακινηθούμε με ίσια δικαιώματα. Ε, προτείνω να καλέσουμε το Δήμο Βρυξελών εδώ στην Επιτροπή να συζητήσουμε μαζί τους και να τους βάζουμε κάποιες προτάσεις που έχουμε και παρατηρήσεις έτσι ώστε τουλάχιστον στο μέλλον να οργανωθεί αυτή η πόλη και να, να είναι προσβάσιμη και από τους ανάπηρους και από τους ανθρώπους που έχουν προβλήματα. Είναι πολλά που μπορώ να συζητήσω Είναι απαράδεκτο όταν μπαίνω στο αεροπλάνο με παιδιά που έχουν μεγάλη αναπηρία στην κινητικότητα. Τους τραβάνε από το καρότσι, τους τραβάνε να τους βάζουν στο παράτερο στη τρίτη καρέκλα με τη σειρά. Μετά το στραβάνι, από εκεί να του βάζουν ξανά στην καρέκλα. Μετά στη δικά του καρέκλα του στραβάνι. Δεν είναι ανθρώπινη συνθήκη αυτή ε, ένα επιβάτη με τόσο μεγάλη αναπηρία και κινδυνότητα στη ζωή. Αυτό δεν είναι ασφάλεια. Δεν είναι κατάλληλη βοήθεια που χρειάζεται ένα ανάπηρο. Είναι τόσο δύσκολο να λείπουν ή να σηκώνονται κάποιε θέσει στο αεροπλάνο και να μπει το δικό του καρότσι, να μην το τραβάμε σαν ένα τσουβάλι. Και μετά αυτό να πονάει τρει μέρε και να προετοιμάσετε ψυχολογικά μήνες ότι θα ταξιδέψει. Ευχαριστώ. Και εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Δυσκολεύεται πολύ. Και ραγίζει η καρδιά μου όταν ακούω πώς είναι η κατάσταση εδώ. Απαράδεικτο είναι. Απαράδεικτο. Τέλειο. Σας ευχαριστώ πάλι πάρα πολύ. Ρώσα. Ρώσα Ευχαριστώ πολύ. Συμφωνώ πολύ τους. Είχαμε πολλές αναφορές για το θέμα αυτό και το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα ζήτησε να γίνει αποστολή στη Ρουμανία. Γιατί ξέρει πρόεδρος και εγώ ότι υπάρχει μεγάλη δυσκολία στις μεταφορές. Πολλές φορές δεν είναι υποχρεωτικό να γίνονται αυτές οι προσαρμογές. Και ακούσαμε ότι στη Ρουμανία υπάρχει πρόβλημα. Τώρα υπάρχει αυτό το πιλωτικό πρόγραμμα της ε, Ευρωπαϊκής Ένωσης σε κάποιες χώρες. Βέλγιο, Κύπρος, Εστονία, Φιλανδία, Ιταλία, Μάλτα, Σλοβανία και Ρουμανία συμμετέχουν για να ανταλλάξουν βέλτιστες πρακτικές έτσι ώστε να υπάρξει και μια κοινή κάρτα στάθμευσης Αυτέ οι 8 χώρε συμμετέχουν μόνο. Και τώρα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή καλείται να αξιολογήσει με αυτό το πρόγραμμα, το πιλωτικό, τι μπορεί να βελτιωθεί και τι θα προτείνει στο μέλλον. Εγώ συμφωνώ και με την κυρία Κούνεβα και με το συνάδελφο μου, τον κύριο Μαριά που μίλησε και με τη Σολεδάθ. Κάναμε την ελεύθερη κυκλοφορία των εμπορευμάτων, των προσώπων, την ψηφιακή, καταργήσαμε την περιαγωγή. Αλλά στα άτομα με αναπηρίες δεν ισχύουν αυτές οι ελευθερίες και δεν υλοποιούνται. Δεν μπορούν να ταξιδέψουν οι άνθρωποι Πρέπει να προειδοποιούν πολύ νωρίς Δεν είναι ανεπτυγμένε όλε οι χώρες στις μεταφορές υπάρχουν πολλά εμπόδια. Για το εράσμους ας πούμε, υπήρξε ένα εράσμους για άτομα με αναπηρίε και πήραν πέντε μόνο. Γιατί δεν προέβλεπαν κάποιον με βαριά αναπηρία να έχει συνοδό. Και δεν προέβλεπαν λοιπόν ότι δεν υπάρχει συνοδό, άρα δεν του δίνανε εράσμους Και για να το πετύχουμε χρειάστηκαν δύο χρόνια. Έχουμε βελτιώσει πολλά πράγματα, έχουμε διορθώσει για άλλα και νομίζω ότι η Επιτροπή μας εδώ αναφορών μπορεί να κάνει πολλά ακριβώς για να υπάρξει αμοιβαία αναγνώριση ε, Τη ε, της αναπηρίας, του βαθμού αναπηρίας. Δηλαδή κάθε επιτροπή σε κάθε χώρα αποφασίζει τι ποσοστό αναπηρίας έχεις. Αυτό δεν μπορεί να ενοποιηθεί στην Ευρώπη σε μία ενιαία κάρτα και να αναγνωρίζουν όλοι τον ίδιο βαθμό αναπηρίας. Γιατί ε, δεν μπορεί κάθε φορά το άτομο με αναπηρία να φτάνει σε μια χώρα και να ξεκινάει η Οδύσσια να αναγνωριστεί Αυτά τα πράγματα είναι αφόρητα και δεν έχουν και νόημα σε μια Ευρώπη που υποτίθεται δεν θέλει να έχει σύνορα. Η Επιτροπή Αναφορών μπορεί να ασκήσει πολύ μεγάλη πίεση και να κάνει πάρα πολλά για να ανοίξουν τα μυαλά αυτών που πρέπει ε, ούτε καν στις κάρτες στάθμευσης για αναπηρικά αυτοκίνητα δεν έχουμε ενιαία. Δηλαδή η κάρτα των Βρυξελών δεν ισχύει στην Κύπρο. Ε, καταλαβαίνετε τι γίνεται εκεί. Μπορούμε πάρα πολλά να επιτύχουμε για να πιέσουμε. Όλοι συμφωνούν και κανείς δεν μετακινείται. Θα πρέπει τώρα να κινηθούν προς τη σωστή κατεύθυνση. Ευχαριστώ. Ακριβώς. Συμφωνούν, αλλά τίποτα δεν κινείται και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή όταν απευθυνθήκαμε για να δούμε τι γίνεται, αν υπάρχουν βελτιστές πρακτικές και πώς αντιμετωπίζονται αυτά τα πράγματα, σε θελοντική βάση, αυτό είναι μαύρη τρύπα. Όταν στέλνουμε κάτι, η απάντηση δεν έρχεται ποτέ. Είναι συνομιλητής και συνεργάτης μας εδώ η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και προσπαθεί να βρει τι συμβαίνει. Να σας πω ότι όταν εγκρίναμε ε, το, το νομοθέτημα για την προσβασιμότητα, το ίδιο είπε και το Συμβούλιο το Δεκέμβριο και το 2018 αναμένεται να ξεκινήσουν διαπραγματεύσεις τριμερούς διαλόγου. Ακόμα περιμένουμε. Και γνωρίζουμε ότι οτιδήποτε είναι σε θελοντική βάση, καταλαβαίνετε. Εγώ είμαι από τη Σουηδία. Είναι από τη χώρα αυτή ε, που ήταν ε, πρωτοπόρα για την προσωπική βοήθεια μέχρι πρόσφατα, που σιγά σιγά έχουμε δει να κατρακυλάει και η χώρα μου. Εμείς στα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα και η Επιτροπή μας θα πρέπει να τονίσουμε ότι η ελεύθερη κυκλοφορία είναι κάτι που αφορά τους πάντες και τους ανθρώπους με αναπηρίες. Και θα πρέπει να εξασφαλίσουμε αυτή η ελεύθερη κυκλοφορία να μην είναι ένα ωραίο όνειρο, αλλά πραγματικότητα για τους ανθρώπους. Και είναι υποχρέωσή μας, πιστεύω, αυτό, καθήκον μας. Εντάξει, νομίζω ότι πρέπει να κλείσουμε τώρα το θέμα αυτό. Ο αγώνας συνεχίζεται και δεν πρόκειται να ε, θα τα βάλουμε κάτω. Τι λέτε κύριε Μαριά. Έχω Μικρόφωνο κύριε Μαριά. Κυρία Πρόεδρε, έχω τις εξής προτάσεις. Βεβαίως θα κρατήσουμε ανοιχτή την αναφορά. Δεύτερον, όπως είπε η κυρία Κούνεβα, να στείλουμε μία επιστολή στο Δήμο των Βρυξελών, διότι οι Βρυξέλλες έχουν πάρα πολλά θετικά λόγω της λειτουργίας εδώ των ευρωπαϊκών οργανισμών και πάρα πολλά χρήματα που κερδίζουν, αλλά θα πρέπει και ο Δήμος να αντιληφθεί ότι έχει υποχρεώσει σε σχέση με την εφαρμογή της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας. Τρίτον, θα πρέπει να ζητήσουμε και θα μπορούσαμε και εμείς να αποστείλουμε μία επιστολή σε όλες τις μόνιμες αντιπροσωπείες των κρατών μελών που δεν συμμετέχουν στο πρόγραμμα αυτό έστω το εθελοντικό, το πιλωτικό διότι είναι μόνο οκτώ χώρες και εν προκειμένου πιστεύω ότι πρέπει να σταλεί η επιστολή και προς την μόνιμη αντιπροσωπεία της Ελλάδος και των άλλων χωρών για να μπουν έστω σε αυτό το πιλωτικό πρόγραμμα. Η επόμενη πρόταση αφορά να αποστείλουμε την ε, αναφορά για ενημέρωση εδώ στις αρμόδιες επιτροπές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Δηλαδή και στην Επιτροπή των Μεταφορών, γιατί έχει μεγάλη σημασία να προωθήσουμε την δυνατότητα του συνοδού είτε δωρεάν είτε με μια έκπτωση να μπορεί να συνοδεύει τα άτομα με αναπηρία. Δεύτερον, να ζητήσουμε την δυνατότητα αναγνώρισης, αμοιβαίας αναγνώρισης της κάρτας αναπηρίας μέχρι να εκδοθεί η Ευρωπαϊκή Κάρτα Αναπηρίας. Επομένως αφορά και τη ΛΥΜΠΕ, νομίζω ότι είναι θέμα και ελευθεριών. Και τέλος, να ζητήσουμε από την Επιτροπή Νομικών Υποθέσεων εδώ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να προβλέψει δικαίωμα αγωγής αποζημιώσεως των ατόμων με αναπηρία εφόσον δεν τηρούν οι εταιρείες μεταφορών, είτε οι αεροπορικές, είτε οι σιδηροδρομικές, είτε οι υπόλοιπες εταιρείες μεταφορών, τα δικαιώματά τους. Και εφόσον προσβάλλονται αυτά τα δικαιώματα, να υπάρξει δικαίωμα αγωγής αποζημιώσεως. Νομίζω με αυτόν τον τρόπο βγάζουμε και ένα γενικότερο συμπέρασμα από αυτή την αναφορά, όχι μόνο για το τι συμβαίνει στο Βέλγιο, αλλά όπως είπατε και εσείς, να πάρουμε πρωτοβουλίες σε ένα ευρωπαϊκό επίπεδο, πιέζοντας ως Επιτροπή και διαμορφώνοντας ένα πλαίσιο δράσης. Ευχαριστώ. Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ. Okay, let's do the We... Ωραία. Λοιπόν, προτείνω το εξή. Βεβαίω θα παραμείνει ανοιχτή η αναφορά. Πιστεύω, όπως ε, είπε και η κυρία Κούνεβα, ότι οι Βρυξέλλες θα πρέπει να είναι ένας φάρος και να δίνει το παράδειγμα και όχι ουραγός ε, στην προσβασιμότητα. Οι Βρυξέλλες, η καρδιά της Ευρώπης πραγματικά θα πρέπει να δώσει το παράδειγμα και να έχει ηγετική θέση. Θα συνεχίσουμε από εκεί. Ωραία, θα κάνουμε αυτό που είπε ο κύριος Μαριάς, να στείλουμε επιστολή στο Δήμο των Βρυξελών και να πούμε πού είναι ο φάρος της προσβασιμότητας οι Βρυξέλλες. Και να στείλουμε και άλλη επιστολή που είπαμε στην Προεδρία του Συμβουλίου και σε όλες τις μόνιμες αντιπροσωπείες λέγοντας ότι ξέρουμε ότι τώρα ε, θα έρθει στο τριμερή διάλογο κάποια στιγμή αργά ή γρήγορα η προσβασιμότητα και το ξέρουμε ότι είναι θελοντικό το πρόγραμμα αυτό το πιλωτικό αλλά και αναγνώριση αλλά τα καλύτερα παραδείγματα θα πρέπει να τα μοιραζόμαστε. Ποιες είναι οι δικές σας βέλτιστες πρακτικές και πώς θέλετε να τα μοιραστείτε και τι προβλέπετε. Και ας ελπίσουμε αυτή τη φορά να μην πέσουμε σε μαύρη τρύπα στο Συμβούλιο, να μας στείλουν κάποια απάντηση στην Επιτροπή μας. Αυτά. Εντάξει, αυτό μπορούμε να κάνουμε. Συμφωνείτε όλοι μαζί και παραμένω ε, στην άποψη, όπως είπε και η Ρώσα, ότι η Επιτροπή αυτή μπορεί να είναι πολύ χρήσιμη. Στην αρχή της αιτίας μας είπα ότι η προσβασιμότητα για τους ανθρώπους με αναπηρίες ε, θα πρέπει να είναι σε καλύτερη μοίρα στο τέλος της θητείας από ό,τι στην αρχή μας. Εκεί εμείς πραγματικά μπορούμε και πρέπει να ε, κάνουμε τη διαφορά. Ας προσπαθήσουμε ξανά λοιπόν. Και ας μην εγκαταλείπουμε ποτέ αυτή την προσπάθεια. Είναι πάρα πολύ σημαντική. Ωραία, σας ευχαριστώ πάρα πολύ και τώρα έχουμε κάποιους προσκεκλημένους. Είστε εσείς οι Φιλανδοί που ήρθατε τώρα, όχι. Καλώς. Ευχαριστούμε για την ανταλλαγή αυτή και πάμε στην επόμενη αναφορά υπαριθμών 745 και την 371. Είναι εδώ αναφέρον ο κύριος ε, Νταβίτ Νάχτ. Είστε εδώ. Εδώ είμαι. Εσείς είστε εδώ και έχετε και το λόγο για 5 λεπτά παρακαλώ. Σας ευχαριστώ που μου δώσατε λίγο χρόνο για να πάρω τον να παρουσιάσω το θέμα. Ήμουνα και πριν δύο χρόνια εδώ, δείχνοντας τις τεράστιες δυσκολίες που έχουν οι αθλητικογράφοι για να μπορούν να ενημερώνουν το κοινό για, τα, για τους αγώνες. Πριν δύο χρόνια είχα πει ότι είχαμε πάρα πολλά δικαιώματα τα οποία ζητούσαν για την αναμετάδοση ραδιοφωνικά των ποδοσφαιρικών αγώνων. Υπήρξαν δύο περιπτώσεις, επίσης επιπλέον πρόσφατα, 16 γιούρο ε, στην Γαλλία. Αυτοί οι οποίοι δεν ήσαν στις εταιρείες που είχαν τα δικαιώματα δεν μπορούσαν καν να είναι παρόντες στις συνεντεύξεις τύπου μετά το τέλος των αγώνων. Δεύτερη περίπτωση, Διεθνής Ομοσπονδία Χειροσφαίρησης και οι ιδιοκτήτες τους που είναι μια εταιρεία του Κατάρ ε, χρέωναν εκατομμύρια. Όταν έγινε το 16 πρωτάθλημα διεθνές στην Γαλλία ο γαλλικός νόμος ο οποίος απαγορεύει την ίσπραξη δικαιωμάτων για το ραδιόφωνο στην ουσία αγνοήθηκε και ήταν τόσο ακριβή η συμμετοχή στα γεγονότα αυτά που οι περισσότεροι αναγκάστηκαν να μην πάνε επί τόπου και να καλύψουν ε, την ραδιοφωνική αναμετάδοση από τα στούντιο στους ραδιοφωνικούς σταθμούς. Δεν μπορούμε να αποκλείουμε έτσι τον τύπο. Ε, στο ποδόσφαιρο σαν παράδειγμα υπάρχουν οι φωτογράφοι του αγώνα, της ομάδας μάλλον, ε, που έχουν όλα τα δικαιώματα, ενώ οι ανεξάρτητοι φωτογράφοι δεν έχουν την δυνατότητα να κάνουν οτιδήποτε. Σε ορισμένες χώρες οι ανεξάρτητοι φωτογράφοι μπορούν να πολλούν τις φωτογραφίες τους ή και να τις διαθέτουν δωρεάν. Νομίζω ότι τέτοιου είδους παραδείγματα Το κόρτμπαλ σαν παράδειγμα είναι ένα μικρό ε, σπόρο και έχουν αποκλείσει από τον τελικό στην Ολλανδία όλους τους φωτογράφες έδωσε τρεις φωτογραφίες στα μέσα ενημέρωσης μέσα από τους επαγγελματίες διαπιστευμένους φωτογράφους. Οι επαγγελματίες που πήγαν οι λίγοι στην ουσία δεν είχαν θέα γιατί τους την έκλειναν οι εκπρόσωποι της εταιρείας. Ε, στο ποδόσφαιρο τώρα ο Άγιαξ ευνοεί το ιδιωτικό του κανάλι, το Άγιαξ TV, ε, το καλοκαίρι, σαν παραδείγμα υπήρξε ο διορισμός νέου προπονητή, έδωσε μία και μοναδική συνέντευξη στο Άγιαξ TV, τα μέσα ενημέρωσης στο ραδιόφωνο δεν μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν ε, την δυνατότητα να θέσουν ερωτήσεις. Μπορούσαν μόνο να θέτουν ερωτήσεις ουσιαστικά και να ενημερώνονται από το κανάλι του Άγιαξ που δεν ήταν και πολύ αντικειμενικό. Και φυσικά ο Άγιαξ συνεχίζει ε, την τακτική αυτή καταρχώντας όλες τις press conference πριν από τους αγώνες του ε, και παραπέμπει μόνο στο κανάλι του. Το ίδιο γίνεται και στη Γερμανία όπου μόνο με ειδικέ προσκλήσεις ε, καλούνται να πάρουν μέρος οι δημοσιογράφοι. on the continent, the national associations και το θέμα λύθηκε στη Γερμανία τοπικά αλλά στην ουσία σε πάρα πολλές χώρες της Ευρώπης και εκτός Ευρώπης οι ομοσπονδίες των δημοσιογράφων αθλητικού τύπου και ραδιοφώνου έπρεπε να φέρουμε το θέμα αυτό ε, προς εξέταση μπροστά σας γιατί νομίζω ότι μια ενιαία ευρωπαϊκή αντίληψη θα ήταν χρήσιμη. Σας ευχαριστώ λέει η Πρόεδρος, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι εδώ. Είστε δύο, ένας από εσά θα πάρει το λόγο. Ο κύριος Μάρκ. Ευχαριστώ πρόεδρε. Θα αναφερθώ στη νέα αναφορά μόνο, γιατί η προηγούμενη απάντηση την οποία είχαμε δώσει για την 745 του 2013 έχει δοθεί. Η νέα αναφορά η 371 του 17 δίνει επιπλέον κάποιες πληροφορίες αλλά στην ουσία καλύπτει το ίδιο θέμα. Αναφέρουμε στην πιθανότητα άρνησης του δικαιώματος των μέσων ενημέρωσης να έχουν πρόσβαση στις αθλητικές διοργανώσεις. Εμείς παραπέμπουμε όμως την προηγούμενη απάντησή μας. Δεν μπορούμε να παρέμβουμε ουσιαστικά και δεν μπορούμε να παρέμβουμε γιατί οι συνθήκες δεν μας δίνουν την δυνατότητα να παρεμβαίνουμε στις διακανονιστικές ρυθμίσεις των αθλητικών οργανώσεων στην Ευρώπη. Και ακόμα και αν υπάρχει μια κάποια δυνατότητα για τα κράτη-μέλη να ζητήσουν εξαιρέσεις, αυτό καλύπτει κάποιες τοπικές ε, ε, τηλεοπτικές ε, εκπομπές και όχι γενικότερα το δικαίωμα των δημοσιογράφων. Εμείς λοιπόν παραμένουμε στη θέση μας και λέμε ότι δεν έχουμε καμία δυνατότητα και αρμοδιότητα να διερευνήσουμε τους ισχυρισμούς που έχουν καταθέσει οι αναφερόμενοι. Λοιπόν, συνάδελφοι, ο κύριος Μαριάς. Θεωρώ την ε, αναφορά αυτή ιδιαίτερα σημαντική, αλλά διαφωνώ με αυτά τα οποία λέει η Επιτροπή. Και θα επαναλαμβάνω εδώ και θα επαναλάβω μάλλον αυτά τα οποία είπα όταν συζητήθηκε η προηγούμενη αναφορά, η 745 του 2013 του κυρίου Βάρα. Το ποδόσφαιρο ή γενικώ τα αθλήματα αυτή τη στιγμή έτσι όπως εξελίσσεται η κατάσταση αποτελούν ένα οικονομικό αντικείμενο. Επομένως εφαρμόζεται και στο ποδόσφαιρο και στα υπόλοιπα αθλήματα τα οποία είναι επαγγελματικά η ίδια η συνθήκη, διότι έχουν οικονομικό αντικείμενο. Και θα πρέπει να δούμε εάν παραβιάζονται συγκεκριμένα οικονομικά δικαιώματα εν προκειμένου, ακόμη και των ίδιων των δημοσιογράφων οι οποίοι ασκούν και παρέχουν μια υπηρεσία η οποία υπηρεσία προβλέπεται στο πλαίσιο της λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το δεύτερο στάδιο που δεν εξετάζει η Επιτροπή στην απάντησή της είναι μήπως υπάρχει μια διαδικασία παραβίασης των κανόνων περί ανταγωνισμού. Δηλαδή μήπως οι διάφορες ομάδες υποδοσφαιρικές αλλά ταυτόχρονα και η UEFA και η FIFA επί της ουσίας με τους κανόνες που έχουν επιβάλει στην ουσία έχουν συγκροτήσει ένα καρτέλ και αυτό το καρτέλ διαμορφώνει τέτοιους όρους οι οποίοι στην ουσία παραβιάζουν τους κανόνες περί ανταγωνισμού και άρα έχει τη δυνατότητα να ελέγξει τη δραστηριότητα της Αθλητικής Ομοσπονδίας και της ΟΕΦΑ και της FIFA και των υπολείπων ομοσπονδιών η ίδια η Κομισιόν. Να αναφερθώ λοιπόν στην λειτουργία όλου αυτού του συστήματος και να πω ότι έχουμε ήδη μια πρώτη απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου στην υπόθεση ΚΟΧ που θεωρούσε ότι το συγκεκριμένο άθλημα είχε οικονομικό αντικείμενο και επομένως μπορούσε να ελεγχθεί η δραστηριότητα της, της Ομοσπονδίας την εποχή εκείνη. Δεύτερον, έχουμε την υπόθεση Μπόσμαν, η οποία δίνει τη δυνατότητα στην Επιτροπή να παρέμβει. Τρίτον, μου κάνει εντύπωση πώς δεν αξιοποιείται τη δραστηριότητα του κυρίου Μπάγκεμαν όταν ήταν μέλος της Κομισιόν και υπεύθυνο στην Επιτροπή Ανταγωνισμού που προσπάθησε να ελέγξει αυτό το καρτέλ και της FIFA και της UEFA και όλων των άλλων ε, ομοσπονδιών. Τέταρτον, μου κάνει εντύπωση που δεν λάβατε υπόψη ότι πριν λίγες μέρες η ίδια η Κομισιόν ελέγχει πλέον και κάνει παρεμβάσεις και έκανε ελέγχους στις εταιρείε διανομής αθλητικών προϊόντων και διανομής και μετάδοσης των αθλητικών γεγονότων κατά πόσο υπάρχει παραβίαση περί ανταγωνισμού. Άρα θα ήθελα να φύγετε από τη λογική που έχετε μπει και να δείτε ότι εδώ πρόκειται για ένα οικονομικό αντικείμενο και δεν μπορεί καμία ομάδα, είτε ποδοσφαιρική, είτε ομάδα μπάσκετ, είτε οποιαδήποτε άλλη ομάδα που ασκεί ένα άθλημα το οποίο έχει οικονομικό αντικείμενο, να δείτε λοιπόν πώς παραβιάζονται οι διατάξεις περί ανταγωνισμού και οι διατάξεις Ευρωπαϊκής Ένωσης περί ελεύθερης παροχής υπηρεσιών, διότι οι δημοσιογράφοι ασκούν ένα λειτουργήμα μεν, αλλά ταυτόχρονα και μια οικονομική υπηρεσία. Και όταν με άνισους όρους και με όρους τέτοιους που επιβάλλονται τους απαγορεύεται να ασκήσουν το δικαίωμά τους να λειτουργήσουν ως επαγγελματίες, εδώ έχουμε παραβιάσεις των διατάξεων της συνθήκης για παροχή υπηρεσιών, για τήρηση των κανόνων του ανταγωνισμού, για απαγόρευση λειτουργίας μονοπωλίων. Άρα λοιπόν αυτή είναι μία πλευρά την οποία δεν έχει λάβει υπόψη η Κομισιόν και εγώ πιστεύω ότι πρέπει να τη λάβει. Ταυτόχρονα υπάρχει και το δικαίωμα ενημέρωσης των ίδιων των πολιτών που φυσικά κατοχυρώνεται εν μέρη στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά νομίζω ότι πρέπει να δείτε με μια ευρύτητα τις διατάξεις περί ενημέρωσης των ίδιων των πολιτών και εκεί να έχετε και μια παρέμβαση. Αλλά δέστε επίσης ξαναγυρνώ στο οικονομικό πεδίο και τους τηλεθεατές ως λήπτες υπηρεσιών, τους πολίτες ως λήπτες υπηρεσιών, δηλαδή την πληροφόρηση που θα πάρουν, αλλά ταυτόχρονα και το δικαίωμά τους στην ψυχαγωγία. Δεν μπορεί λοιπόν να υπάρχουν αυτά τα αποκλειστικά δικαιώματα όλων αυτών των ομάδων, είτε είναι ποδοσφαιρό, ποδόσφαιρο, μπάσκετ κλπ, να έχουν τη δικιά τους τηλεόραση η οποία να απαγορεύει το δικαίωμα ενημέρωσης και πληροφόρησης ή να επιβάλλει τέτοιους οικονομικούς όρους στους επαγγελματίες, φωτογράφους, αθλητικογράφους, δημοσιογράφους που στην ουσία να παραβιάζει τους όρους λειτουργίας του ελεύθερου ανταγωνισμού. Εγώ νομίζω κυρία Πρόεδρε να κρατήσουμε ανοιχτή την αναφορά και να δούμε υπό ποιου όρους μπορούν να γίνουν επιπλέον βήματα. Διότι πλέον σε λίγο η UEFA και η FIFA που είναι κράτος σε κράτη θα βάλουν τέτοιους όρους οικονομικούς που ο μισός πληθυσμός θα αποκλειστεί από το δικαίωμά του να παρακολουθεί αυτή την ψυχαγωγία και οι δημοσιογράφοι δεν θα έχουν τη δυνατότητα μιας αντικειμενικής ενημέρωσης. Ευχαριστώ. Thank you very much. Ε, Virginie. Ευχαριστώ, Virginie. Ε, Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Είναι σύνηθε να έχουμε την ίδια απάντηση από την Κομισιόν στην Επιτροπή Αναφορών. Δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα δεν αφορά την Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν είναι θέμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αυτό μας κουράζει στο τέλος. Ειδικά σε τούτη την περίπτωση, γιατί όσον αφορά ε, ε, τις ευκαιρίες, ε, 7% του Ευρωπαϊκού ΑΕΠ ε, ακριβώς προέρχεται από τις αθλητικές δραστηριότητες και τον αθλητισμό. Ε, στην ε, περιγραφή σαν κατάσταση έχουμε και κάποια στοιχεία τα οποία ε, ε, ε, πραγματικά, όπως είπε και ο συνάδελφος Μαριάς, αποτελούν κατάφορη παραβίαση ευρωπαϊκών αρχών. Ε, ναι, ο καθένας έχει τη δυνατότητα βεβαίως να υπογράψει συμβόλαια με ε, κάποιον που προτιμάει, αλλά παρόλα αυτά υπάρχουν πάντα εχέγγυα, υπάρχουν πάντα προστατευτικά μέτρα. Ε, δεν είναι δυνατόν να έχουμε περιπτώσεις όπως σε αυτήν την περίπτωση όπου κάποιος για να μεταδώσει τα, την, βασική πληροφόρηση έχει τρομακτικές απαιτήσεις. Αυτό πραγματικά ε, αντιβαίνει στην αρχή ε, του δίκαιου ανταγωνισμού και του ε, ορθού ανταγωνισμού. Νομίζω ότι θα πρέπει να υπάρχει πάντα η δυνατότητα μια ορθή κάλυψη ενό αθλητικού συμβάντο. Και νομίζω ότι εδώ θα πρέπει να δούμε το δίκαιο στην πληροφόρηση. Γιατί μια αθλητική διοργάνωση, ναι βεβαίω θέλουμε να ξέρουμε τα αποτελέσματα κτλ. Αλλά την άλλη πλευρά είναι και καθαρά οικονομικό ε, συμβάν αλλά και ένα κοινωνικό συμβάν το οποίο αφορά ε, όλη την ε, κοινωνία γιατί ξέρουμε ότι ο αθλητισμός ξεπερνάει κατά πολύ τα στενά όρια του ίδιου του αθλητικού γεγονότος είναι ένα εργαλείο το οποίο χρησιμοποιείται παντιοτρόπως χρησιμοποιείται και στον πολιτικό στίβο και νομίζω ότι κατά την έννοια αυτή έχουν όλοι το δικαίωμα να έχουν σωστή πληροφόρηση. Δεν είναι δυνατόν να βλέπουμε ε, να είναι εντελώς κλειδωμένη οποιαδήποτε πληροφόρηση αφορά τέτοιου είδους γεγονότα και για λόγους καθαρά οικονομικούς. δεν είναι δυνατόν ε, η εικόνα των όσων συμβαίνουν σε ένα στάδιο να αποτελούν αποκλειστικό δικαίωμα ενός μεταδότη. Ε, γιατί ε, δεν είναι δυνατόν να μην ξέρουμε τι συμβαίνει μέσα σε, στο, στο στάδιο. Και υπάρχουν δημοσιογράφοι οι οποίοι είναι αθλητικοί δημοσιογράφοι, οι οποίοι έχουν τη δυνατότητα να καλύψουν αυτά τα γεγονότα. Είναι άνθρωποι οι οποίοι έχουν τη γνώση, έχουν τη δυνατότητα, έχουν την σφαιρικότητα αν θέλετε που χρειάζεται έτσι ώστε να μπορέσουν να μεταδώσουν αυτά τα συμβάντα και επομένως δεν είναι δυνατόν να βλέπουμε να είναι απολύτως κλειδωμένα ε, τέτοιου είδους συμβάντα και να μην ε, υπάρχει η δυνατότητα να βγουν προς τα έξω. Ε, βλέπουμε ότι αυτό συμβαίνει όλο και συχνότερα. Βλέπουμε ότι οι προϋποθέσεις είναι όλο και πιο απαιτητικέ, όλο και πιο δύσκολες, όλο και πιο αποκλειστικές. Εγώ πιστεύω λοιπόν ότι αυτή η αναφορά πρέπει να παραμείνει ανοιχτή ε, και θα πρέπει να δούμε αν υπάρχει διαδικασία επιπαραβάση, αν μπορεί να ξεκινήσει δηλαδή διαδικασία επιπαραβάση και θεωρώ ότι πραγματικά αυτό συνδέεται και με το δικαίωμα πληροφόρηση που ε- πρέπει να έχουν όλοι οι πολίτες τη Ευρώπη. Ευχαριστώ, ευχαριστώ λέει η Πρόεδρο. Ε, πρέπει να σας πω ότι και εγώ επί της αρχής ε, βλέπω με μεγάλη συμπάθεια το, το θέμα αυτό, αλλά φαίνεται ότι σε όσα είπε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συγκαταλέγεται και η γνωμοδότηση της Επιτροπής πολιτισμού η οποία φαίνεται να λέει ότι δεν υπάρχει παράβαση των, αρχών διανοητικής ιδιοκτησίας έτσι όπως ορίζονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση ε, και άλλωστε ε, και η ίδια η αναφορά δεν ενέχει οποιαδήποτε υπόνοια ε, παράβασης ε, του δικαίου Ε, γι' αυτό θα μπορούσαμε ε, και, γι' αυτό ακριβώς αναφέρεται ότι οποιαδήποτε παράβαση εφόσον και εάν υπάρχει θα πρέπει να φτάσει ενώπιον των εθνικών δικαστηρίων γιατί αυτά τα θέματα αποτελούν αποκλειστική αρμοδιότητα ε, των κρατών μελών. Αυτά έγραψε στη γνωμοδότησή της η Επιτροπή Πολιτισμού όσον αφορά το θέμα. Λοιπόν, νομίζω ότι είναι σαφέ. Ε, όλοι οι συνάδελφοι είπαν ότι θα πρέπει να παραμείνει ανοιχτή αυτή η αναφορά. Δεν μπορώ να κάνω διαφορετικά λοιπόν. Ε, θέλετε ε, μήπως να πάρετε ξανά το λόγο. Θα ήθελα μονάχα να αναφερθώ ε, συντόμως ε, ε, στην γνωμοδότηση της δικής σας Επιτροπής Πολιτισμού. Ναι, είναι γεγονός ότι είναι εθνική αρμοδιότητα, απλώς διαπιστώνουμε ότι υπάρχουν παρόμοια προβλήματα σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ενωσιακή Επικράτεια, άρα συμβαίνουν παρόμοια συμβάντα παντού. Απ' την άλλη πλευρά υπάρχουν αθλητικά γεγονότα τα οποία είναι διεθνή ε, είναι, αναφέρθηκε προηγουμένως η FIFA και η τηλεόραση δεν αφορά μονάχα τι χώρες τη Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και ολόκληρο τον κόσμο. Ε, υπάρχουν λοιπόν ε, πολλές περιπτώσεις αποκλεισμού και στην Αφρική όπου η ραδιοφωνική μετάδοση αποκλείεται ενώ γνωρίζομαι ότι είναι ο, το ραδιόφωνο το αποκλειστικό μέσο ενημέρωσης για τους ανθρώπους αυτούς στην Αφρική. Επομένως βλέπουμε ότι ε, υπάρχουν προβλήματα σε όλη την ενοχή Επικράτεια, άρα θα πρέπει να βρεθούν κάποια μέτρα τα οποία να είναι εγκάτσια και να αφορούν ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευχαριστώ πολύ Πρόεδρος, βεβαίως. Κύριε Μπαριά, πολύ σύντομα όμως σας παρακαλώ. Μα κυρία Πρόεδρε, διότι η Επιτροπή μας έχει ένα δυναμισμό. Βγάζουμε συμπεράσματα από τις συζητήσεις. Επομένως είναι σίγουρο ότι πρέπει να κρατήσουμε ανοιχτή την αναφορά αλλά θα έλεγα ότι πλέον η οικονομική διάσταση που αποκτά και η αναφορά αυτή, δηλαδή το δικαίωμα των δημοσιογράφων για πρόσβαση στους χώρους των αθλητικών γεγονότων, προκειμένου να ασκήσουν το επάγγελμά τους, το οποίο έχει μια οικονομική δραστηριότητα, σε συνδυασμό με το γεγονός ότι τα αθλητικά γεγονότα πλέον τα περισσότερα είναι πανευρωπαϊκά και ρυθμίζονται από αποφάσεις ευρύτερες ομοσπονδιών σε ευρωπαϊκό επίπεδο όπως είναι η UEFA ή σε παγκόσμιο επίπεδο όπως είναι η FIFA. Άρα λοιπόν να στείλουμε την αναφορά με ερώτημα στην Ήτρε εδώ τη δικιά μας Επιτροπή για να εξετάσουμε εάν υπάρχουν οι περιπτώσεις παραβίασης των κανόνων περί ανταγωνισμού και της άσκησης οικονομικού δικαιώματος των δημοσιογράφων για να μπορούν αυτοί να ασκήσουν το επάγγελμά τους, δηλαδή ως πάροχοι υπηρεσιών. Αυτή την πλευρά πρέπει να δούμε σε συνδυασμό με το ότι ήδη η Κομισιόν έχει κάνει ευκαιριαστικού ελέγχους σε τηλεοράσεις και σε επιχειρήσεις διανομής αθλητικού προϊόντος μέσω τηλεόρασης. Αυτές τις ημέρες γίνονται οι έρευνες για το αν υπάρχει παραβίαση περί ανταγωνισμού σε μεγάλα τηλεοπτικά δίκτυα. Να ακολουθήσουμε λοιπόν τις εξελίξεις, να μην μείνουμε στατικοί και να αφήναμε ανοιχτή την αναφορά στέλνοντας επίσης την αναφορά αυτή στην δικιά μας Επιτροπή εδώ στην Ήτρε. Ε, ωραία, εσείς προτείνετε να στείλουμε λοιπόν και στην Ήτρε, αλλά εγώ λέω και στην Έκον μάλλον. ναι, ναι, λέει η Πρόεδρο, είναι πολύ σημαντικό να τα στείλουμε στην ΕΚΟΝ από τη στιγμή που υπάρχει και μια οικονομική διάσταση για το θέμα αυτό. Έτσι θα κάνουμε λοιπόν. Καλώς λοιπόν. Θα δούμε ακριβώς αν μπορούμε να συνεχίσουμε και με αυτό τον τρόπο. Σας ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ για την παρουσία σας για μια ακόμη φορά. Λυπάμαι που δεν υπάρχουν πιο συγκεκριμένοι τρόποι να σας βοηθήσουμε, αλλά είναι ένα μικρό βήμα προς τα εμπρός. Ευχαριστώ λοιπόν. Συνεχίζουμε με την επόμενη παρακαλώ τώρα οδηγία. Είναι η 811 με 844 υπογραφές για τον ποταμό Σεβέζο ε, και για δύο λεκάνες ε, ε, διατήρησης ποσοτήτων ύδατος. Ο κύριος Τζοβάνι Κορτέζε έχει το λόγο. Ελπίζω οι Βρυξέλλες να μην σας ε, δείχνουν μόνο μια κακή εικόνα μέσω του καιρού. Σας καλωσορίζουμε λοιπόν. Έχετε το λόγο για πέντε λεπτά ο κύριος Κοτέσε. E Καλημέρα σε όλους. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας. Η 811 του 2017 αναφέρεται στα δύο, ε, στις δύο δεξαμενές ρύθμισης για τον ποταμό Σεβέσον. Αυτό είναι κάτι το οποίο θα κατα... δεν ακούγεται ο μιλητής γιατί ταυτόχρονα ακούγεται έντονα μουσική. Δεν είμαστε σε θέση να ακούσουμε αυτά τα οποία λέγει ο, ομιλητής che è a quota più alta e con l'aerodispersione We don't, we do not get the translation, so I don't know really what we. Δεν ακούμε τη διερμηνία. Τι να κάνουμε; Δεν μπορείτε να μιλάτε πάνω στο βίντεο. Α, τώρα εντάξει, χαμηλώσαμε λίγο τη μουσική. Παρακαλώ. L'interazione delle luride acque del Seveso con quelle. i διάχυση γενικά και μέσω της διήθησης ανάμεσα στο Σεβέζο και στη Φάλντα θα δημιουργήσει πάρα πολλά προβλήματα ιδιαίτερα από εκεί όπου προέρχονται τα μολυσμένα ύδατα. Τα έγγραφα τα οποία σας έχουμε στείλει εξηγούν τους λόγους για τον οποίο είμαστε εναντίον της κατασκευής αυτών των δύο δεξαμενών λεκανών αν θέλετε. Ε, θα δημιουργηθεί πρόβλημα στην χλωρίδα της περιοχής. Ήδη έχουν απομακρυνθεί πάρα πολλά φύτα Ήδη έχει ξεκινήσει η διαδικασία επί σε σχέση με τον ποταμό Σέβεζο, κάτι το οποίο έχει σαν στόχο την, τον καθαρισμό των υδάτων του ποταμού Σέβεζο και ταυτόχρονα τον σεβασμό της υγείας των κατοίκων και την αποφυγή της μόλυνσης των υπογείων υδάτων. Sì, continua il eh, dottor Borghi, sono io, un saluto a voi. Λέγομαι Μπόργη, ε, σας ευχαριστώ εδώ και 35 χρόνια είμαι παθολόγος και έχω ασχοληθεί ε, πάρα πολύ με τους ζωντανούς οργανισμούς. Αυτές οι δύο προτάσεις δεν είναι, δεν έχουν στόχο την ε, υδραυλική αν θέλετε διαρρύθμιση αλλά την δημιουργία δύο λεκανών απορροής οι οποίες θα δημιουργήσουν πάρα πολλά προβλήματα υγείας και νευρολογικά και ε, περιλαμβάνονται καρκινογενείς ουσίες, τετραχλωρικό εθάνιο το οποίο δημιουργεί προβλήματα επίσης νευρολογικά και καταλαβαίνετε όπως βλέπετε ε, και εδώ ακόμα και σε περιπτώσεις βροχής υπάρχουν προβλήματα, η διήθηση από τις δύο λεκάνες θα μολύνουν τα υπόγεια ύδατα ε, και θα δημιουργήσουν προβλήματα στην υγεία των κατοίκων. Και υπάρχει εκτός από τη μόλυνση των υδάτων και μόλυνση ε, της ατμόσφαιρας ε, όταν εξατμίζονται μετά από τις βροχές οι ουσίες αυτές μέσω της εξάτμισης των υδάτων. Είναι λοιπόν μια προαναγγελθήσα καταστροφή. Παραβιάζει τις οδηγίες, εμείς ζητάμε απλά τον σεβασμό των κανόνων που διέπουν την προστασία της υγείας των κατοίκων. Είμαστε όλοι υπεύθυνοι για την κατάσταση αυτή και πρέπει να αναλάβουμε δράση. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας. Καλή σας μέρα. Λέγομαι Κορτέζη, είμαι μοριακή βιολόγος και, βιολόγος και έκανα ε, διάφορες ε, έρευνες όσον αφορά ε, τα, τις ουσίες τις οποίες βρίσκονται ε, στον ποταμό Σεβέζο. Έχουμε πρώτα απ' όλα ε, οι οποίοι μπορούν να αποτελέσουν ενδοκρινικούς διαταράκτες. άλλες όπως το, την τραζίνα ή το νίκελ που μπορούν να δημιουργήσουν προβλήματα όσον αφορά ε, την ε, όγκους, δημιουργία όγκων κτλ. Το χλωρομεθάνιο επίσης, το οποίο είναι ε, ουσία καρκινογόνος και η οποία δεν πρέπει να έρθει σε επαφή με τον υδροφόνο ορίζοντα. Υπάρχει άλλο στοιχείο το οποίο είναι η γλυφοζάτη, η οποία είναι αποδεδειγμένος ενδοκρινικός διαταράκτης καθώς επίσης και διαταράκτης του P14 και προκαλεί προβλήματα ε, όσον αφορά τον μεταβολισμό μας. Ε, τέτοιες ουσίες μπορούν να δημιουργήσουν προβλήματα στο μεταβολισμό που με τη σειρά του θα ε, δημιουργήσει προβλήματα λοιμώξει κλπ. Ε, χρόνια προβλήματα. Ε, είναι γεγονός ότι με την παρουσία όλων αυτών των ουσιών τα, τα ύδατα δεν είναι καθόλου καθαρά. Ευχαριστώ πολύ λέει η Πρόεδρος. Ε, ευχαριστώ που παραμείνετε στα χρονικά σας όρια. Έχουμε σήμερα μαζί μας και την Μάγδα Μπερέτα η οποία είναι η Δήμαρχος του Σενάγκο. Δύο λεπτά έχετε το λόγο παρακαλώ κυρία Δήμαρχε. Αξιότιμα μέλη της Επιτροπής, λέγομαι Μάγδα Μπερέτα και είμαι ε, ε, δήμαρχος προτέμπορε της, ε, του Δήμου του Σενάγκο και πραγματικά δεν έχω άλλη επιλογή από το να υποστηρίξω τον κύριο Τζοβάνι Κορτέζε για την αναφορά του όσον αφορά τη δημιουργία τεχνητών λιμνών συγκράτησης υδάτων στο Σεβέζο. Από το 2010 μέχρι και σήμερα και οι υποφαινόμενοι και όλοι οι δήμαρχοι προκάτοχή μου από οποιοδήποτε κόμμα και αν προέρχονταν ε, ε, ελάβαμε την εντολή από το Δημοτικό Συμβούλιο να εκπροσωπήσουμε το Σενάγκο ε, με την έννοια αυτής της αναφοράς και για τους λόγους που θα αναφέρω σύντομα. Πρώτα απ' όλα το Σενάγκο αποτελεί ένα άνθος στην βόρεια περιοχή του, του Μιλάνο. Όμως τα τελευταία χρόνια το πρόβλημα το περιβαλλοντικό ε, έχει δημιουργήσει πάρα πολλά προβλήματα. Ε, αποφασίστηκε η δημιουργία αυτών των τεχνητών λιμνών συγκράτησης υδάτων που θα προκαλέσει σημαντικά προβλήματα ε, στην περιοχή μας. Έχει προβληθεί επίσης η τσιμεντοποίηση 17 εκταρίων που συμπεριλαμβάνουν και το πάρκο του Γκροάνε το οποίο είναι πάρα πολύ μεγάλη επιφάνεια. Μετά από την αστικοποίηση του του, του Χίντερλαντ του Μιλάνο καθώς επίσης και λόγω των επιλογών που έκαναν ε, οι γειτονικέ ε, ε, περιοχές και οι δήμοι εμείς βρεθήκαμε να πρέπει να πληρώσουμε τον πιο, το πιο υψηλό κόστος τα τελευταία χρόνια δόθηκε η δυνατότητα να μεταφερθούν ακόμα περισσότερο να, μετα, μετατοπιστεί το εύρος του καναλιού Σκολματόρες στα βόρειο-δυτικά που θα μπορούσε να ε, λύσει κάποια προβλήματα. Εν πάση περιπτώσει, τα τελευταία χρόνια επίσης ε, οι γειτονικέ ε, περιφέρειες αποφάσισαν να αλλάξουν την χωροταξία για να δώσουν περισσότερο χώρο για οικοδόμηση. Αυτήν την και επομένως θα δημιουργηθούν ακόμα περισσότερα προβλήματα στον ήδη επισφαλή, στην ίδια επισφαλή ισορροπία ε, της ε, περιοχής και ε, πιστεύουμε ότι θα υπάρξει και αύξηση των προβλημάτων υγείας. Είναι γεγονός ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση συχνά έχει πει ότι το ποταμό Σεβέζο βρίσκεται μεταξύ το, είναι τρίτο πιο μολυσμένο ποτάμι στην Ευρώπη. Δεν είναι δυνατόν αυτή η κατάσταση να σας αφήσει και εσάς αδιάφορος γιατί τα προβλήματα είναι πολλά και η υγεία των ε, πολιτών επισφαλής. Ε, ε, συγκεκριμένα αυτές οι τεχνητές λίμνες συγκράτησης υδάτων μπορεί να προκαλέσουν προβλήματα όσον αφορά την ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα. Επίσης θα προκαλέσουν μόλυνση του υδροφόρου ορίζοντα. Γι' αυτό ακριβώς μας προκαλεί έκπληξη και δεν κατανοούμε τους λόγους για τους οποίους οι περιφερειακές αρχές αποφάσισαν να προχωρήσουν στη δημιουργία αυτών των τεχνικών ε, των λιμνών. Ε, θα πρέπει οπωσδήποτε να αναρωτηθούμε για τι ε, τις επιπτώσεις οικονομικές, κοινωνικές και υγείας που θα έχουν αυτές οι τεχνητές λίμνες. Και θα πρέπει να σταματήσουν όλες αυτές οι δράσεις. Εξ ονόματος, λοιπόν του Δήμου του Σενάγκο και βάσει της πολιτικής εντολής που έχω σας ζητώ να προχωρήσετε σε απαγόρευση της δημιουργίας αυτών των τεχνητών λιμνών. Ευχαριστώ. Uh, Ευχαριστώ. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, όπως είπαμε προηγουμένως, σήμερα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν πρόκειται να σχολιάσει την παρουσίαση των αναφερομένων, αλλά ταυτόχρονα θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τους αναφερομένους για την ε, τόσο ακριβή και πιστή ε, περιγραφή της ε, κατάστασης για τον ενδεχόμενο κίνδυνο που μπορεί να εγκυμονεί ένα τέτοιο έργο για το περιβάλλον και για τον άνθρωπο. Θα αναλύσουμε τα έγγραφα αυτά, θα τα μελετήσουμε, θα τα αξιολογήσουμε και θα σας στείλουμε τις ε, απαντήσεις και τα συμπεράσματά μας εν ευθέτω χρόνο. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ για τη δήλωση αυτή. Γνωρίζαμε ότι δεν θα μας δίνατε σήμερα νέες πληροφορίε και απαντήσεις και ξέραμε ότι ήταν λίγο πρόωρο αλλά έλαβαν μια πολιτική απόφαση οι συντονιστέ να το εγγράψουν στην ημερήσια διάταξή σου για να εμπνευστείτε κι εσεί οι ίδιοι για το τι συνέχεια θα δώσετε. Ε, αρχίζει η συζήτηση. Ελενόρα Εύη πρώτη. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα ήθελα να υπογραμμίσω ότι το σχέδιο αυτό και η σχετική αναφορά έχει σχέση με κάτι το οποίο γνωρίζουμε εδώ στην Επιτροπή εδώ και καιρό. Οι αναλύσεις και οι αξιολογήσεις τις οποίες έχουμε κάνει επανέρχονται. Τι εννοώ. Ενθυμούμεθα ότι στην Ιταλία εμείς καταναλώνουμε τις δυνατότητες που δίνει η γη με τρομερό ρυθμό κάθε τρία δευτερόλεπτα, κάθε δευτερόλεπτο μάλλον, τσιμεντοποιούνται τρία τετραγωνικά μέτρα, 60 εκτάρια την ημέρα. Τσιμεντοποιούμε λοιπόν την χώρα μας και ε, το Βόρειο Μιλάνο είναι από τις πιο τσιμεντομένες περιοχές, το 70% της περιοχής καλύπτεται. Έχουμε στην ουσία εμείς ε, μετατρέψει τους ποτανού μας σε κανάλια. Ε, περικλείουμε με τσιμέντο τις όχθες του ποταμού και τους μικραίνουμε την έκταση. Αυτό είναι κάτι το οποίο φυσικά θα έχει συνέπειες στην ε, οικολογία της περιοχής Έχουμε βιώσει τις ε, δραματικές ε, ε, εμπειρίες της μόλυνσης και της μείωσης των υπογείων υδάτων. Γι' αυτό λοιπόν θα πρέπει να υπάρξει μια απάντηση εγκάρσια από την πολιτική εξουσία. Υπάρχουν προτάσεις σε επίπεδο τοπικό και περιφερειακό και δυστυχώς το μόνο το οποίο έχουν προτείνει μέχρι τώρα είναι συνολικά πέντε λεκάνες απορροής, συλλογής μάλλον, είναι ένα σχέδιο παλαιό, 20 ετές τουλάχιστον, το οποίο έχει σαν στόχο με κατεπήγοντα χαρακτήρα να δώσει μία απάντηση αγνοώντας τις μακροπρόθεσμες συνέπειες και αγνοώντας τον γενικότερο προγραμματισμό των υδάτινων πόρων που απαιτεί η περιοχή. Θέλω να ευχαριστήσω λοιπόν όλους ε, τους ε, ομιλητές που παρουσίασαν τις αναφορές τους. Υπάρχουν πάρα πολλοί λόγοι και τεχνικού τύπου, σαν παράδειγμα ένα τέτοιο σχέδιο ε, στην ουσία λαμβάνει υπόψη τον, το βάθος το οποίο έχουν οι δεξαμενές αυτό και το οποίο ε, φτάνει σε χαμηλότερο επίπεδο από το ανώτερο επίπεδο των υπογείων υδάτων. Είναι κάτι το οποίο είναι απαράδεκτο και φύγει ε, τα ύδατα τα οποία χρησιμοποιούν και έχουν ανάγκη οι κάτοικοι της περιοχής. Είναι απαράδεκτη αυτή η ρύθμιση και βλέπουμε ότι στην ουσία έχουμε να κάνουμε με μια ουσιαστική μόλυνση των υπογείων υδάτων με όλες τις συνέπειες που θύμισαν οι προηγούμενοι ομιλητές. Ξέρετε ότι υπάρχουν ε, πάρα πολλές εκροές ε, ε, παράνομες που έχουν ανοιχνευθεί, απορρίπτονται ουσίες παράνομα στον ποταμό Σέβεζο και όχι μόνο αυτό, έχουμε πραγματικά και, ε, και πρόβλημα με την ποιότητα, εν πάση περιπτώσει, του χώματος, της επιφάνειας της περιοχής, κάτι το οποίο έχει δημιουργήσει προβλήματα στις ε, δυσκολίες ε, της ποιότητας του εδάφους και δημιουργούνται περαιτέρω δυσκολίες επεξεργασίας ε, της επιφάνειας του εδάφους. Το σχέδιο που προτείνεται δεν λύνει το πρόβλημα, είναι μια ξεπερασμένη απόφαση. Στην ουσία επιβάλλει το μεγάλο έργο εις βάρος των επιμέρους μικρότερων και περισσότερων έργων που θα ήταν πολύ πιο αποτελεσματικά. Υπάρχουν καινοτόμε λύσεις, υπάρχουν καινοτόμε προτάσεις σε διάφορες περιοχές της Ευρώπης. Εμείς σαν κίνημα των πέντε αστέρων έχουμε ζητήσει να υπάρξει ακρόαση για την αναφορά αυτή. Βέβαια το κάναμε γρήγορα και αυτό δεν έδωσε χρόνο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. όχι όμως για να δημιουργήσουμε θέμα στην Επιτροπή, αλλά γιατί το έχουμε ήδη συζητήσει στο παρελθόν σαν κίνημα των πέντε αστέρων σε όλα τα επίπεδα είμαστε παρόντες και κινητοποιούμεθα εναντίον του προγράμματος αυτού, του σχεδίου αυτού και σε κοινοτικό επίπεδο και σε περιφερειακό επίπεδο και σε εθνικό επίπεδο και σε ευρωπαϊκό. Ζητώ να παραμείνει ανοιχτή η αναφορά, να στείλουμε μια επίσημη επιστολή και στις περιφερειακές και τοπικές αρχές, των Δήμο του Μιλάνου, σαν παράδειγμα που προωθεί αυτή την πρωτοβουλία που έχει χρηματοδοτήσει ένα τμήμα των έργων αυτών. και σε σχέση με αυτά τα οποία μόλις είπε η Δήμαρχος ε, μετά από τους ομιλητές που κατέθεσαν την αναφορά θα ήθελα να πω ότι βρίσκω λίγο επικίνδυνο να δίνουμε το λόγο στις τοπικές αρχές εγώ είμαι ικανοποιημένη από την στήριξη των δημοτικών αρχών στην αναφορά αυτή, αλλά θα ήθελα να προειδοποιήσω ότι αυτό θα μπορούσε να γίνει μια μονιμότερη πρακτική και θα μπορούσε να υπονομεύσει το μέσο των αναφορών το οποίο έχει δημιουργηθεί για τους πολίτες τους μεμονωμένους και οι τοπικές αρχές έχουν άλλους τρόπους και λόγους να εκφραστούν δεν πρέπει να δημιουργηθεί ένα προηγούμενο. Κατανοούμε φυσικά την παρέμβαση η οποία έγινε αλλά δεν είναι πάρα πολύ σωστό να μην δίνουμε το λόγο στους πολίτες όσο πρέπει. Έχουμε πολλές φορές ακούσει δημάρχους, αλλά είχαν υπογράψει οι ίδιοι τις αναφορές, ενώ η κατάσταση αυτή εδώ είναι διαφορετική και δεν θα πρέπει να επαναληφθεί. Eleonora, you know what I would like you. Ευχαριστώ. Κοιτάξτε, να το ξανασκεφτείτε πριν αρχίσετε να διαφημίζετε το κόμμα σας εδώ. Αν αρχίσουμε έτσι, το ίδιο θα κάνει το ΕΛΚ και οι σοσιαλιστές. Εδώ είμαστε για να ακούμε τους αναφέροντες και να είμαστε όσο γίνεται πιο αμερόληπτοι. Μην κάνετε ε, τέτοια τώρα και δώσετε το κακό παράδειγμα. Θα αρχίσουν τα διάφορα πολιτικά κόμματα να ε, περιαυτολογούν και να πενεύουν το κόμμα τους. Ας είναι αυτό εξαίρεση, να μην γίνει ο κανόνας. Και ε, σε ό,τι αφορά τις επικρίσεις, ότι έχουμε προσκαλέσει τις αρχές τοπικής αυτοδιοίκησης, αυτό είναι πάγια πρακτική. Ποτέ δεν δεχόμαστε εταιρείε εδώ, αλλά τους μόνιμους αντιπροσώπους και την τοπική αυτοδιοίκηση είναι ανεξαρτήτως πολιτικής τοποθέτησης και παράταξης. Ένα δημοκρατικό σώμα όπως είναι το δικό μας, τους δίνουμε το λόγο, έχει δημοκρατικό βήμα. Θα δώσω το λόγο στον Πέτερ για... Συγγνώμη κυρία Πρόεδρε, διακόπτη κυρία Εύη στα αγγλικά. Θα ήθελα να ξεκαθαρίσω και να τονίσω αυτό που είπα, ότι Βεβαίω είναι ευπρόσδεκτη λίμωνο η παρουσία των αρχών της τοπικής αυτοδιοίκησης όπως και στο παρελθόν. Παρ' όλα αυτά, αυτό ήρθε μετά από πρόσκληση των συντονιστών ή επειδή ε, η δήμαρχος ήταν αναφέρουσα. Ε, είναι λίγο διαφορετική η κατάσταση και θα πρέπει να το σημειώσουμε και να το έχουμε υπόψη μας για να μην δημιουργήσει προηγούμενο. Και προφανώς δεν εκμεταλλεύομαι αυτή την αναφορά για να προβάλλω το κόμμα μου. Είμαστε όλοι εδώ για να ακούσουμε τις αναφέροντες. Εδώ στην Επιτροπή μας καλά θα κάναμε να μην αναφέρουμε καν το όνομα του πολιτικού μας κόμματος. Απλώς να μιλούμε για το στόχο και το περιεχόμενο της αναφοράς και τον τρόπο ε, που θέλουμε να προχωρήσουμε. Αυτός είναι ο τρόπος λειτουργίας και ο στόχος της Επιτροπής μας. Ο Πέτερ Γιά. Ευχαριστώ πολύ. Χαίρομαι και εγώ που έχουμε την αναφορά αυτή στην ημερήσια διάταξη. Äh, είναι πολύ σημαντική αυτή, αλλά το πρόβλημα δεν είναι μόνο αυτό, είναι και διαρθρωτικό, είναι δομικό. Και είπαμε να το εγγράψουμε στην ημερήσια διάταξη, ακόμα και δεν έχουμε ακόμα την απάντηση Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Αυτό είναι το πρόβλημα όταν έχουμε τα περιβαλλοντικά. Το πρώτο βήμα είναι ότι καταγγέλουν οι αναφέροντες και μετά πάντα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχουμε πλήρη εμπιστοσύνη στα κρατημέλη ότι σέβονται ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία στο εκαίρεο κλπ. Και, δεν έχουμε κανένα λόγο να επέμβουμε. Αυτά λέει η Κομισιόν Παγίω. Μετά έχουμε ένα δεύτερο βήμα. Όταν ολοκληρωθεί αυτό το έργο, μετά τη μελέτη σκοπιμότητας και περιβαλλοντικού αντικτύπου, πώς να το διορθώσεις. Ακριβώς για αυτά τα έργα που έχουν ε, αντίκτυπο στο περιβάλλον χρειάζεται εγκαίρως επικοινωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των κρατών μελών και της ε, τοπικής αυτοδιοίκησης. Και θα ήταν ένα καλό παράδειγμα αυτό που κάνουμε σήμερα που το συζητούμε και βρίσκω θετικό αυτό που λέει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ακούσαμε τους αναφερομένους και καλούμε τις αρχές να λάβουν θέση αλλά παραμένουμε σε εντατική επαφή και στενή και όχι μόλις ολοκληρωθεί το έργο. Βεβαίως να παραμείνει ανοιχτή αναφορά και οι αναφορές και περιμένουμε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να διαβιβάσει ε, αυτά που λένε οι ε, ενδιαφερόμενοι να τα ελέγξει, να τα εξετάσει και να τα δούμε την άλλη εβδομάδα αυτά κυρία Πρόεδρε με τον ε, Αντιπρόεδρο Τίμερμανς. Γιατί θα του ασκήσω αυτή την κριτική. Καλύτερη επικοινωνία χρειάζεται μεταξύ της Επιτροπής Αναφορών, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και των κρατών μελών. Το πώς θα γίνει αυτό καλά κάνουμε και το συζητάμε σήμερα που είναι σε πρώιμο στάδιο και δεν έχει ολοκληρωθεί το έργο. Ευχαριστώ πολύ θα παραμείνει ανοιχτή αναφορά. Δεν αμφιβάλλω για την επιμέλεια για στη μελέτη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αλλά εδώ χρειάζεται διπλή προσοχή και εγρήγορση. Ευχαριστώ πολύ, ο κύριος Ευχαριστώ. Νομίζω ότι τα επιχειρήματα είναι αρκετά ε, πιστικά έτσι ώστε να τα αποδεχτούμε έτσι ώστε να μας οδηγήσουν και όλες να παραμείνει ανοιχτή αυτή η αναφορά. Αναρωτιέμαι ακριβώς γιατί τις τελευταίες μέρες ε, από ό,τι κατάλαβα και από ό,τι γνωρίζω και θα θα ε, ε, έχει μπλοκάρει η κατάσταση γιατί ε, η εταιρεία η οποία είχε κερδίσει το διαγωνισμό ε, αποφάσισε ε, να μην προχωρήσει. Να μιλάτε στο μικρόφωνο παρακαλώ. Δεν έχουν ξεκινήσει οι εργασίες, επομένως είμαστε στην κατάσταση που περιέγραψε ο προηγούμενος ομιλητής. Εγώ θα ζητούσα να βγούμε από τις τυπικές διαδικασίες και να προτείνω στην Πρόεδρο, μια και όλοι συμφωνούμε και δεν υπάρχουν αμφιλεγόμενα σημεία, να αποσταείλει επιστολή και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, έτσι ώστε να επιταχύνει την γνωμοδότησή της όσον αφορά ε, το επίδικο ζήτημα και το έργο αυτό. Και νομίζω ότι θα πρέπει, είναι χρήσιμο και σωστό να απευθυνθούμε και στις Ιταλικές αρχές. Ας κάνουμε λοιπόν μια επιστολή εξ ονόματος όλης της Επιτροπής, εξ ονόματος της Επιτροπής δηλαδή να υπογράψει η Πρόεδρος, έτσι ώστε να ανακληθούν οι εργασίες μια και βλέπουμε ότι η εταιρεία που κέρδισε τον διαγωνισμό ε, φαίνεται να μην θέλει να προχωρήσει. Και ε, να σταματήσουμε λοιπόν το έργο μέχρι ότου η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και εμείς οι ίδιοι ε, με τα λόγου γνώσεως γνωμοδοτήσουμε. Γιατί διατρέχουμε τον εξής κίνδυνο ε, όλοι έχουμε την ίδια άποψη με τους ε, αναφερόμενους ε, και όλοι συμφωνούμε και όλα καλά και όμορφα, αλλά φτάνουμε τελικά σε ένα σημείο που έχει προχωρήσει τόσο πολύ το έργο που δεν μπορεί να γυρίσει πίσω. Γι' αυτό λοιπόν πριν ξεκινήσει και πριν προχωρήσει το έργο πιστεύω ότι πρέπει να κινηθούμε. Γι' αυτό λοιπόν όλοι μαζί η Πρόεδρος να αποστείλει μία επιστολή στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή αφενός και στις Ιταλικές Αρχές αφετέρου, έτσι ώστε δρατώμενη της ευκαιρίας που η εταιρεία που έχει αναλάβει το έργο ε, δεν θέλει να το προχωρήσει, να σταματήσει να υπάρξει ανάκληση των εργασιών έτσι ώστε να μην διακινδυνεύσουμε τελικά απλώς και μόνο να αποτελέσουμε αντίχηση των προβλημάτων χωρίς να μπορέσουμε να παρέμβουμε με οποιοδήποτε τρόπο. Νομίζω ότι με τον τρόπο αυτό βοηθάμε ε, και τους ε, αναφερόμενους. Ε, και ναι, εδώ μιλάμε για, μια μικρή, για ένα μικρό δήμο ε, που έκανε πάρα πολλές σημαντικές προσπάθειες, ε, πολλές επενδύσεις ε, μεταξύ άλλων και ευρωπαϊκές έτσι ώστε να διατηρήσει το πάρκο στην περιοχή, άρα να μην τα καταστρέψουμε όλα τώρα. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Βάλλη. Ευχαριστώ Πρόεδρε, θα είμαι σύντομος. Εγώ προέρχομαι από το Μιλάνο και νομίζω ότι οι τεχνικές λεπτομέρειες που έδωσαν οι αρμόδιοι υπογραμμίζουν αυτό το οποίο και εμείς θέλουμε, να υπάρξει δηλαδή ε, ξεκάθαρη ενημέρωση για την ποιότητα των υδάτων αυτών, να δούμε ποιοι είναι οι κίνδυνοι για την υγεία των καταναλωτών που υποφέρουν από την ποιότητα της, του αέρα και των υδάτων. Θα πρέπει να βρούμε μία λύση λοιπόν για να αποφύγουμε έτσι ώστε όταν υπάρχουν πλημμύρες και καταιγίδε να μην δημιουργούνται προβλήματα στις μετακινήσεις αλλά δεν θα πρέπει το μεγάλο αυτό έργο να δημιουργήσει περισσότερα προβλήματα στην υγεία των πολιτών μολύνοντας τα υπόγεια ύδατα και καλό θα είναι στην επιστολή που θα στείλουμε να δούμε τι μέτρα μπορεί να ληφθούν έτσι ώστε να μην κατασκευαστούν αυτές οι λεκάνες, οι δεξαμενές που θα δημιουργήσουν όλα τα προβλήματα τα οποία ακούσαμε. Δεν θέλω να μακρηγορήσω, νομίζω ότι το θέμα αυτό διευκρινίστηκε από τις τεχνικές λεπτομέρειες οι οποίες δόθηκαν. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Εγώ θα είμαι πάρα πολύ σύντομος. Είναι σημαντικό αυτό το πρόβλημα περιβαλλοντικό, αλλά εφόσον αφορά τη δημόσια υγεία, και αυτό είναι το σημαντικό για μας, νομίζουμε ότι θα πρέπει να παραμείνει ανοιχτή αναφορά. so that to come to a good για κάποιο διάστημα ε, μέχρι να ολοκληρωθεί με επιτυχία. Ευχαριστώ. Ολοκληρώνεται εδώ ο κατάλογος των ομιλητών που είχα και με χαρά θα ξαναδώσω το λόγο στους αναφερομένους. Δεν ξέρω αν θέλετε να προσθέσετε τίποτα. Δύο λεπτά το πολύ. Non posso che ringraziarvi. Δεν μπορώ παρά να σας ευχαριστήσω όχι μόνο για την υποδοχή και την ευγένεια αλλά και γιατί αυτό το οποίο εμείς αναζητήσαμε να σας παρουσιάσουμε είναι κάτι το οποίο κινητοποίησε την ευαισθησία σας. Το Σενάγκο έχει δώσει το 43% στο πάρκο της Γκροάνα. Αν αρχίσουμε τώρα να βγάλουμε 17 εκτάρια, 100 δηλαδή 70.000 τετραγωνικά μέτρα, είναι κάτι το οποίο ε, δεν θα εξυπηρετήσει τα εδάφη των τοπικών, τα οποία ελέγχουν οι τοπικές αρχές. Το πρόβλημα λοιπόν είναι η μόλυνση της περιοχής γενικότερα. Τα νερά του Σέβεζο ε, στην ουσία είναι πιο χαμηλά από ε, το ύψος το οποίο βρίσκονται τα υπόγεια ύδατα και είναι βέβαιο ότι θα υπάρξει μία μόλυνση. Και ακόμα και υποτίθεται ε, το επίπεδο απομόνωσης από αργυλώδη πετρώματα το οποίο σκοπεύουν να κάνουν για να προστατεύσουν τα υπόγεια ύδατα, τον υδάτινο ορίζοντα δεν είναι κάτι το οποίο ε, θα λειτουργήσει. Είμαι βέβαιος ότι θα κάνετε το σωστό και θα εξετάσετε το θέμα αυτό με την απαιτούμενη προσοχή. να κοιτάξτε να προσθέσω κάτι που δεν ακούστηκε, που είναι σημαντικό. Κάποια από τα προβλήματα που δημιουργούνται ε, έχουν ε, κάτι, έχουν σαν στόχο όχι μόνο εμάς που ζούμε εκεί το 2018 αλλά έχουν τεράστια χρονική διάρκεια και θα επηρεάσουν αρνητικά τις επόμενες γενναίες και παθολογίες όπως η λευχαιμία που συνδέεται με συγκεκριμένες ουσίες που διαχέονται είναι σαφές ότι όσοι αρρωστήσουν από τέτοιου είδους παθολογίες δεν έχουν προσδόκιμο ζωής πάνω των 12 μηνών. Θέλω να σας ευχαριστήσω για το ενδιαφέρον σας και αν έχετε ανάγκη από περισσότερα στοιχεία είμαστε στη διάθεσή σας να επικοινωνήσουμε. Σας ευχαριστώ όλους. Σου κλείνουμε λοιπόν προς το παρόν την υπόθεση αυτή. Θα επανέλθουμε όταν έχουμε μια πλήρη απάντηση της Ευρωπαϊκής <coughs> Επιτροπής και εν τω μεταξύ θα στείλουμε και μία αποστολή στις τοπικές και περιφερειακές αρχές όπως ζητήθηκε από ορισμένους συναδέλφους. Όταν έχουμε λοιπόν μία πλήρη απάντηση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα έχουμε περισσότερα στοιχεία. Σας ευχαριστώ όλους που ταξιδέψατε εδώ. Σας εύχομαι καλή επιστροφή, καλό ταξίδι και θα συνεχίσουμε να επικοινωνούμε. Περνάμε τώρα στην επόμενη, την 857 για την δίγλωση εκπαίδευση στα καταλωνικά σχολεία για τις οικογένειες που εγκαθίστανται στην περιοχή. Έχει κατατεθεί η αναφορά από την Άννα Λοσάδα. Έχει τον λόγο για 5 λεπτά. Okay, my uh, ε, δικό μου λάθος, λέει η Πρόεδρος. Έγινε κάποιο λάθος. Στο φάκελό μου. Πρώτα έχουμε την προηγούμενη αναφορά υπαριθμών 857 εξ ονόματος ομάδας πολιτών Impulso Ciudadano, ε, όθηση πολίτων, ε, σχετικά με πινακίδες εμπορικά καταστήματα της Καταλωνίας. Στη συνέχεια εσείς με αυτή τη σειρά έχει εγγραφεί στην ημερησία διάταξη. Έγινε κάποιο λάθος στα δικά μου έγγραφα. Είναι παρόν ο κύριος Κάρλος Σίλβα. με χαρά σας δίνω το λόγο. Παρακαλώ. Καλημέρα σας. Θα σας διαβάσω την αναφορά μου. Τα ε, ισπανικά ή ε, καστελιάνο, καστελικά είναι η ε, ε, επίσημη γλώσσα της ε, Ισπανίας και το άρθρο 3 του συντάγματος τα ορίζει. 16% του πληθυσμού ζουν στην Καταλωνία ε, και οι περισσότεροι είναι ισπανόφωνοι και το 50% ε, μιλάει ισπανικά και καταλανικά μόνο 36%. Τα τελευταία 40 χρόνια είχαμε κυβερνήσεις τοπικιστικές, εθνικιστικές που χρησιμοποίησαν ως ιδεολογικό όπλο τη γλώσσα για να προωθήσουν μια επιθετική πολιτική ε, επιβολής των καταλανικών παρόλο ε, ή μάλλον ε, με την ε, δικαιολογία ότι ήταν μειονοτική γλώσσα. Αυτό λοιπόν είναι μια κοινωνική μηχανική που έχει επιβάλει ως αιχμή του του στη γλώσσα στα σχολεία, στη δημόσια διοίκηση και από το 1998 αφορά και τις αρχές του ιδιωτικού δικαίου στις εταιρείες και στα καταστήματα. Το 98 είναι ο νόμος που ορίζει ότι πινακίδες και γενική ενημέρωση και ε, τα φυλάδια, τα εμπορικά ε, και διαφημίσεις για τους καταναλωτές και τις εγκαταστάσεις που είναι ανοιχτές στο κοινό θα πρέπει να ε, έχουν συνταχθεί τουλάχιστον στα καταλανικά. Και ο νόμος του 2010 για την κατανάλωση όριζε λεπτομερώς για τους καταναλωτές το δικαίωμα να έχουν τα έγγραφα για τα συμβόλαια στα καταλανικά και διάφορα άλλα εμπορικά, καθώς επίσης και τις απαραίτητες πληροφορίες για την κατανάλωση, τη χρήση και τη διαχείριση ε, εμπορευμάτων και υπηρεσιών. Δεν ισχύει κάτι αντίστοιχο για τους Ισπανόφωνους, άρα έχουμε αποκλειστική χρήση στο εμπόριο της καταλανικής γλώσσας. Δύο μέτρα και δύο σταθμά. Προστατεύονται οι καταναλωτές και στον αντίστοιχο κώδικο της ε, κατανάλωσης με αντίστοιχε ποινέ και κυρώσει για όσους παραβιάζουν την νομοθεσία στα καταλανικά και των καταλανοφών. Στι αρχές του 2010 ο συνήγορος του πολίτη ε, προσέφυγε στο συνταγματικό δικαστήριο μετά από ε, την ε, πρόταση της οργάνωσης Impulsos Ciudadano. 4 Ιουλίου 2017. Απόφαση. Θεωρεί το δικαστήριο ότι θα πρέπει ως εξής να ερμηνεύεται ο νόμος στα ισπανικά θα πρέπει να γίνεται η πληροφορία γιατί αυτή είναι η κοινή και επίσημη γλώσσα σε όλη την Ισπανία. Στα θέματα της κατανάλωσης η αυτόνομη περιφέρεια ε, έχει αρμοδιότητες ε, να προβεί σε ε, διαφορετικές ρυθμίσεις για την προστασία των πολιτών και των καταναλωτών. Δηλαδή μπορεί να προωθούν τη γλώσσα την καταλανική αλλά δεν σημαίνει ότι αυτό θα είναι εις βάρος των Ισπανών και Ευρωπαίων πολιτών που έχουν δικαίωμα να ενημερώνονται στα Ισπανικά. Η ε, ε, υπηρεσία κατανάλωσης ε, χρησιμοποιεί μόνο καταλανικά αρκεί να το δει κανείς στην ιστοσελίδα της. Από το 1998 θέλουν να επιβάλλουν στο εμπόριο την τοπική γλώσσα και χιλιάδες Μεγάλες και μικρές επιχειρήσεις έχουν υποστεί δρακόντιους ελέγχους και κυρώσεις για τις πινακίδες που δεν είχαν στα καταλανικά ή στις διαφημίσεις. Ε, ε, ε, οι επιθεωρητές κατανάλωσης έχουν γίνει θεματοφύλακες της καταλανικής γλώσσας χωρίς να ελέγχουν αν υπάρχει στα ισπανικά η αντίστοιχη ενημέρωση που είναι επίσημη γλώσσα τα ισπανικά της Ένωσης και γλώσσα που καταλαβαίνουν όλοι οι Ισπανοί πολίτες. Διακρίσεις αυτό. Άρα ενημέρωση δεν θέλουν να είναι στα ισπανικά ε, στη διάθεση των καταναλωτών και των πολιτών. Αυτή η εθνικιστική πολιτική ήταν πάρα πολύ αποτελεσματική. Στη Χερόνα, στη Λέιδα και στην Ταραγώνα ε, είναι αποκλειστική κατά πλειονότητα ε, η αναγραφή στα καταλανικά και στην Βαρκελόνη 15,8% και 31,3% μόνο στα ισπανικά. Τα καταλανικά που υποτίθεται ότι είναι γλώσσα μειονότητας έχει κυριαρχήσει ε, στις πινακίδες, στη γραπτή ενημέρωση και στην πληροφόρηση των εμπορικών καταστημάτων. Άρα έχει κάνει μειονοτική τη γλώσσα του κράτου στην επίσημη, τα ισπανικά. Ε, τέλος, το δικαίωμα που αναγνωρίζει για τους πολίτες ε, και τους ε, καταναλωτέ η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είναι εγγυημένη. Με απόφαση των αρμοδίων αρχών της Καταλωνία που υποτίθεται ε, ότι ε, τους ενδιαφέρει ε, η ενημέρωση των Ισπανών πολιτών. Στο άρθρο 38 του Χάρτη Μιλιοδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης ορίζεται ότι οι πολιτικές της Ένωσης θα πρέπει να εγγυώνται υψηλή προστασία των καταναλωτών. Οι διακριτικές πρακτικές της διοίκησης της Καταλωνίας όχι απλώς ε, παραβιάζει το άρθρο 21 του λόγου χάρτη που αναγνωρίζει τη μη διάκριση με βάση τη γλώσσα αλλά και στην ε, ποικιλομορφία Τη Ένωση, τη γλωσσική και αρνούνται την προστασία σε όλου του καταναλωτέ, Για να υπάρχει υψηλή προστασία του καταναλωτού είναι εκ των όνου κάνευ να έχει πρόσβαση ο καταναλωτή σε μια γλώσσα που καταλαβαίνει για να διαφυλάξει τα συμφέροντά του με βάση τα άρθρα που αναφέραμε και το άρθρο 4 παράγραφος 2 ε, ψηφίο F 12, 114 και 116 της ΛΕ συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης ζητούμε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να ελέγξει τη γλωσσική πολιτική της κυβέρνησης Καταλωνίας γιατί δεν εγγυάται τα δικαιώματα και την πληροφόρηση των καταναλωτών στα ισπανικά, τη γλώσσα που καταλαβαίνουν. Να ε, ε, μεταβεί εκεί αντιπροσωπεία που να ε, εξετάσει την κατάσταση επιτόπου και να ληφθούν τα απαραίτητα μέτρα για να αυτή η γλωσσική πολιτική που είναι αντίθετη με την Ευρώπη των πολιτών διότι παραβιάζει τα δικαιώματα ενημέρωσης των καταναλωτών στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ταυτόχρονα ζητούμε να παραμείνει ανοιχτή η ε, αναφορά μέχρι να αρθεί αυτή η παράβαση και η παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των Ισπανοφόνων στην Καταλωνία. Ευχαριστώ πολύ και τώρα θα δώσουμε το λόγο στην πρόσωπο ε, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Κριστέλ Μάρκετ Επικέρας. Σας ευχαριστώ Πρόεδρε, ευχαριστώ για την αναφορά. Έχει σαν στόχο ο το μιλητής τον σεβασμό των πολιτιστικών και γλωσσικών δικαιωμάτων των πολιτών που περιλαμβάνεται και στο άρθρο 3 της Συνθήκης και στο άρθρο 21 της Χάρτας για τα θεμελιώδη δικαιώματα. Σύμφωνα με την Συνθήκη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν έχει αρμοδιότητα παρέμβαση στα κράτη-μέλη σε σχέση με τα θεμελιώδη δικαιώματα. Μπορεί να το κάνει όταν τίθεται θέμα μη σεβασμού ε, ευρωπαϊκής νομικής ρύθμισης. Η χάρτα εφαρμόζεται από τα κράτη-μέλη ε, όταν εφαρμόζουν τον Ευρωπαϊκό Νόμο, την Ευρωπαϊκή Ρύθμιση. Η χρήση των περιφερειακών και εθνικών γλωσσών είναι αποκλειστική αρμεδιότητα των κρατών μελών που έχουν την πλήρη εξουσία να ρυθμίζουν αυτή την ε, λειτουργία σύμφωνα με τον καταστατικό τους χάρτη σχετικά με την χρήση των περιφερειακών γλωσσών, την αναγνώριση γλωσσικών δικαιωμάτων σε συγκεκριμένα εδάφη. Η εφαρμογή των γλωσσικών καθεστώτων ανήκει στις αρμοδιότητες είτε των περιφερειακών αρχών είτε του εθνικού επίπεδου. Γι' αυτό θα πρέπει τα κράτη-μέλη να χρησιμοποιήσουν όλα τα μέσα που έχουν στην διάθεσή τους έτσι ώστε τα θεμελιώδη δικαιώματα όπως προβλέπονται και καταγράφονται από τις εθνικές ρυθμίσεις και τις διεθνείς συμφωνίες να γίνονται σεβαστά. Εμείς δεν μπορούμε να δώσουμε συνέχεια εδώ γιατί η τα γλωσσικά δικαιώματα είναι αποκλειστικά εθνική αρμοδιότητα. Καλώς. Θα δώσουμε τώρα το λόγο στα μέλη της Επιτροπής η Μάιτε, παρακαλώ, Ευχαριστώ πολύ. Πρώτα απ' όλα θα ήθελα να σας ευχαριστήσω που ήρθατε εδώ να μας ε, μιλήσετε ε, για μια κατάσταση η οποία ε, αποτελεί σαφή διάκριση και οπωσδήποτε θα πρέπει να αποφεύγεται και να αποφευχθεί ε, στην ε, προκείμενη περίπτωση. Ναι, βεβαίω, εδώ υπάρχει απλωστική αρμοδιότητα ε, του κράτου μέλους και επομένως αυτό το κράτος μέλος θα πρέπει να δει με ποιο τρόπο θα αντιμετωπίσει αυτήν τη μορφή διακριτικής μεταχείρισης που τόσο ορθά και συγκεκριμένα μας αναφέρατε. Προσωπικά, εγώ να πω ότι εμένα δεν μ' αρέσουν οι ιερεοεξεταστές ε, της γλώσσας ε, και που μας λένε ε, πώς πρέπει να μιλάμε και τι πρέπει να κάνουμε και να ελέγχουν πώς μιλάμε και πιστεύω ότι με τον τρόπο αυτό πραγματικά παραβιάζονται τα δικαιώματα των πολιτών. Και δεν είναι αυτό που επιθυμούμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευχαριστώ Μάιτε, λέει η Πρόεδρος. Θα δώσουμε το λόγο Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θέλω να ευχαριστήσω πολύ την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Εδώ βλέπουμε ότι πρόκειται για διάκριση και παραβίαση των θεμελιωδών αρχών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το διαπιστώνει αυτό η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αλλά όπως λέει και ο χάρτης θεμελιωδών δικαιωμάτων, αυτό είναι στην επικουρικότητα και δεν μπορεί να επέμβει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή βάσει του άρθρου 51 που το βρίσκουμε απέναντι μας τόσες φορές εδώ στην Επιτροπή μας. Θεωρείται Ευρωπαϊκή Νομοθεσία ο χάρτης γιατί υπάρχει ένα άρθρο το 51 ε, το οποίο επιτέχει ερμηνείες. Ξέρουμε ότι προσπαθούμε να το λύσουμε αυτό το πρόβλημα με όλες τις δυνάμεις μας. Θα ήθελα όμως να θυμίσω ε, στην Επιτροπή και να τη ζητήσω και θα το ζητήσω και στην Επιτροπή μας. Γιατί ζητάει ο αναφερόμενο να γίνουν σεβαστά και να προστατεύονται τα δικαιώματα των καταναλωτών. Βεβαίως υπάρχει θέμα διάκρισης, αλλά εδώ ε, πρόκειται για τους καταναλωτές, τους Ευρωπαίους και τους Ισπανούς, αλλά και τους Ευρωπαίους, γιατί πολλοί Ευρωπαίοι ζουν στην Ισπανία, μη Ισπανοί, να έχουν πρόσβαση στην ενημέρωση στη γλώσσα που καταλαβαίνουν. Αυτό είναι ευρωπαϊκή νομοθεσία. Στο άρθρο 38 αναφέρεται η προστασία των καταναλωτών, όπω γνωρίζετε. Και πέρα από τις διακριτικές πρακτικές θα ήθελα να τονίσω το εξής. Η εσωτερική αγορά είναι εμβληματική μας ε, πολιτική και θέλουμε η ευρωπαϊκή ηθαγένεια, η ιδιότητα του Ευρωπαίου πολίτη να συνάδει με τη συμβίωσή μα σε ένα ενιαίο χώρο. Οι γλώσσε είναι εργαλεία και μπορεί να υπάρχουν ε, εθνικές νομοθεσίες, γιατί το ορίζουν οι συνθήκες, αλλά για να υπάρχει εσωτερική ενιαία αγορά και οι Ευρωπαίοι πολίτες να μπορούν να απολαμβάνουν απολύτως αυτές τις δυνατότητες, θα πρέπει να προστατεύσουμε τα δικαιώματα των καταναλωτών. Και υπό την έννοια αυτή ζητώ από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να ε, έχουν λόγο και επιτροπές Γιούρι και ΙΜΚΟ ε, και να παραμείνει ανοιχτή αναφορά γιατί θεωρώ ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να προσπαθήσει να μελετήσει σε βάθος αυτή τη γλωσσική πολιτική της κυβέρνησης Καταλωνίας γιατί δεν εγγυάται στους καταναλωτές αυτό το δικαίωμα να ε, έχουν ενημέρωση στη γλώσσα που καταλαβαίνουν. Ε, απευθυνθείτε στην κυβέρνηση της Καταλωνίας και να ρωτήσετε ποια είναι η πολιτική της η γλωσσική στο συγκεκριμένο θέμα. Ευχαριστώ. Thank you very much and, and... Ευχαριστώ πολύ. Και θέλω να σας ευχαριστήσω όλους σας για την υπομονή σας. Χρειάστηκε να βγω και ευχαριστώ τη Ρόζα που προείδρευσε για λίγο. Η Τερέσα Χιμένεθ. Ευχαριστώ πολύ. πολύ ενδιαφέρον αυτό που κάνουμε εδώ, γιατί νομίζω ότι είμαι η μόνη Καταλανή που έχω μητρική γλώσσα τα καταλανικά και που δεν είμαι εθνικίστρια και που δεν συμφωνώ με πρακτικές τις οποίες η κυβέρνηση της Καταλωνίας, η Generalidad, έχει κάνει ε, ε, παραβιάζοντας δικαιώματα καταναλωτών ε, γιατί θεωρούν ότι μια τέτοια γλωσσική στρατηγική όπως λένε οι ίδιοι μπορεί να αποτελέσει οικοδόμηση εθνικής στρατηγικής. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι έχουν μαγαζιά, κάνουν εμπόριο που υποφέρουν από τέτοιες ε, ε, καταστάσεις που αφορούν την γλώσσα. Είναι γεγονός επίσης ότι υπάρχει το άρθρο 51 ε, αλλά υπάρχουν και άλλα στοιχεία τα οποία μας οδηγούν στην έννοια της παραβίασης των δικαιωμάτων των καταναλωτών. Εγώ, καταναλωτών. Εγώ θα ήθελα να σταλεί στην κούλτ τη Ζούρη και την, την Γιούρη και την Ίνκο έτσι ώστε αυτή η αναφορά έτσι ώστε να μπορέσει να λυθεί το πρόβλημα γιατί είναι σοβαρό. Και εδώ στο Κοινοβούλιο πρέπει να βρούμε τρόπο έτσι ώστε να βρεθεί κάποια λύση. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Η Σολεδάδ Καμπεθών. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Πρώτα απ' όλα να σας πω ότι αισθάνομαι θλίψη. Γιατί Ε, έχουμε κάποιες αναφορές με το θέμα αυτό. Και μετά έχουμε και το θέμα της εκπαίδευσης μετά από το ΕΛΚ. Και τα δύο θέματα έχουν πρόσφατη απόφαση του συνταγματικού δικαστηρίου και στις δύο υποθέσεις. Η καταλανική κοινωνία αυτή την περίοδο αντιμετωπίζει μια δύσκολη κατάσταση. Είναι μοιρασμένη η κοινωνία και δεν είναι η κατάλληλη στιγμή έτσι ώστε αυτή ακριβώς τη στιγμή και αυτή την περίοδο να κάνουμε και μια τέτοια συζήτηση. Η Ισπανία είναι πολύμορφη, ε, από την Ανδαλουσία μέχρι την Καταλωνία έχει μεγάλο πολιτιστικό πλούτο και ε, θα πρέπει οι πολιτικές οι οποίες εφαρμόζονται να χρησιμοποιούν, να αναδεικνύουν τον πλούτο αυτό και να μην φέρνουν σε αντίθεση τον ένα πολιτισμό με τον άλλον. Θα πρέπει να ληφθούν τα μέτρα τα οποία θα βοηθήσουν την ειρηνική συμβίωση η οποία τόσο έχει υποφέρει το τελευταίο διάστημα. Το 2010 ε, υπήρχε απόφαση Ε, απόφαση του συνδεγματικού δικαστηρίου ε, μετά από μήνυση 50 βουλευτών του ΕΛΚ. Ε, και εν πάση περιπτώσει εδώ μιλάμε για επίσημα στοιχεία ε, ε, που λένε ότι, και νόμους που λένε ότι δεν μπορεί στον, στον ιδιωτικό τομέα ε, να υποχρεωθεί κάποιος να χρησιμοποιήσει τη μία ή την άλλη γλώσσα. Απλώς θα πρέπει να είναι σαφής ο νόμος ότι θα πρέπει ο καταναλωτής να έχει την δυνατότητα να ψωνίσει, να κάνει τη δραστηριότητά του στη γλώσσα την οποία κατανοεί. Θα πρέπει να λυθούν τα προβλήματα αυτά Ειρήνη, δεν ε, είναι δυνατόν να υπάρξει επιβολή στην μία ή στην άλλη περίπτωση. Και βεβαίως ε, υπάρχει η δυνατότητα όπως έκανε άλλωστε και η κυβέρνηση της Καταλωνίας να εφαρμόσει ε, κάποια πρόστιμα ή κάποιες ε, κυρώσεις σε περίπτωση που παραβιάζεται ο νόμος που έχει δικαίωμα να εφαρμόσει. Εν πάση περιπτώσει το θέμα είναι, αποτελεί εθνική αρμοδιότητα. Εγώ αυτό δεν το αμφισβητώ. Αυτό που λέω είναι ότι θα πρέπει με ηρεμία να αντιμετωπίσουμε τα θέματα αυτά. Πριν από μερικούς μήνες κάναμε μια συζήτηση ε, στα πλαίσια της Επιτροπής μας μετά από αναφορές που προέρχονται από την ε, Καταλωνία. Ε, και εμείς είπαμε ότι δεν είναι δυνατόν να κάνουμε τέτοιες συζητήσεις οι οποίες καθόλου δεν βοηθούν τη συνύπαρξη. Δεν είναι ο κατάλληλος χρόνος, δεν είναι σκόπιμο να συζητηθούν αυτά τα θέματα τώρα. Αυτή τη στιγμή στην Καταλωνία και στην Ισπανία διεξάγονται πολύ ευαίσθητες συζητήσεις. Η περίοδος είναι ευαίσθητη και επομένως το πρόβλημα θα πρέπει να λυθεί στην Ισπανία και δεν πρέπει το ΕΛΚ, ε, το, Ευρωπαϊκό, συγγνώμη, το Λαϊκό Κόμμα της Ισπανίας να προσπαθεί ε, να κρυφτεί πίσω από τέτοιου είδους ε, αναφορές έτσι ώστε να κερδίσει. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ Σολεδάτ και σε ευχαριστώ πολύ που τόνισε στο στοιχείο της συμβίωσης και της συμφιλίωσης ή δυνατόν και τις ενιαίες δράσεις ε, τονίζοντας και τις εθνικές αρμοδιότητες ε, στο θέμα αυτό. Κύριε Στερικά Μπράς. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κοιτάξτε, εγώ δεν είδα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να υποστηρίζει την αναφορά. Εγώ άκουσα την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να λέει ότι δεν είναι δική της αρμοδιότητα. Δηλαδή να έρθουν όσες φορές θέλετε, αλλά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πάντα αναρμόδικα ε, θα δηλώνει. Ευχαριστώ τη Σολεδάδ Καμπεθόν Ρουίθ για τα όσα είπε. Γιατί καταδεικνύει κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Μπορεί να έχουμε διαφορετικές ιδεολογικές θέσεις, αλλά αυτό δεν θα πρέπει να γίνει ιδεολογικό το πρόβλημα, όπως επιδιώκουν ορισμένες πολιτικές ομάδες. Είναι ένα θέμα γλωσσικό, συμβίωσης και ζήτημα των πολιτών. να έρθουν στις πόλεις μας και στη Βαρκελόνη όσοι δεν έχουν πάει εκεί και θα διαπιστώσουν ότι δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Και ρωτώ, επιβλήθη καμία κύρωση σε κάποιον που χρησιμοποιεί μόνο ισπανικά στις πινακίδες, όχι. Τώρα γίνεται λόγος για αποκλεισμό των Ισπανικών για επιθετική πολιτική Μα για όνομα του Θεού, ξέρετε ότι οι δικαστέ στην Καταλωνία δεν είναι υποχρεωμένοι να γνωρίζουν καταλανικά και να μπορούν να δικάζουν στα ισπανικά. Μιλάμε για άκαμπτη αστυνομική πολιτική. Μα τι είναι αυτά. Υπερβολικά πράγματα. Αυτά είναι μια, ε, παραμύθια για να τρομάζουν τα μωρά. Εγώ ερωτώ. Δεν υπάρχει γλωσσικό πρόβλημα διότι ο νόμος ορίζει τάδε τάδε και και το λένε και τα δικαστήρια να αναγράφεται τουλάχιστον στα καταλανικά για να ε, ε, προάγονται τα καταλανικά, αλλά δεν λέει αποκλειστικά στα καταλανικά, λέει τουλάχιστον στα καταλανικά να αναγράφονται κάποια ε, στοιχεία στις διαφημίσεις και τις πινακίδες. Και όσο και αν συμπαθώ τη φίλη μου, για τους ξένους που ζουν στη Βαρκελόνη, στην Καταλωνία. Θα πρέπει να ενημερώνονται σε μια γλώσσα που να καταλαβαίνουν, που είναι τα ισπανικά. Αυτό σε αντίληψη μου φαίνεται υπερβολικό. αυτή είναι η γλώσσα που κατανοούν τα ισπανικά οι ξένοι στην Ισπανία. Μα τι μυστήρια πράγματα είναι αυτά. Πρέπει να σας πω ειλικρινά και το λέω και με αγάπη και με προσοχή και ό,τι θέλετε. Μου φαίνεται ανόητο όλα αυτά και τελείως ανυπόστατα. Αυτή η νόμη είναι προστατευτική για την κατάσταση στην ε, Καταλωνία και μιλάτε τώρα για δικαστήρια εμείς ξέρουμε ότι οι πολίτες εκεί είναι δίγλωση. Δεν υπάρχει πρόβλημα κανένα στη χρήση των γλωσσών, ούτε διάκριση καμία, ούτε πολιτική, ούτε επιθετική πολιτική, ούτε τίποτα από όλα αυτά. Αν θέλετε να το ε, διαπιστώσετε η σώμαση ελάτε. Ε, εγώ νομίζω ότι πρέπει να κλείσει αυτή η αναφορά, διότι δεν έχει καμία προοπτική πορεία, ας πούμε. Θέλετε να την αφήσουμε ανοιχτή, θα συζητάμε τα ίδια και τα ίδια αιώνε ολόκληρες επειδή είναι ανυπόστατη, δεν θα έχει και μέλλον. Ευχαριστώ. Thank you very much. And I see that colleagues Ευχαριστώ πολύ. Βλέπω ότι υπάρχουν συνάδελφοι που ζητούν το λόγο για δεύτερη φορά, αλλά δεν μπορώ να σας το δώσω, γιατί ε, θα προχωρήσουμε στην επόμενη. Ε, η Ρόζα όμως, στην επόμενη. Η Ρόζα ζήτησε το λόγο για πρώτη φορά. Ρόζα. Εγώ είμαι δίγλωση. Μιλώ και καταλανικά και ισπανικά. Ε, αφού είμαι από τη Μαγιόρκα και έχω να σας πω το εξής στις αυτόνομες ε, περιφέρειες στις ε, Βαλεαρίδες στην Καταλωνία παντού έχουμε πραγματικά την ευκαιρία να έχουμε δύο γλώσσες και η κυβέρνηση πρέπει να προστατεύει και τους δύο είναι γεγονός ότι στις στις έχουμε τα καταλανικά των νήσων στην υπόλοιπη Καταλωνία έχουμε τα καταλανικά ε, και είναι ε, γεγονός ότι τα παιδιά από πολύ μικρή ηλικία ξέρουν και τις δύο γλώσσες. Η αρμονική συμβίωση μεταξύ των δύο γλωσσών μας έχουν οδηγήσει εδώ, σε αυτό που εμείς ονομάζουμε ε, στον εγκάρδιο, σεβαστικό και συμβιωτικό δίγλωσο πολιτισμό. Εμείς δεν έχουμε κανένα πρόβλημα ε, να διδασκόμαστε και να διδάσκουμε στις δύο γλώσσες. Αυτό που δεν μας... Ε, αυτό που ε, με φέρνει κάπως σε αντίθεση με τον φίλο που μίλησε προηγουμένως ε, είναι ότι ε, υπάρχουν αυτοί οι ε, πολίτες οι οποίοι είναι υπέρ της ανεξαρτησίας και οι οποίοι πιστεύουν ότι μπορούν να χρησιμοποιήσουν σαν όπλο ανεξαρτησίας αυτό το, αυτή την γλώσσα. Η γλώσσα μου, τα καταλανικά, την, την αγαπώ και τη χρησιμοποιώ, αλλά διαφοροποιούμε όταν χρησιμοποιείται σαν όπλο. Ε, και όταν μιλάμε για υποχρεώσεις ε, τότε πραγματικά ε, δεν υπάρχει πια η, αυτή η, εγκάρδια συμβίωση, ο η εγκάρδια διγλωσία. όταν σε μια επιγραφή ή σε ένα σχολείο είναι υποχρεωτική η μόνη αναφορά της καταλανικής γλώσσας, τότε πραγματικά δεν υπάρχει η εγκάρδια συμβίωση και, αυτή η εγκάρδια σωστή διγλωσία η οποία πρέπει να χρησιμοποιείται και στον ιδιωτικό και στο δημόσιο τομέα, σε δημόσιες υπηρεσίες κλπ. Ωστόσο, είναι αλήθεια ότι δεν ξέρω πώς να σας μεταφέρω αυτή την έννοια ε, στην οποία αναφερόταν και η Μάιτε και η Μπεατρίθε σχετικά με την συμβίωση, όχι την αντιπαράθεση των δύο γλωσσών, αλλά την δυνατότητα της ένταξης, ε, της ε, σύμπτυξης των δύο γλωσσών. Ε, ισορροπία λοιπόν βάσει της κοινή λογικής αυτό που ζητούμε και αυτό που ζητούν οι αναφερόμενοι είναι η κοινή λογική, είναι αυτή η αρμονία. Ε, βεβαίως η Κομισιόν μπορεί να πει ότι ε, δεν έχει ε, αρμοδιότητα αλλά Ζουζέπ και στην Δονιάνα είπε ότι δεν έχει αρμοδιότητα και σε ένα σωρό άλλα πράγματα είπε ότι δεν έχει αρμοδιότητα ενώ εμείς ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι οι πολίτες καίγονται από τα ζητήματα αυτά. Ε, Ωστόσο, είναι ε, γεγονός ότι ε, όταν αρχίζει μία κυβέρνηση να τρελαίνεται και να λέει ότι 100% ε, αποκλειστική χρήση μονάχα της μίας γλώσσας, αυτό αρχίζει και είναι επικίνδυνο. Πιστεύω λοιπόν ότι μέσα από την αγάπη της χώρας μας, από την αγάπη της γης μας, από την αγάπη της καταλανικής γλώσσας να προχωρήσουμε. Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, στην παρούσα φάση θα ήθελα να δώσω το λόγο στον αναφερόμενο για μια πάρα πολύ μικρή παρέμβαση. Ακούσατε τις παρεμβάσεις, δεν ξέρω αν θέλετε να αντιδράσετε. Καταρχάς να εκφράσω αυτά τα οποία είπε η σοσιαλίστρια Ευρωβουλευτής ε, στην ουσία σε σχέση με την σιωπή η οποία θα πρέπει να επικρατήσει και θα αμφισβητήσω επίσης αυτό το οποίο είπε ο κύριος Κάμπρας ότι δεν είναι ιδεολογικό, μα είναι ιδεολογικό. Πρόκειται για ένα σχέδιο εθνικής οικοδόμησης ε, και με βάση κανονικά τις αρχές με τις οποίες θα συμφωνούσαμε την προάσπιση των μειονοτικών γλωσσών. Βλέπουμε τις Βρυξέλλες ότι υπάρχει μια μεγάλη πλειοψηφία γαλλόφωνων στις Βρυξέλλες και οι ταμπέλες υπάρχουν και ε, ε, ταμπέλες, ε, όχι όμως μόνο στα φλαμανδικά, ενώ αυτό σημαίνει στην Καταλωνία. Οι εθνικιστικές αρχές στην Καταλωνία χρησιμοποιούν με στρεβλά μέσα τις αρχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω μιας προσπάθειας δημιουργίας τελεσμένων και απομόνωσης του, της, των Ισπανικών, των επίσημων Ισπανικών. Δεν μπορούμε εμείς να το αποσιωπήσουμε αυτό και να πω επίσης προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να εξετάσει το θέμα αυτό και να εξετάσει την κατάσταση την οποία βιώνουμε στην Καταλωνία. Καλώς σας ευχαριστώ πολύ για την παρέμβασή σας ένα μόνο άκουσα να ζητά να κλείσει η αναφορά και θα πρέπει να ε, πράγματι ισχύει αυτό. Θέλετε να κλείσει κύριε Τέρη Κάμπρας. Όχι, ναι ή όχι. Ναι, κάποιος θέλει να κλείσει, αλλά η πλειοψηφία θέλει να παραμείνει ανοιχτή, θα την κρατήσουμε ανοιχτή να δούμε αν υπάρχουν νέα επιχειρήματα, δεν ξέρω ποια θα μπορούσαν να είναι, δεν το φαντάζομαι, αλλά δεν μπορώ να κλείσω την αναφορά εφόσον οι συνάδελφοι διαφωνούν. Σας ευχαριστώ, περνάμε στο επόμενο θέμα, στο οποίο αναφέρθηκα προηγουμένως, στην 857 για την ε, καταλανόφωνη εκπαίδευση αποκλειστικά στις οικογένειες οι οποίες μετακομίζουν στην περιοχή αυτή. Καλημέρα σας. Έχω κάποιες διαφάνειες. Λέγομαι ένα Ρωσάδα και απευθύνομαι σε εσά ως πρόεδρος ενός δίκλου σχολείου και μητέρα δεκάχρονου παιδιού. Εγώ είμαι Καταλανή αλλά Ισπανόφωνη και εκπροσωπώ μία οργάνωση που υπερασπίζεται τα δικαιώματα πολλών γονέων που ανησυχούν από τις επιπτώσεις ε, που έχει η εκπαίδευση των παιδιών μας, περιθεροποιείται η γλώσσα μας στην Καταλωνία, ιδιαίτερα ε, για τα πιο ε, ευαίσθητα και ευάλωτα παιδιά. Οι μισοί Καταλανοί είμαστε Ισπανόφωνοι. μας, η γλώσσα μας είναι και αυτή η επίσημη γλώσσα στην αυτόνομη περιφέρεια της Καταλωνίας και η κοινή γλώσσα που στην υπόλοιπη Ισπανία. Το Υπουργείο Παιδείας της Καταλωνίας δεν σέβεται τα γλωσσικά δικαιώματα των Ισπανόφωνων μαθητών. Το ο εκπαιδευτικό πρότυπο στην Καταλωνία επιβάλλει την καταλανική γλώσσα ως βασική γλώσσα της εκπαίδευσης. Τα παιδιά μας δεν μπορούν να μάθουν να διαβάζουν και να γράφουν στη γλώσσα τους. Στην ηλικία των τριών ετών θα πρέπει να αρχίσουν να ξεχνάνε τις πρώτες λέξεις που συζητούν, που χρησιμοποιούν στο σπίτι τους, με τις οικογένειές τους και οι γονείς θα πρέπει να υπογράψουν ότι συμφωνούν με την ε, γλωσσική πολιτική του σχολείου για να γράψουν τα παιδιά τους στο σχολείο. Τα καταλανικά είναι η μόνη γλώσσα ε, που διδάσκεται και χρησιμοποιείται στις δραστηριότητε, εσωτερικές και εξωτερικές του σχολείου. Κοιτάξτε παρακαλώ αυτή τη διαφάνεια ε, με προσοχή. Στα περισσότερα σχολεία έχουν από μηδέν ε, ώρες ισπανικά την εβδομάδα ε, στον υπηαγωγείο, δύο στο δηματικό και τρεις στο, στην δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Άρα, στα παιδιά μας με τρόπο άμεσο ή έμεσο ε, τους μαθαίνουν ότι δεν είναι γλώσσα πολιτισμού τα ισπανικά. Δεν τα χρησιμοποιούν για να τους διδάξουν μαθηματικά ιστορία ή επιστήμες. Ούτε τραγουδούν τα κάλαντα, ας πούμε, ε, τα Χριστούγεννα, ούτε στο θέατρο, ε, ούτε μιλούν με τους ε, καθηγητές ισπανικά, ούτε τα μαθήματά τους κάνουν στα ισπανικά. Αυτό είναι πάρα πολύ μεγάλο τίμημα για τους ισπανόφωνους μαθητές που αποτεχάνουν και καταλείπουν το σχολείο και ε, εγκαταλείπουν πολύ περισσότεροι ισπανόφωνοι από ότι καταλανόφωνοι μάθητες στο σχολείο. Τώρα βλέπετε ε, τι λέει η UNESCO για την ε, κατάληψη του σχολείου. Μέχρι 10% πιο υψηλή είναι αυτή η κατάσταση στους Ισπανόφωνους. Και με μαύρο βλέπετε τι γίνεται στη χώρα κατά μέσο όρο και στα παιδιά που δεν έχουν ως μητρική τη γλώσσα που χρησιμοποιείται στο σχολείο. Και ε, όσοι είναι καταλανόφωνοι και βγαίνουν στο σχολείο στη μετρική τους γλώσσα, ε, δεν έχουν τόσο μεγάλα προβλήματα. Τα, τα ισπανόφωνα παιδιά ε, θεωρούν ότι είναι λιγότερο ενταγμένα στο σχολείο από ότι σε άλλε αυτόνομε περιφέρειες τη Ισπανία. Εδώ έχουμε δύο ομάδε που πλήττονται ιδιαίτερα. Τα παιδιά με ιδιαίτερε ε, ανάγκε, με αναπηρίε, που είναι ισπανόφωνα δηλαδή έχουν κάποιο πρόβλημα στην ακοή, στην όραση, η σωματική αναπηρία ή διαταραχές στην επικοινωνία. Αφήστε που έχουν ε, δυσκολίες ε, ε, Μαθησιακέ στο σχολείο λόγω τη αναπηρία έχουν κι άλλο εμπόδιο. Ε, ούτε σε αυτά τα παιδιά δεν του επιτρέπουν ένα τμήμα των μαθημάτων να τα κάνουν στα ισπανικά. Υποχρεωτικά μόνο στα καταλανικά όλα τα μαθήματα. Ούτε καν ε, στην ειδική στήριξη, στην ε, ενισχυτική διδασκαλία που δικαιούνται το φροντιστήριο δεν μπορούν να το κάνουν στα ισπανικά. Και κάθε χρόνο μετά το πίσω ότι μετακινούνται χιλιάδε ε, πολίτες προς την Καταλωνία είτε από την Ισπανία είτε από αλλού από την Ευρώπη όταν... και έχουν παιδιά που θέλουν να γράψουν στο σχολείο. Και πάνε να τα γράψουν στο σχολείο και δεν βρίσκουν ε, ότι να υπάρχουν δημόσια σχολεία που να γίνεται με το μάθημα στα ισπανικά. Και ρωτάνε πώς θα συνεχίσουν τις ε, σπουδές τους αργότερα και τους ε, ενημερώνουμε ότι πρώτα τους διαχωρίζουν από τους υπόλοιπους μαθητές και πάνε να τους μάθουν καταλανικά. Και όλα τα μαθήματα θα τα κάνουν στα καταλανικά και δεν μπορούν να του εξετάσουν γιατί δεν του αφήνουν να απαντήσουν στα ισπανικά. Και πολλοί γονεί δεν δέχονται μια θέση εργασία στην Καταλωνία και όσοι έρχονται κινδυνεύουν να δουν τα παιδιά του να μένουν στην ίδια τάξη ή να παίρνουν χειρότερου βαθμού. Το άρθρο 14 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης αναγνωρίζει το δικαίωμα στην παιδεία και στην εκπαίδευση. Λογικά το δικαίωμα αυτό θα πρέπει να γίνεται αδιακρίτω γλώσσα και να ε, γίνεται σεβαστή πάντα η διαφοροποίηση των γλωσσών και η ποικιλομορφία. Ε, στην Καταλωνία αυτό δεν γίνεται για τους Ισπανόφωνους μαθητές. Αυτό στρέφεται κατά των συστάσεων και των νόμων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει αρμοδιότητες για να συντονίζει, να βοηθάει να συμπληρώνει τη δράση των κρατών μελών ε, στα θέματα της εκπαίδευσης. Κυρίες και κύριοι βουλευτές, σήμερα έχω έρθει για να σας ζητήσω να ελέγξετε ε, κατά πόσο αυτά που ισχυριζόμαστε εδώ είναι αλήθεια. Η γλωσσική πολιτική στην εκπαίδευση στην Καταλωνία ε, σημαίνει διάκριση εις βάρος των ισπανόφωνων μαθητών. Ε, επαρεμποδίζει την ατομική του ανάπτυξη, την κινητικότητα και δυσκολεύει την ένταξη των παιδιών με αναπηρίε. Γι' αυτό τι ζητάμε. Πρώτον, από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να ε, εξετάσει και να διερευνήσει τις καταχρήσεις εις βάρος των παιδιών που όλες αναφέραμε. Δεύτερον, ζητούμε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να τα καταδικάσει αυτά και να στείλει επιστολή στην τοπική κυβέρνηση, στη Βουλή της Καταλωνίας και στην Ισπανική κυβέρνηση, εκφράζοντας την ανησυχία της και απαιτώντα την άμεση λύση τη ε, κατάσταση αυτή τη διάκριση. Και τρίτον, ζητούμε να παραμείνει ανοιχτή αυτή η αναφορά μέχρι να μάθουμε ότι έγιναν οι συγκεκριμένε δράσει και αποκαταστάσει αποκαταστάθηκαν τα θεμελιώδη δικαιώματα που αυτή τη στιγμή παραβιάζονται και τα δικά μας και των παιδιών μας. Ευχαριστώ. Thank very much. Σας ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα τώρα να στραφώ στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ο κύριος Μάρκ έχει το λόγο. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Η αναφορά αυτή αναφέρεται στην υποχρεωτική εκπαίδευση ε, στα σχολεία της Καταλωνίας, ιδιαίτερα για οικογένειες που μετακινούνται από άλλες περιοχές ε, στην Καταλωνία. Είναι αποκλειστική αρμοδιότητα των κρατών μελών. Είναι θέματα που άπτονται της εκπαιδευτικής πολιτικής και τα κράτη-μέλη είναι υπεύθυνα για την διδασκαλία και την κατάρτιση των προγραμμάτων. Θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση να σέβεται την πολιτιστική ποικιλία των κρατών μελών και γι' αυτό η επιλογή της γλώσσας εκπαίδευσης ή οποιοδήποτε άλλου θέματος σχετικά με την χρήση των γλωσσών στην εκπαίδευση είναι αποκλειστική αρμοδιότητα ε, των κρατών μελών τα θέματα αυτά δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και πρέπει να αντιμετωπιστούν σε επίπεδο εθνικό. Και ε, ε, όπως είπα προηγουμένως, το θέμα της Χάρτας των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων εφαρμόζεται για τα κράτη-μέλη μόνο σε σχέση με τις πιθανές παραβιάσεις του ευρωπαϊκού δικαίου. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Θα ξεκινήσουμε τη συζήτηση με τα μέλη. Μπεατρίς, ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Ε, καταλαβαίνω ότι δυσκολεύεστε να κατανοήσετε και να αποδεχτείτε ότι συμβαίνει αυτό. Ότι στην Καταλωνία αυτοί που μιλούν ε, ισπανικά υφίστανται διακρίσεις. ακόμα και αν προσπαθούμε εδώ στο Κοινοβούλιο να πούμε ότι όλα είναι καλά, ε, δεν είναι έτσι. Δηλαδή δεν προστατεύονται αποτελεσματικά τα δικαιώματα των παιδιών στην εκπαίδευση. Και επίσης ε, υπάρχουν και στοιχεία του νόμου, των νομοθετημάτων ευρωπαϊκών, τα οποία παραβιάζονται σε σχέση και με το άνθρωπο, που ανέφερα και προηγουμένως τη ε, χάρτα Θεμελιωδών Δικαιωμάτων. Ε, εγώ όμω εδώ μιλάμε, ε, δεν συμφωνώ ότι μιλάμε για την εκπαιδευτική πολιτική μιλάμε για, την, για τα δικαιώματα των παιδιών, των ανηλίκων, μιλάμε για εγχειρηματοποίηση των παιδιών. Και εδώ μιλάμε επίσης για πολιτικές ε, τις οποίες, ε, οι οποίες είναι ελλειπτικές όσον αφορά ε, τα όσα κάνει η καταναλική κυβέρνηση. Και γι' αυτό οι πολίτες στρέφονται προς την Ευρωπαϊκή Ένωση προσπαθώντας να βρουν άκρη, προσπαθώντας να βρουν το δίκαιο τους. Γιατί αν και εμείς πούμε αποστρέφουμε το βλέμμα και δεν μας ενδιαφέρει, τι θα κάνουν τότε προς τα που θα στραφούν εδώ εμείς είμαστε το παράθυρο ευκαιρίας για 500 εκατομμύρια πολίτες που αισθάνονται ότι παραβιάζουν τα δικαιώματά τους ε, και νομίζω ότι θα πρέπει οπωσδήποτε ε, όπως ζήτησε και η αναφερομένη ε, να στείλουμε μια επιστολή και στα ανώτερα δικαστήρια Κόρτες χενεράλες αλλά και στην τοπική κυβέρνηση της También συγγνώμη, και στην Βουλή, καθώς επίσης και στην κυβέρνηση της Καταλωνίας, έτσι ώστε να παραμείνει ανοιχτή η αναφορά και να γνωστοποιήσουμε και σε εκείνους τον προβληματισμό μας. Και να δούμε εάν πραγματικά υπάρχουν αυτά ή αν είναι, όπως ακούστηκε προηγουμένως, φανταστικές ιστορίες και βεβαίως να παραμείνει ανοιχτή. Well, Καλώς. Θα επανέλθουμε. Η Γιούρη τι σχέση έχει τώρα με αυτό το θέμα, αλλά θα δούμε με άλλες επιτροπές που θα μπορούσαν να ε, εμπλακούν. Θα ήθελα τώρα να δώσω το λόγο στη Μάιτε Παπασορτούντουα. Muchas, muchas gracias, Presidenta. Σας ευχαριστώ, Πρόεδρε. Νομίζω ότι θα πρέπει να στηρίξουμε την αναφορά. Εγώ είμαι καθηγήτρια φιλόλογος ε, και στην Βασκική και στην Ισπανική και γνωρίζω το θέμα των γλωσσών και τις διδασκαλίες τους στην γλώσσα στη χώρα μου και έχω εργαστεί στην εκπαίδευση για πολλά χρόνια στην αυτονομή περιοχή από την οποία προέρχομαι Υπάρχουν πολλοί τρόποι διάσωσης και προώθησης του γλωσσικού μας πλούτου. Μιλάμε για πολύ μεγάλες ε, ομάδες ε, ε, μαθητών και αν υπάρχουν ειδικέ ανάγκες και το επιθυμούν οι γονείς μπορούν να κάνουν εγγραφή στη μητρική τους γλώσσα. Είναι θεμελιώδες δικαίωμα των ίδιων των παιδιών και όταν κάποιες διοικήσεις αναλαμβάνουν την εξουσία και το εμποδίζουν αυτό είναι απαράδεκτο. Εγώ είμαι φυσικά υπέρ της πολυγλωσσίας. Υπάρχουν ε, πολλοί τρόποι προώθησης της πολυγλωσσίας. Αλλά δεν μπορούμε να θεωρούμε τα παιδιά κατώτερα της γλώσσας όταν φυσιάζουμε τις ειδικέ ανάγκες ορισμένων παιδιών και των οικογενειών τους και επιβάλλουμε ένα και μόνο αποκλειστικά ένα πρότυπο εκπαίδευσης και γλωσσικό. Στην ουσία εδώ υφίστανται δίωξη οι πολίτες, υπάρχει ένα πρόβλημα που δεν είναι μόνο εκπαιδευτικό. Στο παρελθόν έχουν υπάρξει προβλήματα από άλλου είδους φυσικά μορφές εξουσίας, αλλά είναι απαράδεκτο να μην υπάρχουν τάξεις με διδασκαλία της ισπανικής. Η γλώσσα, η γλώσσα του πολιτισμού είναι κάτι το οποίο γίνεται αντικείμενο δουλειάς ε, και στα σχολεία και δεν πρέπει να επικρατεί αυτή η διγλωσία σήμερα. Δεν μπορούν οι διοικητικές αρχές να αρνούνται το δικαίωμα στα παιδιά στην διγλωσία αυτή. Νομίζω λοιπόν ότι όχι μόνο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να ασχοληθούν με το θέμα γιατί μιλάμε για τα παιδιά. Τα παιδιά είναι πιο σημαντικά από τις εκπαιδευτικές πολιτικές και πιο σημαντικά από τις κυβερνήσεις και τα συμφέροντά τους. να προσθέσω κάτι σε αυτά που είπαμε προηγουμένως. Όταν μια κυβέρνηση σε μια περιοχή είναι δίγλωση, συμβαίνουν αυτά γιατί στην εκκίνηση της γλωσσικής διδασκαλίας σημαίνει ότι δίδεται προτεραιότητα σε μία γλώσσα και αυτό σημαίνει ότι φύγονται τα δικαιώματα των πολιτών. Εγώ ήμουνα για 10 χρόνια αντιπρόεδρος της κυβέρνησης ε, της Περιφερειακής των Βαλεαρίδων Νήσων Είχαμε πάρει πολλές αποφάσεις γύρω από τα θέματα τα γλωσσικά. Στις περιφέρειες αυτές το ιδανικό είναι να είμαστε ευέλικτοι, να χρησιμοποιούμε το θέμα των γλωσσικό, ιδιαίτερα για τα παιδιά με ειδικέ ανάγκες και εγώ έχω ένα παιδί με τέτοιες ειδικέ ανάγκες, τα παιδιά που δεν ακούν καλά, τα παιδιά που έχουν προβλήματα γενικότερα, να προσαρμόζεται το σύστημα, να καλύπτει τις ανάγκες αυτές να προσαρμόζεται στις ανάγκες του παιδιού, διότι ακριβώς τα παιδιά είναι ο στόχος ακριβώς της ε, παιδείας. Θα πρέπει λοιπόν το σύστημα να είναι ανοιχτό σε όλες τις γλώσσες με ευελιξία, να μαθαίνουν και τις δύο γλώσσες, γιατί εμείς ε, που είμαστε από τις ε, περιοχές αυτές λατρεύουμε την τοπική μας γλώσσα. Εγώ λατρεύω την καταλανική αλλά θέλω όμως να μην επιβάλλονται οι εκπαιδευτικές διαδικασίες με τέτοιο τρόπο. Όταν επιβάλλονται τέτοιες αποφάσεις οδηγούν σε διαιρέσεις και σε διαφωνίες. Αυτό θα πρέπει να το λάβει υπόψη η Επιτροπή. Γιατί υπάρχουν ορισμένα κόμματα τα οποία έχουν αιμονή με το θέμα της εθνικής γλώσσας. Μα τι είναι η γλώσσα είναι ένα μέσο επικοινωνίας, επαφής και όχι ένα όπλο επιθετικότητας. Λοιπόν, κάτι λέει ο κύριος Κάμπρας, αλλά εκτός μικροφώνου. Εγώ θέλω να ακολουθήσουμε έναν κοινό δρόμο. Δεν ε, θα ήθελα να πω στις Βαλεαρίδες υπάρχει ένα μια κυβέρνηση 7 κομμάτων και υποχρεώνει τους ιατρούς όταν θέλουν να ασκήσουν το δικαίωμά τους να είναι υποχρεωμένοι να ομιλήσουν την καταλανική ε, για να μπέξει κανείς στην συμφωνική ορχήστρα πρέπει να ξέρει την καταλανική λοιπόν τώρα αυτά όταν φτάνουμε σε τέτοια κατάσταση δεν έχει πια νόημα. Αυτό το οποίο ζητούν λοιπόν οι αναφερόμενοι και αυτό το οποίο ζητώ εγώ είναι η κοινή λογική. Να μην επιβάλλουμε τέτοιου είδους καταστάσεις. Μια γλώσσα την αγαπάει κανείς με την καρδιά και όχι με την επιβολή εκ των άνω και έτσι θα μάθουμε δύο, τρεις και τέσσερις ε, ε, ε, γλώσσες. Θα πρέπει λοιπόν να ακολουθήσουμε ένα κοινό δρόμο, ευελιξία, καρδιά και κοινή λογική. Εδώ νομίζω ότι δεν θα πρέπει να παίρνουμε μέτρα για να διαιρέσουμε την κοινωνία. Νομίζω ότι ε, μια κυβέρνηση δεν μπορεί να επιβάλλει διαιρώντας, θα πρέπει να επιβάλλει ίσως αποφάσεις οι οποίες να ενώνουν, να στραφούμε στο μέλλον λοιπόν με δύο γλώσσες σε κοινή πορεία και με τη μέγιστη δυνατή ευελιξία. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Λόπεθ Αγγελάρ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Η πρόεδρος Βίξτρομ της Επιτροπής μας γνωρίζει ότι δεν είμαι πλήρες ε, μέλος εδώ. Αλλά προσπαθώ να έρχομαι όταν έχουμε θέματα που αφορούν την εκλογική μας περιφέρεια, δηλαδή το κράτος μέλος μας. Οι Ισπανοί βουλευτές και το συγκεκριμένο θέμα είναι τέτοιο. Πάντα έρχομαι με σεβασμό και με τιμή για τα μελήματα των αναφερμένων που είναι συμπολίτε μας, όχι απλώς Ευρωπαίοι, αλλά και Ισπανοί. Ξέρει, Πρόεδρο ότι εδώ και χρόνια ασχολούμαι με τα θεμελιώδη δικαιώματα και τι ελευθερίε, Γιατί ε, είναι κοινέ πολλές οι προσπάθειές μας στην Επιτροπή ΛΥΜΠΕ. Συμμετέχουμε εκεί με την Πρόεδρο Βίξτον και με άλλα μέλη της Επιτροπής ε, Αναφορών στην Επιτροπή Ελευθεριών. Και αυτό το θέμα άπτεται των θεμελιωδών δικαιωμάτων ανηλίκων δια του εκπαιδευτικού συστήματος. Επιπλέον είμαι άκρευτνής υποστηρικτής της συνταγματικής ποιότητας της Ισπανίας ως κράτους μέλους. Δυστυχώς χρειάστηκε πάρα πολλές φορές τα τελευταία χρόνια να την περασπιστώ απέναντι σε εκείνους που προσπαθούν να μειώσουν ή να υποτιμήσουν την σημασία της συνταγματικής τάξης στην Ισπανία, που είναι κράτος με σύνταγμα. Υπάρχει ένα άρθρο στο Ισπανικό Σύνταγμα, το άρθρο 3, που είναι πάρα πολύ δύσκολο να μεταρρυθμιστεί, που θεωρεί και καθιερώνει ως επίσημη γλώσσα του κράτους τα Ισπανικά. Υπάρχουν και άλλες γλώσσες ε, στο Ισπανικό κράτος, που επίσης προστατεύονται ε, χαιρετίζονται μάλιστα στο προήμιο του συντάγματος και έχουν επίσημο χαρακτήρα στις λόγω αυτόνομες περιφέρειες και ορίζεται έτσι από το ίδιο το καταστατικό του το σύνταγμα το τοπικό. Έτσι κι αλλιώ είναι τεράστια η πολιτιστική κληρονομιά στην Ισπανία και αξίζει και υποστήριξη και προστασία και σεβασμό. Οι αυτόνομες λοιπόν περιφέρειες που έχουν μία συνεπίσημη γλώσσα ανέπτυξαν και σωστά ε, γλωσσικές πολιτικές. Ε, στην περίπτωση της αυτόνομης περιφέρειας της Καταλωνίας η γλωσσική αυτή πολιτική επικυρώθηκε με διαδοχικές αποφάσεις του Συνταγματικού Δικαστηρίου από την αρχή της δεκαετίας του 80. Και παρόλα αυτά υπάρχουν προβλήματα. Προβλήματα που αφορούν τα δικαιώματα των πολιτών και ιδιαίτερα ευάλωτων προσώπων όπως είναι εξορισμού οι νέοι και τα παιδιά μας στο εκπαιδευτικό μας σύστημα. Και αυτά τα προβλήματα χρειάζονται προσοχή ε, και λύση ε, και υπάρχουν συστήματα προσφυγής για προστασία. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναφέρθηκε στις αρμοδιότητες των κρατών μελών. Μάλιστα. Έρχονται εδώ οι αναφερόμενοι με λόγο διαρθρωμένο. Ε, θα πρέπει να δώσουμε συνέχεια ε, εμείς ε, στην Επιτροπή μας και να παραμείνει ανοιχτή αυτή η αναφορά. Ευχαριστώ. Τερέσα. Η Τερέσα Χιμένεθ. Ευχαριστώ πολύ. γιατί έτσι αναπτέρωσε στο ηθικό μου μετά από την ε, θλίψη που μου προκάλεσε η παρέμβαση της ε, συναδέλφου σου. Ε, εδώ μιλάμε για τα θύματα της πολιτικής της Καταλωνίας. Εγώ επαναλαμβάνω, είμαι Καταλανή. Εγώ μιλάω με τα παιδιά μου και με τα εγγόνια μου με, στα καταλανικά. Ε, εγώ επέλεξα καταλανικό σχολείο για το παιδί μου γιατί θέλω να ξέρουν να μιλάνε καλά καταλανικά. Εγώ υποστήριξα το δίγλωσσο σύστημα της Καταλωνίας και τα τελευταία χρόνια όμως ε, η κατάχρηση ήταν τόσο μεγάλη που πλέον συνειδητοποίησα ότι δεν πρόκειται για εθνικιστές ε, που θέλουν να προστατεύσουν τη γλώσσα τους αλλά πρόκειται για ανθρώπους που προσπαθούν να χρησιμοποιήσουν τη γλώσσα όπως λένε γίνει σαν ένα εργαλείο εθνικής οικοδόμησης ε, και πλέον ε, εγώ σχεδόν αισθάνομαι να, να απεχθάνομαι τη γλώσσα. Μια αποστροφή αισθάνομαι πια ε, σχεδόν για τα καταλανικά. Αυτό συμβαίνει στην Καταλωνία. Μαζί με κάποια άλλα πράγματα τα οποία και οι άνθρωποι μεγάλοι ή και τα παιδιά κατανοούν αυτή την διάχυτη ισπανοφοβία που προκύπτει και από τον τρόπο με τον οποίο τα ισπανικά ε, ε, αντιμετωπίζονται στα καταλανικά σχολεία. Αυτό είναι το πρόβλημα ε, είναι ότι χωριζόμαστε δύο, σε δύο κοινότητες και ενώ εμείς πρέπει να ξαναενωθούμε και όπως είπαν προηγουμένως οι συνάδελφοι να υπάρχει ανεκτικότητα ναι αλλά και πλήρης σεβασμός του νόμου. Δεν υπάρχει, ε, ίσως εκτός από τη Ιρλανδία, άλλη ε, χώρα όπου να μην μπορεί κανείς να μάθει και να εκπαιδευτεί στην επίσημη γλώσσα της χώρας του, ενώ ζει μέσα στη χώρα του. Αυτά. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ, ο κύριος Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Τι να πω τώρα. Δεν έχω λόγια. Να λέτε ότι δεν μπορεί κανείς να μάθει Ισπανικά στην Καταλωνία, τι δεν το χωράει το μυαλό μου. Με κάθε σεβασμό για όποιον έχει διαφορετική άποψη, αλλά πραγματικά έχω μείνει ευρώντιτος με αυτά που ακούω. Δογματικός δεν είμαι και μπορώ να επικρίνω και την κυβέρνηση της Καταλωνίας και όποιον άλλον θέλω. Και τον εαυτό μου τον ίδιο. Δεν έχω κανένα πρόβλημα. Και καλό θα ήταν να κάνουμε καμιά φορά την αυτοκριτική μας. Όχι, ε, μπορείτε να με επικρίνετε. Λοιπόν, θα ήθελα να μιλήσω για κάτι πραγματικό, αν υπήρχε αυτό. Αλλά και πάλι σε αυτή την αναφορά, τη 19 και την 20, Είναι διαδοχική η κατάθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Τι σύμπτωση είναι αυτή, τυχαίο, δεν νομίζω. Είναι μια συντονισμένη επιχείρηση αυτή. Και πάλι πρόκειται για έναν ύπαρκτο πρόβλημα. Μας έδωσε κάποιες στατιστικές η αναφορά που δεν αντιστοιχούν στα στοιχεία που έχω εγώ. Και θα πρέπει να τα δούμε αυτά κατά αντιπαράσταση. Και ποιο είναι το πρόβλημα. Παιδαγωγικό είναι ή μήπως άλλου τύπου. Γιατί είναι παιδαγωγικό και αυτό είναι το ενδιαφέρον στο σχολείο, η μηπω αλλου τυπου γιατι ειναι παιδαγωγικο και αυτο ειναι το ενδιαφερον στο σχολειο η παιδαγωγικη Στην Καταλωνία έχουμε 300 γλώσσες. 3-0-0 γλώσσες. Τι έγινε, θα δώσουμε τώρα σε όλα τα παιδιά τη δυνατότητα να διαβάζουν, να γράφουν στη γλώσσα τους. Ναι, να είμαστε συνεπείς λεκτός μικροφώνου η Μάιτε. Ναι, ναι, πολύ ωραία αυτά που λέτε. Αλλά εγώ ξέρω ποιο είναι το πρόβλημα. Τι θα κάνουμε τώρα. Υποθέτω ότι θα πρέπει να διευκολύνουμε ε, όλα τα παιδιά. Δεν υπάρχουν μια-δυο γλώσσε όπω είναι τα καταλανικά και τα ισπανικά που να βοηθήσουν τα παιδιά να αναπτυχθούν. Για να είναι τα παιδιά από τη Ζιμπάμπου, Ζιμπάμπου ή η ίδια χώρα ή ε, ε, από πουθενά αλλού. Es lo que te acabo de decir, que me parece que no me escuchas. Μα αυτό προσπαθώ να πω, Ρώσα, δεν με ακούς κιόλα. Η Μπεατρίτ. Τώρα λέει ότι οι γονείς πρέπει τίποτα, για μια στιγμή. Δεν πρέπει τίποτα να κάνουν οι γονείς. Ε, το κάνουν οι γονείς. Για ποιο λόγο. Εσείς μπορείτε να το παρουσιάζετε έτσι, αλλά ορισμένοι γονείς είστε που δεν εκπροσωπείτε σε καμία περίπτωση την πλειονότητα των γονέων στην Καταλωνία. Σε καμία περίπτωση. Και θυμίζω σε όλους ότι η ένταξη η σχολική ένταξη ήταν κάτι που προωθήθηκε βασικά από Ισπανόφωνους γονείς στην Σάντα Κολόμα de και για όσοι δεν γνωρίζουν αυτό το χωριό είναι πάρα πολύ Ισπανόφωνο ή Καστιγιανόφωνο εν πάση περιπτώσει και αυτοί το αποφάσισαν για ποιο λόγο γιατί θέλουν τα παιδιά τους να έχουν ίσες ευκαιρίες και με όλα τα υπόλοιπα παιδιά ε, στην Καταλωνία άρα είναι κοινωνικό εγχείρημα πάρα πολύ ενδιαφέρον και δεν μου άρεσε. Τώρα έχει φύγει η κυρία ε, Ρώσα Εσταράς και δεν με ε, βολεύει καθόλου αυτό. Γιατί αυτό που είπε για την επιβολή της γλώσσας, αυτό το ψήφισε το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα. Το Λαϊκό Κόμμα της Ισπανίας, μάλλον. Που κυμαίνεται τις απόψεις. Και πολύ θα ήθελα να μου πει μια μέρα τι γίνεται με τους νομικούς που υπάρχουν μόνο γερμανόφωνοι στη, στην Πάλμα τη Μαγιόρκα. Μα το πρόβλημα είναι οι Καταλανοί, οι άλλες εθνικότητες εντάξει. Και πολλές διεθνείς οργανώσεις ε, έχουν ε, εκφράσει την ικανοποίησή τους για αυτά και η Ευρωπαϊκή Ένωση κτλ. Όλες αυτές οι αιτιάσεις δεν έχουν αποδειχθεί. Υπάρχει εγκατάλειψη του σχολείου. Όχι. Α, τα άκουσες. Εδώ ήσουν. Ε, αυτά με τους Γερμανούς. Ωραία. Ευχαριστώ. Υπάρχει έκθεση πίζα που λέει ότι τα παιδιά μας ξέρουν καλύτερα ισπανικά από το μέσο όρο των Ισπανόφωνων ή των παιδιών στην Ισπανία. Οπότε δεν θα τα κάνουμε όλα και τόσο στραβά μάλλον. Ε, ζητώ να κλείσει αυτή η αναφορά και να μην αποστείλουμε καμιά επιστολή για τη διάκριση. Γιατί αν τη στείλουμε σημαίνει ότι συμφωνούμε με τη διάκριση. Αυτό δεν έχει ακόμα αποδειχθεί. Αν ισχυριζόμαστε ότι υπάρχει η διάκριση, είμαστε χαμένοι. Και τι λόγο έχει ύπαρξη τότε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και εμεί οι ίδιοι. Να κλείσει αναφορά. Γιατί εδώ μυρικάζουμε ξανά και ξανά όλα αυτά τα πράγματα χωρίς αξιόπιστα στοιχεία και χωρίς να υπάρχει λίμα στο σχολείο στην Καταλωνία. Θεέ μου, Θεέ μου. For me. Ωραία, εγώ που είμαι Σουηδέζα, ναι. ε, είναι πάρα πολύ δύσκολο να, έτσι, να αντιμετωπίσω μια τέτοια επιτροπή γεμάτη Ισπανούς που μιλάνε με ένταση, με ζέση, με πάθος. Λοιπόν, θα, ξανα, θα δώσω το ρόλο στο Σολιδάδη και μετά ξανά στην αναφερόμενη. Πολύ ε, γρήγορα. Νομίζω ότι όλοι εξέθεσαν ε, τα ε, επιχειρήματά τους. 28 Φεβρουαρίου του 2018 ε, η Καταλωνία έχει την καλύτερη επίδοση στην γνώση της Ισπανικής ε, σε σχέση με όλες τις άλλες δίγλωσες ε, αυτόνομες κοινότητες. εντάξει, μπορούμε να πούμε πολλά, αλλά υπάρχουν κάποια στοιχεία τα οποία δείχνουν ότι γνωρίζουν Ισπανικά και μελετούν Ισπανικά τα παιδιά στην Καταλωνία. Ε, είναι γεγονός ε, ότι εδώ μιλάμε για μια περιοχή ιδιαίτερα πλούσια, ε, πλούσια πολιτιστικά και η γλώσσα αποτελεί ένα στοιχείο πλούτου και γι' αυτό λέω ότι θα πρέπει και το ξαναλέω θα πρέπει να αποφύγουμε οπωσδήποτε οποιαδήποτε διάκριση αλλά να μην, δεν είναι δυνατόν να εφαρμόσουμε να μην μάθουν, να μην μαθαίνουν τα παιδιά αυτά και καταλανικά και να μαθαίνουν μόνο ισπανικά. Έχουν δικαίωμα τα παιδιά αυτά να μαθαίνουν καταλανικά. Ε, κοιτάξτε, υπάρχουν και αποφάσεις του συνταγματικού ε, δικαστηρίου όσον αφορά και το θέμα αυτό. Μπορεί να θέλετε να το ξεχάσετε, αλλά οι αποφάσεις είναι εκεί. Ε, και, εν πάση περιπτώσει, εκεί αναφέρονται απλώς ότι κάποια πράγματα είναι δυνατά δυνάμει και του, των σχετικών άρθρων του καταστατικού της καταλανικής κυβέρνησης. Ε, ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι και η Θιουδαδάνος και το Λαϊκό Κόμμα της Ισπανίας ε, έχουν βασίσει πολιτικές τους ε, εκστρατείες πάνω σε τέτοια τόσο ευαίσθητα θέματα. Τι να σας πω. Ήδη τα πράγματα είναι δύσκολα, η κατάσταση είναι δύσκολη στην ε, Ισπανία για να χρησιμοποιούνται αυτά τα θέματα ε, ψηφοθυρικά για να κερδίσει κανείς ε, λίγες ψήφους. Καλώς. Θα ήθελα να καταλάβω τώρα πόσο μεγάλη είναι η διαφορά. Υποθέτω ότι η διαφορά είναι ανάμεσα όπως ας πούμε νορβηγικά και σουηδικά ε, καταναλβαίνει ο ένας τον άλλο. Γιατί να δημιουργούνται τέτοιου είδους διαφορές όταν καταλαβαίνουν οι μεν τους δε. Θα ήθελα να μου εξηγήσετε τις μεγάλες διαφορές ανάμεσα στην Ισπανική και την Καταλανική. Θα δώσω το λόγο στην κυρία Λοσάδα. Ευχαριστώ. Θα ήθελα να απαντήσω στις τελευταίες παρεμβάσεις. Να πω στην ε, εκπρόσωπο της σοσιαλιστικής ομάδας να κάνω μια διόρθωση γιατί είπε ότι κάτι ζήτησα το οποίο δεν το είπα. Εγώ δεν ζήτησα να γίνονται οι σπουδές μόνο στην ε, ε, Ισπανική. Εμείς είμαστε Καταλανοί δίγλωση Θέλουμε λοιπόν να γίνονται σεβαστά τα δικαιώματα των ομιλητών της, και της καταλανικής και της ισπανικής, όλων των καταλανών δηλαδή και των δύο γλωσσών. Η συμβίωση βασίζεται στον σεβασμό και των δύο. Αν ε, ένα σχολείο περιθωροποιεί τη μία γλώσσα, ε, ε, επιβάλλει τη μία γλώσσα εις βάρος της άλλης θα ήθελαμε τα παιδιά μας να μπορούν να σπουδάζουν και στις δύο γλώσσες, να διδάσκονται και οι δύο γλώσσες γιατί είναι χρήσιμο για τα παιδιά όταν ενηλικιωθούν. Ε, αυτό το ότι θέλουμε εμείς να επιβάλλουμε τα ισπανικά επειδή υποτίθεται είναι ανώτερα, αυτό είναι επιχείρημα των εθνικιστών. Υπάρχουν ε, εξετάσεις πάρα πολύ δύσκολες. Λοιπόν, το θέμα είναι με ποιο τρόπο προωθούνται οι δύο γλώσσες, οι δύο διαφορετικές γλώσσες. Όπως είμαι μητέρα λοιπόν, είμαι πολίτης που δεν ανήκω σε κανένα ακόμα και θα ήθελα να πω ότι η κόρη μου μπόρεσε να επικοινωνήσει με τα παιδιά τα οποία μιλούσαν την καταλανική αλλά φοβάμαι ότι αναγκάζομαι να επικοινωνώ, είπε το παιδί. Καταλάν, Ή και castellano es para hablar en casa. Yo lo que quiero συναντηθήκαμε στο δρόμο με μια φίλη μου και τη μίλησα καταλανικά ε, και η, η, μικρή μου κόρη των τεσσάρων ετών μου είπε «Μαμά, γιατί μιλά τη γλώσσα του σχολείου και όχι τη γλώσσα που μιλάμε εμεί στο σπίτι». Ε, το θέμα είναι λοιπόν να μην φέρουμε τη μία γλώσσα απέναντι στην άλλη και να έχουμε όλοι ίσα δικαιώματα. Ευχαριστώ πολύ να συνοψίσω, να συνοψίσω αυτό το πολύ δύσκολο θέμα. Νομίζω όμως ότι μπορούμε να προχωρήσουμε ήρεμα και ωραία. Να τα ξαναδούμε λοιπόν, να ξαναδούμε πολύ ε, προσεκτικά ε, την κατάσταση. Μπορούμε να αφήσουμε αυτήν την ε, υπόθεση ανοιχτή. Υπάρχει όμως και μία απόφαση η οποία αποφασίζει ότι τα ισπανικά εξίσου με τα καταλανικά πρέπει να χρησιμοποιηθούν. Επίσης το ανώτατο δικαστήριο τον Απρίλιο του 2015 απεφάνθη ότι τα καταλανικά σχολεία οφείλουν να παρέχουν 25% των μαθημάτων στα στα ισπανικά, να διδάσκουν στα ισπανικά. Σύμφωνα με αυτά που μας δείξατε όμως, τα μικρά παιδιά έχουν μηδέν ώρες ισπανικής διδασκαλίας. Ε, ε, αυτό λοιπόν είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να το καταδείξουμε, γιατί μια απόφαση δικαστηρίου είναι μια απόφαση δικαστηρίου. Μπορεί κανείς ε, να δείχνει τα συναισθήματά του με όποιο τρόπο θέλει, αλλά οπωσδήποτε πρέπει να ε, ακολουθείτε και να γίνεται σεβαστή μια απόφαση δικαστηρίου. Θα πρέπει λοιπόν επίσης να πούμε ότι η Ευρώπη ε, θέλει να διευκολύνει την ελεύθερη κυκλοφορία όλων. Άρα ε, υπάρχουν οικογένειες οι οποίες θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να πάνε στην Καταλωνία για μικρή χρονική περίοδο και να μην έχουν χάσει εντωμεταξύ από τη διαμονή τους στην Καταλωνία την γνώση της Ισπανικής στα παιδιά τους γιατί αυτό είναι κατά των αξιών αυτής της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Άρα παραμένει ανοιχτή η αναφορά. Στέλνουμε επιστολή στις ε, τοπικές ε, αρχές προς πληροφόρηση αναφερόμενη στις αποφάσεις ε, του δικαστηρίου και αυτά μπορούμε να κάνουμε για την ώρα. Δεν νομίζω ότι μπορούμε να κάνουμε κάτι άλλο. Και φαίνεται ότι συμφωνούν όλοι, Σολεδάδ. Όχι, συμφωνώ, συμφωνώ. Ίσως ενδιαφέρουσα θα ήταν μια επίσκεψη στην ε, ε, Καταλωνία για να δούμε σε τι γλώσσα διδάσκονται και τι γλώσσα μιλάνε τα παιδιά στο σχολείο. Ναι, λέει η Πρόεδρος, αφήνουμε ανοιχτό το θέμα και αν θέλετε αργότερα μπορούμε του χρόνου να κάνουμε με τους συντονιστές μια, να πάρουμε μια απόφαση ε, σχετική με αυτό και αν υπάρχει απόφαση σχετική των συντονιστών να το κάνουμε. Προς όρος όμως κρατάμε την αναφορά αυτή ανοιχτή, ε, παραπέμπουμε ε, μέσω επιστολής στις τοπικές αρχές ε, στην απόφαση του δικαστηρίου. Ευχαριστώ πολύ. λίγη τη συνεδρίασης.